Dear colleagues, I think I will start the meeting. I uh, think we have to gradually try to um, establish a tradition. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσουμε γιατί περνάει η ώρα. We have for our meetings. Uh, so I would like to open the meeting. I would like to welcome all those present. Να μην χάσουμε και τον πολύτιμο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Να ευχαριστήσουμε και όλους τους προσκεκλημένους μας εδώ σήμερα, διότι ε, σήμερα έχουμε ε, διάφορα εργαστήρια για σημαντικά θέματα στην Επιτροπή. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη φυσικά είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Να σας ενημερώσω επίσης ότι ως συνήθως η συνεδρίαση μεταδίδεται μέσω διαδικτύου. Σας διανεμήθηκε η ημερήσια διάταξη την περασμένη Πέμπτη και θα ήθελα να προτείνω μια μικρή αλλαγή επειδή σήμερα είναι και στις 2 η ώρα συνεδρίες των συντονιστών και θα πρέπει να σας ενημερώσω για τις συστάσεις προς την Επιτροπή των Συντονιστών πριν τη σημερινή συν τις συστάσεις που θα προκύψουν και σήμερα, καλό θα ήταν να σας πω τα των συντονιστών μία φορά και να τα πω στις 3 στην ημερήσια διάταξη, το σημείο 3 να πάει δηλαδή από το πρωί στην απογευματινή συνεδρίαση. Αν δεν υπάρχουν ε, ενστάσεις ε, στην ε, μικρή αυτή προσαρμογή της ημερήσιας διάταξης, να σας πω επίσης ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη, ανακοινώση της Προέδρου τρία θέματα. Προϋπολογισμός 2015. Είχαμε δύο σημαντικές τροπολογίες για την πρωτοβουλία για τους Ευρωπαίους πολίτες και οι δύο αυτές υπερψηφίστηκαν στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο. Επομένως θεωρώ ότι αυτά είναι καλά νέα για μας. Και για όσους παρακολουθούν και τις εργασίες της Επιτροπής Προπολογισμών, γνωρίζετε ότι είναι δύσκολη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Από ό,τι φαίνεται το Κοινοβούλιο δεν είναι διατεθειμένο να διαπραγματευτεί το προπολογισμό του 2015 εάν δεν συμφωνηθούν οι αλλαγέ στον προπολογισμό του 2014. Επομένω, ε, θα υπάρξουν αρκετέ δυσκολίε στη διαπραγμάτευση του προπολογισμού. Δεύτερη πληροφορία. η συμμετοχή μου στην ε, συνεδρίαση των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων στη Ρώμη για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Μέχρι τούδε η Επιτροπή μας δεν συμμετείχε, αλλά στα πλαίσια του άρθρου 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου που λέει ότι το, αλφα, ε, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη συνθήκη μέχρι το τέλος του 2017, ζήτησα να υπάρχει και δική μας παρουσία στη διάρκεια αυτών των συνεδριάσεων και ελπίζω να μην ήταν μία εκδήλωση μεμονωμένη, αλλά να υπάρξει και συνέχεια αυτών των συνεδριάσεων και να συμμετέχουμε κι εμείς. Και ε, τρίτη παρατήρηση για την απογευματιμένη μας συνεδρίαση. Είχαμε καλέσει τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Φρανς Τίμερμανς, για να έρθει ε, λίγο τελευταία στιγμή ήταν η πρόσκληση και μάλιστα και πολύ νωρίς ε, το ανέλαβε καθήκοντα η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, και ε, του ζητήσαμε να έρθει για λίγο χρόνο, ε, μπορούμε να του αφιερώσουμε μόνο μια μέρα, αλλά δέχτηκε να έρθει. Και αυτή η δεβιασμένη ίσως πρόσκληση ε, σχετίζεται με το γεγονός ότι η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να είναι ανοιχτές οι συνεδριάσεις με τον ε, πρόεδρο, αντιπρόεδρο επειδή αποφασίστηκε τελευταία στιγμή να είμαστε τρει οι επιτροπέ που ήταν αρμόδιε για τα θέματα του κυρίου Τίμερμαν, η συμμετοχή μα στην επιτροπή ήταν πιο περιορισμένη από όσο θα θέλαμε. Γι' αυτό και τον καλέσαμε για να του αναφέρουμε και ποιε είναι οι προσδοκίε μα. Και τουλάχιστον να έχουμε καλή συμμετοχή των μελών της ομάδος στην απογευματινή συνεδρίαση γιατί έχουμε και μια ευκαιρία να μοιραστούμε λίγο περισσότερα με τον ε, κύριο Τίμερ μας για τις προσδοκίες μας, για το έργο του και επίση να σας ενημερώσω ότι η συνεδρίαση θα είναι πολύ σύντομη, επομένως θα πρέπει να είμαστε πολύ πειθαρχημένοι, μόνο τρία λεπτά για ερωτήσεις και θα ήθελα να ε, γίνει σεβαστός αυτός ο κανόνας και από εσά. Αυτά λοιπόν από πλευράς μου το σημείο 3 λοιπόν ε, ε, μεταφέρεται στο για το απόγευμα και να πάμε τώρα στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Μ' αρέσει όταν μου λένε ότι πρέπει να πω κάτι τώρα, αλλά εγώ δεν θα το πω τώρα. Περνάμε λοιπόν στο εργαστήριό μας, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. είναι πολύ σημαντικό για το έργο μας. Το εργαστήριο αυτό αφορά τις προκλήσεις στον τομέα της αρμοδιότητάς μας για τα επόμενα χρόνια. Όπως γνωρίζετε, οι ευρωεκλογέ μας έχουν δώσει πολλά θέματα να συζητήσουμε όσον αφορά τη δημοκρατική νομιμοποίηση και την ε, νομιμοποίηση της παρούσας ε, θεσμικής ε, διευθέτησης και επομένως ε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα και για μας και πώς οι διοργανικές σχέσεις, οι θέσεις μεταξύ των θεσμών μας οδηγούν στα αποτελέσματα που θέλουμε. Ουσιαστικά λοιπόν με αυτό το εργαστήρι προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με την εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς αυτούς και ε, ευχαριστώ πολύ το Τμήμα Πολιτικής που κατάφερε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να προετοιμάσει αυτό το εργαστήρι. Ελπίζω να γίνει μια πολύ καλή συζήτηση και να μπορέσουμε φυσικά να ε, δημιουργήσουμε και επαφές με τους εμπειρογνώμονες ε, στα πλαίσια των μελλοντικών μας εργασιών. Τέσσερις μεγάλες ενότητες θα συζητήσουμε, το έχετε δει το πρόγραμμα άλλωστε, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες και θα ήθελα να ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Με το πρώτο πάνελ ε, για τις ε, διοργανικές σχέσεις, πρόκειται για ένα πάνελ Ο καθηγητής ε, Μπετοντσίνη θα ξεκινήσει, ο οποίος είναι καθηγητής ε, στο Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ και θα μας κάνει μια παρουσίαση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη νέα πολιτική και θεσμική σύνθεση, καθώς επίσης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Μπερτοντσίνη για να μας πει την άποψή του. Θα ήθελα να σας πω ότι έχετε λιγότερο χρόνο από ό,τι είχε προβλεφθεί και ίσως μπορείτε να περιοριστείτε μια παρέμβαση 15 λεπτών. Α, ίσως μετά να μιλήσω γαλλικά γιατί ε, στα γαλλικά μπορώ να εκφραστώ μεγαλύτερη ακρίβεια ε, και ε, με μεγαλύτερη ταχύτητα. Να σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε, κύριοι Ευρωβουλευτές για την ευκαιρία που μου δίνετε να ανταλλάξω απόψει μαζί σα για τις ε, θεσμικές ε, και πολιτικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτή τη νέα θητεία που μόλι ξεκίνησε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, σας παρουσιάσουμε καταρχάς ένα μικρό έγγραφο εργασία και επίση να γίνεται και αυτή η ανταλλαγή απόψεων επ' αυτή τη βάση για να μπορέσουμε να διορθώσουμε, να συμπληρώσουμε και να τελειοποιήσουμε αυτές ε, τις σκέψεις. Ε, αυτή είναι και η έννοια βέβαια ενό ε, think tank, τουλάχιστον αυτό που διευθύνω εγώ, να συμμετέχουμε σε αυτές τις εργασίες. Θα επικεντρωθώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως μου ζητήσετε, στο νέο πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο Και ξεκινώ από μια διαπίστωση. Το εφαλτήριο είναι... Είναι η συνθήκη της Λισαβόνας. Το πολιτικό πλαίσιο είναι αυτό το οποίο ε, προέκυψε από τις εκλογές, αλλά πέραν αυτού η διαπίστωσή μας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια ενός θεσμικού τριγώνου και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να υπάρχει διπλή εμπιστοσύνη και από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού ε, Συμβουλίου, Συμβουλίου των Κρατών Μελών, έτσι υπάρχει διπλή νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομιμοποίηση για τους πολίτες, νομιμοποίηση για τα κράτη-μέλη η διπλή νομιμοποίηση η οποία φυσικά είναι και εγγεγραμμένη στις συνθήκες. Γι' αυτό λοιπόν και η επιχειρηματολογία μου θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικές προκλήσεις. Καταρχάς τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο τρόπος δηλαδή που δημιουργήθηκε η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεύτερον οι λειτουργίες της και τα καθήκοντά της και τρίτον ε, φυσικά το τι θα μπορέσει να ε, καταφέρει μέσα από τις δράσεις της, πώς ε, θα διεξάγει θα εφαρμόσει τις πολιτικές ε, στα επόμενα πέντε χρόνια. Για τα δύο έχω, πρώτα έχω κάποιες απαντήσεις. Ε, για το τρίτο η συζήτηση είναι ανοιχτή. Ίσως ο αντιπρόεδρος Τίμερμας που θα έρθει το απόγευμα θα μπορέσει να σας πει λίγο περισσότερα. Πρώτον λοιπόν, για να προσπαθήσουμε λίγο να αξιολογήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια αυτού του νέου θεσμικού και πολιτικού πλαισίου ε, και τη σύνθεσή της. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια σύνθεση που αντικατοπτρίζει αρκετά καλά τις πολιτικές ισορροπίες και τις θεσμικές ισορροπίες Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποιες φυσικά αποχρώσεις τις οποίες θα ήθελα να σας παρουσιάσω. Η Επιτροπή Juncker ε, από πλευράς κρατών μελών είναι μία ε, ομάδα 28 εκπροσώπων από τα 28 κράτη-μέλη και με την ισορροπία που εξευρέθη μεταξύ των ε, κρατών μελών. Έχουμε μια σχετικά ικανοποιητική λύση ε, και ουσιαστικά ε, όλα αυτά απορρέουν από άγραφες κανόνες ε, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι από την Ευρωζώνη και από τη Σέγγεν, ο Επίτροπος Οικονομικών Θεμάτων είναι από μια χώρα της Ευρωζώνης. Και πρέπει να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι προέρχομαι και από τη Γαλλία, θα, παρόλα αυτά θα μείνει μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου οι μεγάλες χώρες που παλιά θα θυμάστε ότι είχαν και δύο επιτρόπους αντί για έναν. Για μας ε, παρόλα αυτά θεωρούμε ότι υπάρχουν προβληματικά σημεία όσον αφορά την νομιμοποίηση τους ε, για το σύνολο του, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι και μια επιτροπή στην οποία υπάρχουν επίτροποι ε, από χώρε που δεν συμμετέχουν στην ε, Ευρωζώνη και αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποια ερωτηματικά και αυτοί θα συζητούν οικονομικά ζητήματα. Και η βασική πρόκληση είναι η ε, πολιτική ε, συνάφεια των επιτρόπων. Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ έχει προκύψει από μια καινοτόμο διαδικασία του Spitzenkandidat, του επικεφαλής της λίστας. Ο Επίτροπος Γιούνκερ ανέλαβε, ο πρόεδρος Γιούνκερ ανέλαβε καθήκοντα γιατί ήταν επικεφαλής ε, των κομμάτων που κέρδισαν τις ευρωεκλογέ. Αυτό ε, διευκρίνησε και την συζήτηση πριν από τις εκλογές, όλη την προεκλογική εκστρατεία ε, και είχε μεγάλη βαρύτητα ακριβώς γι' αυτό. Όσον αφορά τη σύνθεση από εκεί και πέρα του υπόλοιπη της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα πράγματα δεν είναι τόσο σαφή. Από ποσοτικής ε, πλευράς, όσον αφορά τις ε, εκλογικές δυνάμεις ε, που προέκυψαν από τις ευρωεκλογές, καθώς επίσης και τις διάφορες πολιτικές συνέφειες που υπάρχουν στο Συμβούλιο Υπουργών, βλέπουμε ότι οι δεξιές κυβερνήσεις είναι λιγότερο επικρατούσε από ό,τι προηγουμένω. Θα σα εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ. Από ποσοτικής πλευράς βλέπουμε ότι 20 στου 28 επιτρόπους ε, ουσιαστικά ανέκουν στο ΕΛ και στου φιλελευθέρου, ε, και υπάρχει και ένας επίτροπος από το ECR και οι οχτώ επίτροποι είναι από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Και αυτό ουσιαστικά δημιουργεί το ίδιο status quo που είχαμε και στην Επιτροπή Μπαρόζο, γιατί εκεί ήταν 21-7 εκεί. Και παρά το γεγονό ότι ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτή τη διαδικασία των Spitzenkandidaten και ε, ε υπήρξε μια προσπάθεια να εξισορροπηθούν τα πράγματα, δεν είναι τόσο εξορροπημένα σε σχέση με το 2009. Επίσης υπάρχει και μια ποιοτική παρατήρηση εδώ να κάνουμε. Ε, υπάρχει ένας αντιπρόεδρος, ο κύριος Τίμερμανς, ο οποίος είναι σοσιαλδημοκράτης που είναι το άλλο ρέγκο του και το δεξί και το αριστερό του χέρι, ε, αυτό λένε και υπάρχουν ε, και τρεις αντιπρόεδροι από το ΕΛ και τρεις σοσιαλιστές, επομένως και εκεί υπάρχει μια ισορροπία και φυσικά οι αντιπρόεδροι έχουν να διαδραματίσουν πιο σημαντικό ρόλο. Από πλευράς όμως ποσότητας, Υπάρχει αυτό το ερωτηματικό, το οποίο φυσικά ε, θα εξαρτηθεί και από το τι θα κάνουν, ε, μπορεί να δημιουργήσει ερωτηματικά για την Επιτροπή Γιούνκερ. Τρίτο στοιχείο, το προσωπικό προφίλ των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει ένα άρθρο της συνθήκης, ε, το 7.3, που ε, λέει ότι οι ευρωβουλευτές ε, επικυρώνουν τις γνώσεις και τις αρμοδιότητες και το κατά πόσον είναι ικανοί είναι επίτροπη. Να σας πω ότι κάποιος ο οποίος θα βλέπει προς τα έξω, από τα έξω, αυτή η μάχη μεταξύ των κομμάτων ε, θεωρήθηκε ως διαστροφή σε σχέση με το άρθρο 17.3 των συνθήκων. Είναι ανησυχητικό ε, να διαβάζει κάποιος ότι ανεξάρτητα από το προφίλ των υποψηφίων ε, ε, επιτρόπων που καλείται να επικυρώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή ανήκουν στο ΤΑΔΕ ή στο ΔΙΝΑ πολιτικό κόμμα, είναι ανέγγιχτοι, δεν μπορεί να τους επηρεάσει κανείς. Και υπήρξε η εικόνα ότι οι ακροάσεις έγιναν με βάση αυτό. Και υπάρχει αυτή η εικόνα δημοσίως ότι ε, βαραίνει ε, η πολιτική τους ε, συνάφεια και όχι το προφίλ του κάθε επιτρόπου. Και έτσι θεώρησαν οι πολίτες ότι έγιναν οι ακροάσεις. Και το θέμα είναι, είναι δυνατόν σε αυτή τη βάση, σε αυτό το πολιτικό ε, και συνταγματικό πλαίσιο να προχωρήσουμε και να πάμε λίγο πιο πέρα ώστε να είναι ακόμα πιο ικανοποιητικά. Εγώ θεωρώ ότι ναι, ε, μπορεί να γίνει αυτό. Μία πρόταση που θα μπορούσε ίσως ε, να συζητηθεί στη συνέχεια είναι αυτό. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει αυξημένη νομιμοποίηση γιατί ήταν ο επικεφαλής της λίστας του κόμματος, επομένως έχει προκύψει από εκλογές έχει και την εξουσία να ανακαλέσει τους επιτρόπους που ανοίγουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους, αλλά δεν έχει δικαίωμα να τους διορίσει. Οι συνθήκες λένε σαφέστατα ότι τα συμβούλια ε, είναι αυτά τα οποία καθορίζουν τους ε, επιτρόπους ε, μαζί με τις κυβερνήσεις οι οποίες έχουν τα ενία. Και επίσης ε, ε, δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο το 17-3 και να, να πάμε λίγο παραπέρα και να πούμε αφού μπορούμε να εκλέξουμε τον πρόεδρο γιατί να μην εκλέγονται και οι επίτροποι. Φυσικά θα γίνεται αυτό σε σχέση με τα κράτη-μέλη, σε σχέση και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά έτσι θα υπάρχει και η πολιτική βαρύτηκα και τα κατάλληλα ε, θεσμικά μέσα ώστε να γνωρίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται οι ισορροπίες ε, μεταξύ των κομμάτων θα ε, του δίνει μια μεγαλύτερη νομιμοποίηση. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω όσον αφορά τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, μια δεύτερη σειρά παρατηρήσεων για τη λειτουργία και τα καθήκοντα της Επιτροπής Juncker, ε, εδώ με τις εξελίξεις οι οποίες είναι σχετικά θετικές και ευνοϊκές. Ξέρετε ότι η μείωση του αριθμού των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε προβλέψει η συνθήκη της Λισαβόνας δεν έγινε. Έχουμε πάντα έναν επίτροπο από ένα κράτος μέλος ε, και αυτό ε, έχει ίσως ε, σημασία ως προς την εκπροσώπηση. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν δεν είχαμε έναν επίτροπο από κάθε χώρα. Είναι και θέμα πολιτικής ευαισθησίας της κάθε χώρας και μπορεί να υπήρχε πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση και θα έπρεπε να οργανωθεί διαφορετικά το, ε, η Επιτροπή και αυτό έκανε ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ άλλαξε λίγο τον τρόπο και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με βάση λοιπόν τη νέα οργάνωση, ο κύριος Γιούγκερ δημιούργησε ένα σύστημα το οποίο είναι λίγο πιο κάθετο. Έχουμε αντιπροέδρους, 7 αντιπροέδρους αντί για 6, αλλά κυρίως αντιπροέδρους οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα σε σχέση με τα μέλη το, της Επιτροπής που έχει ο καθένας στο χρωτοφυλάκιο του. Ε, βέβαια, ακόμα θα πρέπει να αλλάξει λίγο αυτή η δοκιμή, ε, ε, γιατί οι εσωτερικοί κανόνες ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κανονικά δεν το επιτρέπουν. Θα πρέπει λοιπόν να αναδιατυπωθεί ώστε οι αντιπρόεδροι να είναι λίγο πιο ισχυροί σε σχέση με τους υπόλοιπους επιτρόπους και ε, να είναι και υπόλογη ουσιαστικά στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει όμως μια θετική εξέλιξη, την οποία προώθησε ο Ζαν Κλοντ Ιούνκερ, διότι θα είναι λιγότερα τα χαρτοφυλάκια, θα είναι πολύ σαφώς καθορισμένες οι πολιτικές προτεραιότητε, βάσει των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί ε, να κινηθεί συλλογικά. Και υπάρχει και μία ακόμα πρόκληση, ε, αυτό της ομάδος. Το στοιχείο της ομάδος ως προς τα καθήκοντα των επιτρόπων και αυτό είναι ουσιαστικό. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πώς νομιμοποιείται σε σχέση με το Συμβούλιο αφενός ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφετέρου, ε, από το γεγονός ότι έχει 28 επιτρόπους, ο καθένας από ένα κράτος μέλος, ο καθένας με το προσωπικό του προφίλ, που ανταλλάσσουν απόψεις για όλα τα θέματα, όχι ο καθένας για το χαρτοφυλακιό του, αλλά για όλα τα θέματα, ε, κάνουν ανταλλαγές απόψεων σε πολιτικό επίπεδο και ίσως αυτή η ανταλλαγή απόψεων να μεταφραστεί στη συνέχεια ε, και να, σε, υλοποιηθεί μέσω μιας ψηφοφορίας. Και αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει, διότι ο κανόνας είναι απλή πλειοψηφία. Είναι ε, εύκολο λοιπόν να έχουμε τους μισούς επιτρόπους ας πούμε, που να ε, δέχονται, αλλά αυτό σημαίνει ότι ο επικεφαλής της Επιτροπής θα δέχεται αυτή τη συλλογικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να τελειώνει η συζήτηση με μια σαφή ψηφοφορία. Και... Ε, Ακούσατε ότι ο, ο πρόεδρος Γιούγκερ είναι διατεθειμένος να χάσει και κάποια εξουσία ε, λόγω των αντιπρόεδρων. Μπορεί να είναι και διατεθειμένο ε, να χάσει και λίγο ισχύ ακόμα μέσω της ψήφου του. Για να μην είναι ένας ε, πρόεδρος που θα είναι περάν όλων, αλλά να είναι μία ψήφος που θα μετράει, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να αποφασίσει βάσει πολιτικής συζήτησης και όχι απλώς να επικυρώνουν κάποιες τεχνικές αποφάσεις οι οποίες πηγαίνουν προς τη μία στην άλλη κατεύθυνση. Τρίτη, και τελευταία σειρά παρατηρήσεων, ε, ο τρόπος με τον οποίο επ' αυτής της βάσεως μία επιτροπή που είναι, ε, έχει τη συγκεκριμένη σύνθεση και έχει προκύψει με τον τρόπο που προέκυψε μπορεί να υλοποιήσει και να ε, φέρει εις πέρας αποστολές βάσει πρωτοβουλειών και αποφάσεων και αν θα αυξηθεί η νομιμοποίησή της. Εδώ υπάρχουν δύο προκλήσεις κατά την άποψή μου. Υπάρχει μια πρώτη πρόκληση που είναι το στρατηγικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαδικασία του Spitzenkandidat, ε, του επικεφαλής της λίστας, ε, είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία ανάθεσης που στην ε, Γερμανία στη συνέχεια μας οδηγεί στους συνασπισμούς. Υπάρχει και ο σχετικός γερμανικός όρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να γίνει το ίδιο, αλλά σε ένα ε, διαθεσμικό πλαίσιο. Και αυτό το οποίο μας εκπλήσει, αν δούμε τα πράγματα εκ του μακρόθεν, είναι ότι υπάρχει μια θεσμική συμφωνία μεταξύ των τριών επικεφαλής ε, του τριγώνου για τον ε, προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός ουσιαστικά είναι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά τι γίνεται ως προς τους στόχους, πού είναι η συμφωνία. Έγιναν διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ζαν Κλοντιούνκερ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε ένα πρόγραμμα δράσης. Βεβαίως και θα υπάρχει το ετήσιο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την άλλη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθόρισε ποιες είναι οι προτεραιότητες Σαφώ του. Σαφώς υπάρχουν και διαφορές, υπάρχει και διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, Συμβουλίου, αλλά πού είναι η συμφωνία η οποία θα καθορίσει ουσιαστικά έναν χάρτη πορείας ε, για τη συνέχεια. Ε, ναι, εντάξει, όλα αυτά θα προσαρμοστούν από εκεί και πέρα, αλλά ίσω θα έπρεπε να επισημοποιηθούν κάπω τα πράγματα και για τη συνέχεια. Αυτό είναι το στρατηγικό πλαίσιο. Και μία τελευταία παρατήρηση οι πρωτοβουλίες οι οποίες θα αναλυθούν από την Επιτροπή Juncker και ε, οι δράσεις που θα προωθήσει, διότι όπως σας είπα αυτό είναι καθοριστική σημασία για την ομοποίησή της και φυσικά και για την αποτελεσματικότητά της. Εδώ υπάρχει μια σημαντική πρόκληση ε, με διαφιλονικούμενες προσδοκίες οι οποίες προέκυψαν και από τις ευρωεκλογέ και υπάρχουν και διαφορές οι οποίες ε, διαφάνησαν και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ είπε ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει με αποφασιστικό τρόπο ε, στις μεγάλες προκλήσεις ε, και να μην χρειάζεται να δώσει τόσο μεγάλη σημασία στις μικρές προκλήσεις. Είναι πολύ συγκεκριμένη απόφαση και είναι και παιδαγωγικού χαρακτήρα. Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας προκύπτει από το γεγονός ότι ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουν υπόψη τους την επικουρικότητα μέχρι τέλους. Εάν χαθεί αυτός ο σύνδεσμος ότι το 80% τη νομοθεσία που εγκρίνονται σε επίπεδο κράτους μέλους προέρχονται από τις Βρυξέλλες, ε, τότε ε, μπορεί να μην έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Αν δεν διευκρινίσει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, ότι από εδώ και πέρα σε επίπεδο οικονομικό και νομισματικό υπάρχουν ε, αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται συγκεκριμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια ελευθερία για να λαμβάνονται αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να φανεί κάπου αυτός ο παιδαγωγικός χαρακτήρας, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ αυτού του οποίου προέκυπτει ε, ακρεφνώς από τον ε, νόμο και ε, κάποια άλλα τα οποία προκύπτουν από κάποιες μικρές λεπτομέρειες που μπορεί ας πούμε να διαφύγει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί αυτές είναι οι λεπτομέρειες, οι κανόνες δε μήνυμης, με τις οποίες ασχολείται η Επιτροπολογία. Ε, και εδώ πρέπει να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ έχουμε και τον παιδαγωγικό αυτό χαρακτήρα. Επίσης υπάρχει και ανάγκη να δράσουμε ε, και λίγο προληπτικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να τα κάνει τα πάντα και φυσικά δεν μπορεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να το πούμε. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε περισσότερα ε, και να είναι πιο ισορροπημένη η προσέγγιση μας. Το να κάνουμε λιγότερα σε κάποια ε, ζητήματα σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση ε, τεχνικο-οικονομική στο κόστος της μη Ευρώπης. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τίμημα να πληρώσουμε όλοι για τη μη Ευρώπη, αλλά υπάρχει και ένα τίμημα να πληρώσουμε για την υπερβολική Ευρώπη. Μπορεί να είναι λίγο υποκειμενικό, να ακούγεται υποκειμενικό, αλλά υποκειμενικότητα είναι τμήμα της ζωής μα και τη πολιτική ζωή. Επομένως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα και να πει ότι ναι, σε κάποιου τομείς ε, πρέπει να κάνουμε περισσότερα και θα πρέπει φυσικά να καλύψουμε και τις προσδοκίες και να λάβουμε υπόψη τις προσδοκίες των πολιτών και υπάρχουν κάποια άλλα θέματα στα οποία θα πρέπει να γίνουν λιγότερα. Και φυσικά και ο κύριος Τίμερμανς έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, αλλά σίγουρα αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον ελεγχό σας και με τη βοήθειά σας να μπορέσει να ε, εξισορροπήσει τον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγει τις πολιτικές της για τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτά λοιπόν εν είδη ε, εισαγωγής. Ελπίζω να επανέλθουμε στα θέματα αυτά στη συνέχεια της συζήτησης. Ευχαριστώ. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο ε, θεσμικό όργανο, το Συμβούλιο. Και τώρα έχουμε τον, τον καθηγητή κύριο Πίτερ από το Κεντρικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Βουδαπέστη και που έχει κάνει πολλές δημοσιεύσεις και έχει εργαστεί πάρα πολύ και για το Συμβούλιο και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οπότε έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Αυτό που θα ήθελα να κάνω κατά τη διάρκεια των επόμενων 15 λεπτών είναι να παρακολουθήσουμε ένα θέμα το οποίο απέκτησε ιδιαίτερη σημασία στη διάρκεια της κρίσης. Αλλά πιστεύω πως είχε απασχολήσει τους ερευνητές πολύ προηγούμενα δηλαδή ε, τον αυξανόμενο ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Δεν σημαίνει πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο δεν έπαιζαν ανέκαθεν ε, ένα σημαντικό ρόλο στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ε, περισσότερο αυτό θα γίνει στα επόμενα χρόνια, ότι δηλαδή και οι δύο θεσμοί έχουν κατά κάποιον τρόπο αναπροσανατολιστεί ε, στο πλαίσιο της καινούργιας δυναμικής που διαμορφώνεται. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας ε, εξηγήσω είναι γιατί διαπιστώνουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο σε πάρα πολλού ε, τομεί ε, δραστηριοτήτων. Και επίση πρέπει να διερωτηθούμε κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε κάτι σχετικά με δραστηριότητε του Συμβουλίου, κυρίω ε, με όργανα όπω είναι το Eurogroup ή για το θέμα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, πάλι σε σχέση με το Eurogroup. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε λιγάκι τι ακριβώ συμβαίνει με αυτού του θεσμού. Πρώτα απ' όλα, το σημείο κίνησης για να κατανοήσουμε αυτό τον όλο και μεγαλύτερο ρόλο των ε, διακυβερνητικών ε, οργάνων είναι το εξής. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αν θέλετε, έχει κερδίσει πάρα πολλά μετά το Μάστριχτ ε, όσον αφορά την προβολή που του προσφέρεται ως προς τη λήψη αποφάσεων. Και θα σας εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Η ολοκλήρωση μετά το Μάστριχτ σε μεγάλο βαθμό βασίζεται σε ένα παράδοξο. Ότι από τη μια πλευρά αναφέρεται όλο και περισσότερο υποχρέωση ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ολοκλήρωση κυρίως σε τομείς που δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονταν συστηματικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά παρελθόν και εδώ το Μάστριχ ήταν ημερομηνία ορόσημο. Όμως τα κράτη-μέλη δεν επιθυμούν ανθίστανται στο να εκχωρήσουν αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων σε κλασικούς υπερεθνικούς οργανισμούς όπως είναι η Κομισιόν ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εμείς οι αναλυτές και άλλοι που ασχολούνται με την πολιτική σκέφτηκαν καταρχήν ότι αυτή ήταν μια μεταβατική ρύθμιση. Όμως αυτό που βλέπουμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι ότι τελικά προκύπτει ένα νέο είδος διακυβερνητισμού στην ε, διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο θα πρέπει να το αναλύσουμε σε βάθος και να δούμε τις πρακτικές του προεκτάσεις βλέπουμε ότι προκύπτουν νέες δραστηριότητες, νέοι τομείς πολιτικής που συστήθηκαν μετά τη συνθήκη του Μάστριχτ. Αναφέρομαι κυρίως στην οικονομική διακυβέρνηση και στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, ε, στην ΚΠΑ, στο συντονισμό πολιτικών και σε μεγάλο βαθμό ε, σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων θέματα τα οποία προέκυψαν και εξετάζονται στο πλαίσιο μιας ε, κοινοτικής μεθόδου. Με λίγα λόγια πιστεύω ότι υπάρχει μια λογική πίσω από το ότι ο συντονισμός ε, πολιτικών είναι ένας εναλλακτικός μηχανισμός λήψης αποφάσεων για ε, να νομοθετούμε. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε και να κατανοήσουμε και τις συνέπειες για την εξέλιξη των θεσμών κυρίως έχοντας κατά νου το μοντέλο της ε, αποκέντρωσης και όχι το κλασικό μοντέλο της ε, ολοκλήρωσης. Παναλαμβάνω λοιπόν, η συνθήκη της Λισαβόνας επιβεβαίωσε όλα αυτά, κυρίως όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση και αποκλεί την ε, λήψη νομοθετικών αποφάσεων, κυρίως στην ΚΠΑ, Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε λιγάκι τις σχέσεις ανάμεσα στους θεσμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πιστεύω, μία συνέπεια αυτού του προβλήματος, το οποίο προκύπτει από το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με μοντέλα αποκεντρωμένης πολιτική, όπου ε, τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που σε τελική ανάλυση λαμβάνουν τι αποφάσει σε πάρα πολλού νέου τομεί είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνένεση για συγκεκριμένα θέματα αλλά και η Κομισιόν γίνεται καθοριστικό παράγων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είτε αποκτά κανεί ε, τη συνένεση είτε δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και όπω ξέρουμε η συνένωση είναι πολύ εύθραυστη, άρα δηλαδή υπάρχει μόνιμη πρόκληση στη, ε, στη λήψη αποφάσεων. Ε, Βλέπουμε ότι σε θέματα από τη συνθήκη της Λισαβόνα έχει αμφισβητηθεί η συνένεση και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί κάποια συγκεκριμένη πολιτική γιατί όπως σας είπα ε, δεν προέκυπτε δέσμευση ή υπήρχε κάποια αντίδραση ε, στα κράτη-μέλη. Είδαμε ότι προέκυψε κρίση, κυρίως σε θέματα οικονομικής διακυβέρνησης ε, και οποτεδήποτε όμως λαμβάνονται αποφάσεις προκύπτουν πολύ σημαντικές προεκτάσεις, άρα δηλαδή πρέπει αυτή η υπηρχε καποια αντιδραση στα κρατη μελη ειδαμε οτι προεκυψε κριση κυριως σε θεματα οικονομικης διακυβερνησης και οποτεδηποτε ομως λαμβανονται αποφασεις προκυπτουν πολυ σημαντικέ προεκτασεις αρα δηλαδη πρεπει αυτη η διαδικασια της συνένεσης εσεί να είναι επιτυχή. Εξάλλου, στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων βλέπουμε και εκεί να υπάρχουν παρεμφερεί προκλήσει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πάντα ότι οι διαδικασίες και στέφεται από επιτυχία. Αυτό όμω που διαπιστώνουμε τα τελευταία 20 χρόνια είναι ότι καταβάλλονται προσπάθειε για να επενδύσει κανεί στην ε, απόκτηση συνένεση. Μεγάλε προσπάθειε. Επίση, ε, υπάρχει κάτι άλλο που σχετίζεται με όλα αυτά. Η ε, ανάληψη πρωτοβουλειών στον τομέα τη πολιτική και η εκχώρηση αυτών δεν μπορεί να λαμβάνει η χώρα ε, στην προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μια συλλογική διαδικασία. Βεβαίω και περιλαμβάνεται η Κομισιόν, αλλά και τα κράτη-μέλη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Κατόπιν τούτου, λόγω του ότι υπάρχει αυτό το συγκεντρωτικό μοντέλο, τα κράτη-μέλη πρέπει να δεσμεύονται ότι θα επιδιώξουν συγκεκριμένους στόχους, ε, να ε, δουν τι μπορούν να κάνουν με περίπτωση αποτυχίας και εδώ ε, τα οι οργανισμοί, αυτοί οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Οι αποφάσει μετά την κρίση, το six pack και το two pack αυτά δεν θα αλλάξουν. Γιατί τα θέματα που διακυβεύονται εδώ ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι η Κομισιόν έχει σημαντικότερο ρόλο εποπτείας, αυτή η μορφή συλλογικής ε, διακυβέρνησης και συλλογικής ε, πολιτικής, αυτή η μορφή ε, θα εξακολουθήσει να υπάρχει και θα ενταθεί περαιτέρω λόγω του ότι ο συντονισμός είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι υπήρχε κατά τα τέλη της δεκαετίας του 90 όταν ξεκίνησε η οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό λοιπόν που βιώνουμε εδώ και η μελέτη μου αυτά αφορά, δεν είναι απλά μία θεωρητική σκέψη, αλλά βλέπουμε ότι όλα αυτά έχουν και πρακτικές επιπτώσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής. Και βλέπουμε ε, να παίζουν ρόλο και οι αποχρώσεις ε, στους θεσμούς, ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αλλά και σε επίπεδο Συμβουλίου. Και θα αναφερθώ σε αυτά εντός ολίγου. Πολύ συχνά λοιπόν αυτές οι διαδικασίες που ακολουθούν οι θεσμοί έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στους σημαντικότερους εκπροσώπους των κρατών μελών αφενός και την Επιτροπή Αφετέρου. Μιλάμε εδώ για διοργανικές θέσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κομισιόν ε, αναλαμβάνει πολιτικές πρωτοβουλίες αλλά στο τέλος της ομιλίας μου θα σας δείξω ότι όλα αυτά έχουν σημαντικές επιπτώσεις και στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα βασικό στοιχείο αυτής, αυτού του νέου ε, διακυβερνητισμού είναι ο καθοριστικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και εδώ πρέπει να δούμε πώς θα το εξηγήσουμε αυτό. Δεν είναι μόνο το Συμβουλίο, δεν είναι μόνο μία τεχνοκρατική διαδικασία, είναι οι πρωθυπουργοί και οι αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων που παίζουν σημαντικό ρόλο και αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε και νέε δραστηριότητε, κυρίω, σα είπα, οικονομική διακυβέρνηση, στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, αλλά και στην κοινωνική πολιτική και στην απασχόληση. Στα τέλη τη δεκαετία του 90, τότε υπήρχαν πάρα πολλέ επιπτώσει από το συντονισμό των πολιτικών και οι επιπτώσει αυτέ γίνονταν αισθητέ σε επίπεδο κρατών μιλών. Εκεί πρέπει να είμαστε επιτυχημένοι και πρέπει πρέπει να δεχτούμε ότι έχουν αλλάξει οι πολιτικές των κρατών μελών και προκύπτουν συνέπειες για τις κυβερνήσεις. Η κρίση προφανώς είναι ένα καθαρό παράδειγμα, αλλά μπορούμε και να σκεφτούμε μέχρι ποιο βαθμό οι οικονομικές και οι δημοσιονομικές πολιτικές, κυρίως ο συντονισμός τους, έχουν επιπτώσεις. Αυτό το βιώσαμε κυρίως κατά τη διάρκεια της κρίσης και αυτό αποτελεί μια εξήγηση για το γιατί οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων εντάσσονται σε αυτή τη διαδικασία. Οι παρεμβάσεις λοιπόν υψηλού επίπεδου είναι ένα κλειδί για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Αν δεν υπάρχει αυτός ο συντονισμός σε ανώτατο επίπεδο τότε δεν προκύπτει και πρόοδος. Επίσης ε, κάτι άλλο που θέλω να πω και νομίζω αν δει κανείς ε, το θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εγώ το έχω δει, δει θέματα πούμε, που έχουν εξεταστεί κατά τα τελευταία 20 χρόνια από την εποχή του Μάστρικ και διαπίστωσα ότι από το δεύτερο ήμιση του 90 ε, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ασχολούνται περισσότερο με θέματα οικονομικά και εξωτερικής ε, πολιτικής. Ε, περίπου τα δύο τρίτα όλων των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι οικονομικά και εξωτερικών υποθέσεων. Αυτά συζητούνται σε κάθε συνεδρίαση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και αν δούμε λιγάκι το χρόνο που δαπανάτε για αυτά τα θέματα, θα δείτε ότι επιβεβαιώνεται αυτή η άποψή μου. Περίπου το 60% αφιερώνεται μόνο σε αυτά τα δύο θέματα. Και αν δείτε λιγάκι και τη συχνότητα των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αρχικά είχαμε τρει συναντήσεις το χρόνο, τώρα έχουμε φτάσει στι 7 και μάλιστα σε κάποια έτη φτάσαμε και μέχρι 11 συναντήσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ε, Πολλέ ήταν ε, χωρίς ε, μακροπρόθεσμο προγραμματισμό κατά την περίοδο της κρίση το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναλαμβάνει όλο και περισσότερο καθήκοντα άλλων θεσμών και εδώ αναφέρομαι κυρίως σε θέματα όπου είναι απαραίτητο να υπάρχει καθοδήγηση εντολές που δίδονται προς την Κομισιόν αλλά και προς το Συμβούλιο. Και δεν μιλάμε για γενικές κατευθυντήρες γραμμές αλλά μιλάμε για θέματα που έχουν σχέση με το 2-pack και το 6-pack. Ε, πρέπει να δίδονται εντολές ε, να ε, μην υπάρχουν ανεξάρτητες ε, πρωτοβουλίες. Έτσι λοιπόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε βασικά θέματα όπου υπάρχουν καινοτομίε και εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Σε σχέση με όλα αυτά έχει και το, θέμα το, της αναδιάτοξης των θεσμών ε, σας είπα, μίλησα για το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά αυτές οι μεταρρυθμίσεις ε, ε, δυσδύουν και σε άλλα επίπεδα, σε αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις. Κατόπιν τούτου Υπάρχουν κάποια στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για αυτή τη διαδικασία. Το άτυπο των συνεδριάσεων. Είχε μύθια Πολλές φορές ε, οι συνεδριάσεις ε, τελειώνουν αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία ε, σε προσωπικές συμφωνίες και σε κατηδίαν συζητήσεις. Βλέπουμε να υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ευελιξία στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υπάρχουν συναντήσεις ad hoc, αλλά υπάρχουν και θεσμοθετημένες συναντήσεις σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Και κάτι που είναι πάρα πολύ πολύ σημαντικό στη συνθήκη της Λισαβόνας. Όλο και περισσότεροι είχαν κάνει κασίες για τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού του Συμβουλίου μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Εδώ μιλάμε για ένα θεσμοθετημένο ρόλο ο οποίος έχει ως στόχο περισσότερο να μεσολαβεί για την επίτευξη συμφωνίας. Δεν θα αναφέρω κάποια στατιστικά δεδομένα για τις εξελίξεις που έχουν προκύψει. Πάρα πολύ σύντομα ε, θα ήθελα να πω κάποια άλλα θέματα γιατί πια δεν έχω χρόνο. Θέλω όμως να πω ότι βλέπουμε αυτές οι εξελίξεις αντικατοπτρίζονται στο Συμβούλιο. 13 Συμβούλια έχουν διαμορφωθεί ε, για θέματα συντονισμού πολιτικής, αποκεντρωμένης ε, πολιτικής, ε, θέματα οικονομικά, εξωτερικών υποθέσεων, κοινωνικές εξελίξεις. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι το Eurogroup και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων βρίσκονται στο επίκεντρο όλων αυτών των διαδικασιών. Βλέπουμε να έχουν προκύψει και διάφορα διάφορες άτυπε μέθοδοι εργασίες, όμως ε, και άλλε θεσμοθετημένες, όπως σας είπα, το Eurogroup και το ε, Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Μπορεί να μην φαίνονται τόσο πολύ ε, κάποιες αποφάσεις και γι' αυτό και εξηγούνται κάποια προβλήματα που έχουν προκύψει. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι το ΕΠΣΚΟ ασχολείται κυρίως με νομοθετικές διαδικασίες και είναι κάτι τελείως διαφορετικό ας πούμε από το Eurogroup ή από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που δεν αγγίζουν θέματα νομοθετικά. Φτάνω λοιπόν στην τελευταία μου παρατήρηση. Ας δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις αυτής της ε, νέας διαδικασίας που έχει προκύψει για δημοκρατικό έλεγχο ε, της νέας τάξης πραγμάτων. Υπάρχουν προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο δημοκρατικός έλεγχος. Ε, αυτό που έχουμε τώρα δεν είναι εύκολο δεν διευκολύνει την καλύτερη νομιμοποίηση, αλλά κατ' ουσίαν απλά αναδιατάσσει τις ήδη υπάρχουσες απόψεις για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Εγώ πιστεύω ότι οι κυβερνητικοί φορείς, όπως σας είπα, είναι επιφυλακτικοί και αυτό απαιτεί νέους θεσμούς και νέες ε, απαντήσεις. Αυτό είναι απαραίτητο τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και σε επίπεδο Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αρχίσαμε να λέμε ότι εκτός από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ίσως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να θεωρηθεί ο θεσμός εκείνος ο οποίος έχει αποκτήσει πάρα πολλές αρμοδιότητες μετά το Μάστριχ. Όμως το παράδοξο είναι ότι όλες οι διαδικασίες και οι αρμοδιότητες που έχει αποκτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν σχέση με το νομοθετικό έργο. Και εδώ προκύπτει μια ένταση. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη τοποθετηθεί ως προς αυτήν την πρόκληση. Έχει αυξήσει τον έλεγχο των νέων τομέων δραστηριοτήτων. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι δραστηριοποιείται η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, οι ακροάσεις. Μία σημαντική δυσκολία όμως είναι η εξής, ότι δεν μπορεί κανείς ε, τα άτομα, οι πρόεδροι να είναι υπόλογοι, προσωπικά υπόλογοι. Σε κάποιο βαθμό μόνο. Γιατί δεν εκφράζουν απαραίτητα ως άτομα την ευρύτερη πολιτική. Κατόπιν τούτου θεωρώ ότι ο ρόλος ε, του ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικός, άπτεται πολλών θεμάτων. Οι εξουσίες του βέβαια είναι αρκετά περιορισμένες και εδώ καλούνται τα εθνικά κοινοβούλια να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο. Τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να ελέγχουν τις κυβερνήσεις τους ως προς τη συμμετοχή τους στο Eurogroup ή στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έχουμε λοιπόν ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε, αλλά αν δούμε λιγάκι τη διαδικασία λήψη αποφάσεων σε νέους τομείς πολιτικής, τα εθνικά κοινοβούλια διαπιστώνουμε ότι έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν κυρώσεις, να επιπλήξουν, αν θέλετε, τις κυβερνήσεις τους και να τις ελέγξουν. Τελειώνω με την αναφορά ενός προβλήματος το οποίο δεν έχει εξεταστεί κατά την άποψή μου ότι τελικά είναι απαραίτητο να υπάρχει μια διτή απάντηση και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προς τα Εθνικά Κοινοβούλια. Μάλλον και οι δύο αυτοί φορείς καλούνται να δραστηριοποιηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και τώρα θα κινηθούμε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον καθηγητή Ολιβιέ Κώστα που είναι Διευθυντής ε, Σπουδών στο Κολέγιο της Ευρώπης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ ε, για την πρόσκληση ε, κλήθην από τους διοργανωτές να γράψω στα γαλλικά και να μιλήσω στα γαλλικά. λοιπόν, να το πω γαλλικά μου ζήτησαν ε, να ε, μιλήσουμε για, να μιλήσω για το θέμα των προκλήσεων που έχει να μετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ομοθέσια τον έλεγχο και τη διοργάνωση. Είναι τεράστιο το θέμα βέβαια. Ε, θα αναλύσω κάποια από αυτά τα θέματα υπό το αγωνιώδες βλέμμα ορισμένων ευρωβουλευτών. Να μιλήσω καταρχήν για μια πραγματική δυσκολία ε, εάν σκεφτεί κανείς ε, τη στρατηγική του Ευρωκοινοβουλίου για τα επόμενα πέντε χρόνια, είναι, ε, θα πρέπει να δει ότι έχει στόχους αντιφατικούς. Έχει την, το στόχο της αντιπροσωπευτικότητας, θα πρέπει το Ευρωκοινοβούλιο να εξακολουθήσει να αντιπροσωπεύει την, πολυ, την χαρακτήρα των μελών, των πολιτών κτλ. Έπειτα έχουμε θεσμική πρόκληση, δηλαδή πρέπει να αντιποκριθεί στις προκλήσεις που είναι οι δικές του, στις αποστολές του και να ανταποκριθεί και στο θέμα του ορθολογισμού, εξορθολογισμού από τότε που εισήχθη ενιαία πράξη. Επίση, το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να είναι δημοκρατικό και να διατηρήσει δημοκρατική λειτουργία του, πράγμα το οποίο δεν είναι πάντοτε συμβατό με, τις με τα προηγούμενα ε, αιτήματα. Επίση, η ορθή λειτουργία, χρηστή λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου που καλείται να συνεργάζεται τακτικά και αγαστά με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και εδώ μπορεί να υπάρξει αντίφαση. Και τέλο υπάρχει άλλη μια, μια απέτηση που είναι η λογοδοσία. Η λογοδοσία που πρέπει να δώσει το Ευρωκοινοβούλιο στου εκλογείς τους, τα ΜΜΕ, στους ε, ε, υπεύθυνου για το σχηματισμό της κοινή γνώμης, πράγμα το οποίο μπορεί και να περιορίσει τη λειτουργία του και αυτό είναι ένας ε, κάπω αντιφατικό ρόλος με τους στόχους τους προηγούμενους. Θα ξεκινήσω με τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το Κοινοβούλιο σε νομοθετικό επίπεδο. Καταρχήν, οι τριμερείς διάλογοι που σήμερα αντιπροσωπεύουν το 90% της νομοθεσίας και που υιοθετούνται από το στάδιο της πρώτης ανάγνωσης στην περίπτωση ε, νομοθεσίας με περιορισμένο αριθμό φορέων ε, ε, και κλεισμένων των θυρών. Φυσικά αυτό θέτει το πρόβλημα ορατότητας όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά θέτει και θέματα εσωτερικής νομιμότητας εντός του Ευρωκοινοβουλίου γιατί ε, το, η απόφαση θα ληφθεί από τρεις-τέσσερις ε, βουλευτές ε, βοηθούμενος από κάποιους υπαλλήλου, αλλά με διαφάνεια που δεν είναι η βέλτιστη. Και ξέρω πως το Ευρωκοινοβούλιο έχει προσπαθήσει να αναπτύξει τις διαδικασίες για να πλαισιώσει αυτή την πρακτική αλλά νομίζω πως δεν υπάρχει ακόμα η αρκετή δυνατότητα ε, στρατηγικού προβληματισμού όσον αφορά το κέρδος για τις επιτροπές ε, της τριμερής αυτές. Κάποιες φορές ε, χασκογελάνε οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου όσον αφορά την αθωότητα, την αγαθοσύνη των ευρωβουλευτών, αλλά έτσι δεν μπορούν ίσως να αντιμετωπίσουν τις εκθέσεις που ίσως να αξίζει να φύγουν από τις πρώιμες αποφάσεις, πρώιμες συμφωνίες και να περάσουν επίσης από αυτή τη διαδικασία του τριλόγου. Έπειτα, σημαντική, άλλη, άλλη ε, σημαντική πρόκληση είναι ε, τη πρωτοβουλία, η νομοθετική που του αποδόθηκε από το Μάστριχτ και τώρα έχει κωδικοποιηθεί στο άρθρο 225, αλλά που δεν έχει πολύ καλέσει την ε, συμφωνία των Ευρωβουλευτών, αλλά ούτε και της Κομισιόν που κατά κάποιο τρόπο κακομεταχειρίζεται το Ευρωκοινοβούλιο όταν προβαίνει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Και άρα το Ευρωκοινοβούλιο βρίσκεται σε ανταγωνισμό με άλλα θεσμικά όργανα που έχουν επίσης το δικαίωμα για νομοθετική πρωτοβουλία αλλά και από το Συμβούλιο το οποίο ορίζει σήμερα την νομοθετική ατζέντα για τα μισά σημεία και το Ευρωκοινοβούλιο ε, μπορεί να έχει μεγαλύτερη εξουσία μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας με τους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να αντιμετωπίζει τουλάχιστον το, με τον ίδιο τρόπο το Κοινοβούλιο όπως με τις πρωτοβουλίες των πολιτών, να είναι δηλαδή αντικείμενο ανακοινώσεων. Επίσης το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να τοποθετηθεί ως ένας πρώτος τάξης συνομιλητής όσον αφορά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που στόχο έχουν να χρησιμοποιηθεί η πρωτοβουλία των πολιτών, η οποία θα πρέπει να είναι μια διαδικασία τελευταίας διαφυγής και ότι καταρχήν το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να τοποθετηθεί ως ο πρώτος συνομιλητής για αυτά τα θέματα, λέγοντας ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να προβούμε σε νομοθετική πρωτοβουλία και να μην τρέχουμε να μαζεύουμε ένα εκατομμύριο υπογραφές. Κάτι ακόμα σε νομοθετικό επίπεδο που είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι ε, η διαδικασία των εκκρεμών προτάσεων που θα γίνει με τη νέα Επιτροπή. Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ήταν ξεκάθαρο στην επιστολή στον ε, κύριο Τίμερμαν ε, ζητώντας του να επανεξετάσει όλες τις εκρεμείς νομοθετικέ διαδικασίε προτάσεις και επιμένοντας σε μια νέα αρχή της ε, πολιτικής ασυνέχειας. Ο κύριος Γιούνκερ ε, μοιάζει με μια κυβέρνηση λοιπόν κατά τον κύριο Γιούνκερ και όχι με μια, ένα διοικητικό μηχανισμό και ότι δεν θα δώσει τα συνέχεια σε όλες τις προτάσεις ε, Μπαρόζο, της Επιτροπής Μπαρόζο. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος πολλές προτάσεις να αποσυρθούν. Οι εκρεμείς προτάσεις δεν μπορούν να αποσυρθούν έτσι ε, αθώα. Είναι πολιτικές κινήσεις αυτές. Αν λοιπόν πολλές πρωτοβουλίες εκκρεμής ε, αποσυρθούν θα πρέπει να επανεπαβληθούν ε, το 16, το 17 εν ώψη των ευρωεκλογών και το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να βρεθεί σε τρελή πίεση από πλευρά ατζέντα και όπως τις προηγούμενες θητείες να οδηγηθεί να υιοθετήσει τόσα κείμενα στα τελευταία χρονιά εντολής του, όσα κατά τη διάρκεια των τριών προηγουμένων ετών. Άρα δηλαδή να υποχρεωθεί σε πρώτη ανάγνωση να τα εγκρίνει όλα και να μην μπορεί να μπει στην ουσία των θεμάτων. Όσον αφορά τους πολιτικούς ελέγχους, ε, ε, Εμβέαθηναν εκεί οι δύο συνάδελφοι. Ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω πως είναι σημαντικό το Ευρωκοινοβούλιο να καταφέρει να διατηρήσει τον πολιτικό διάλογο που έχει ήδη θεσπιστεί με την ευκαιρία αυτής της νέας αιτία και έχουμε μπει σε μια νέα φάση, σε μια νέα φύση του διαλόγου και είναι προς το συμφέρον του Κοινοβουλίου να διατηρήσει αυτό το διάλογο θα έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο θα επιδράσει το Κοινοβούλιο με τους 7 αντιπροέδρους, ε, γιατί υπάρχουν τεχνικά θέματα. Ποια είναι η επιτροπή που θα έρθει σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, πώς θα μπούμε σε επαφή με τους επιτρόπους και τους αντιπροέδρους που κατά κάποιο τρόπο ηγούνται αυτών. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα λύσει η Γραμματεία, αλλά θα πρέπει να προσέξει πολύ το Κοινοβούλιο, κυρίως αν φανεί πως ο αντιπροέδρος κατά κάποιο τρόπο ελέγχει την νομοθετική ατζέντα της Κομισιόν. Και εδώ νομίζω πως θα πρέπει να γίνει μια στρατηγική σημασία σε επιλογή για το Ευρωκοινοβούλιο. Παραμένει το Κοινοβούλιο σε μια λογική ε, θεσμικής ανεξαρτησίας που είναι στο γενετικό του κώδικα από το ε, δεκαετία του 50 ή μήπω μπαίνει σε μια λογική στήριξη της Κομισιόν ε, για να μπορέσει να επιτύχει για παράδειγμα ο κύριος Γιούνκερ να διαβουλευτεί με τους ηθήνοντες των τριών μεγάλων ομάδων πριν να ε, συντάξει νομοθετικές προτάσεις, να μπορέσει δηλαδή κάπως έτσι να ψηφίσει συλλαφίσει ε, το έδαφος ε, στο Ευρωκοινοβούλιο όπως το κάνει και με το Συμβούλιο Κομισιόν. Όπως είπε τώρα ο συνάδελφος Πούτερ, είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να δίνει μεγάλη σχέση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η υπόθεση με τον κύριο Βαν Ρομπάη, που ήταν ε, θετικά διατεθειμένος απέναντι στο Ευρωκοινοβούλιο. Η πρωτοβουλία του Ευρωκοινοβουλίου δεν σημαίνει ότι δεν, ε, ε, δεν χρειάζεται το Συμβούλιο να δίνει λογαριασμό, να λογοδοτεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή είναι μια βασική λειτουργία. Εφόσον ο πρόεδρο του Συμβουλίου έρθει εδώ θα πρέπει να αιτιολογήσει και τις επιλογές του και να τις εξηγήσει. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό για το ρόλο που παίζει το Ευρωκοινοβούλιο στη συζήτηση των ευρωπαϊκών θεμάτων. Τρίτο, η πρόκληση του ελέγχου είναι πιο τεχνικής φύσης, έχει να κάνει με τις ε, κατεξουδότητες πράξεις και την επιτροπολογία. Εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή από πλευράς του Ευρωκοινοβουλίου Ξεκινά μια διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή από αυτού του θέματος και, η Ευρωπαϊκή, και το Ευρωκοινοβούλιο χρειάζεται να δώσει απόλυτα η προσοχή γιατί εδώ κρύβεται με πολύ πολιτική και συχνά υπάρχει έλλειψη των Ευρωβουλευτών για τόσο έτσι, ε, άχαρα θέματα. Υπάρχουν διαδικασίες πριν τη Λισαβόνα και νέες διαδικασίες, πολλές ad hoc διαδικασίες, ε, εξαιρέσεις, ε, ε, παρεκκλήσεις κτλ. Και υπάρχουν νομοθεσίες όπου οι κατεξουσιοδότηση νομοθεσίες βρίσκονται τελικά στα χέρια των υπαλλήλων και όχι στα χέρια των ευρωβουλευτών. Έχουμε πραγματικό έλλειμμα διαφάνειας απέναντι στους Ευρωκοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών και έπειτα υπάρχει το θέμα της κατανομής ανάμεσα στις κατεξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις. Ε, εδώ θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι ρετοί μας άρχοντες για τα θέματα αυτά και γιατί πρέπει όλοι να γνωρίζουν ε, ποια είναι τα διακυβεύματα αυτής της δευτερεύουσας νομοθεσίας και το Κοινοβούλιο να έχει περισσότερο διοικητικό, διοικητικά μέσα για να ασκήσει αυτό το καθήκον του που είναι πολύ άχαρο όπως είπα και τεχνικής φύσης. Έχει ευθύνη όμως το θέμα και νομίζω περισσότερο οι γραμματείες των επιτροπών, των κοινοβουλευτικών επιτροπών πρέπει να ασχολούνται με τα θέματα και όχι οριζόντια όργανα που δεν γνωρίζουν καλά τα θέματα και θα χρειάζεται διαφάνεια ακόμα και κατάρτιση του μικρόκοσμου των φορέων της, κοινωνικής, ε, της ε, κοινωνίας των πολιτών στην ε, μια ειδική κατάρτιση για να μπορούν να καταλάβουν τα θέματα της επιτροπολογίας καλύτερα. Τώρα, όσον αφορά την το Κοινοβούλιο το ίδιο για τη λειτουργία του, εξορθολογισμός. Χρειάστηκε να εξορθολογίζεται διαρκώς η λειτουργία του θεσμού. Έχουμε νέες αρμοδιότητες, άρα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό ήταν το ε, μότο. Ε, όμως ε, μέσω διαφόρων αναθεωρήσεων του κανονισμού τελικά γίνεται ανακατανομή των εξουσιών μέσα στο ίδιο το θεσμό. Δηλαδή τα ιεραρχικά ε, όργανα του, του, του Κοινοβουλίου, δηλαδή το Προεδρείο, η Διάσκεψη των Προέδρων και ένα περιορισμένο αριθμό βουλευτών, δηλαδή πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και οι βουλευτέ οι οποίοι συντάσσουν πολλέ εκθέσει, κάπω παίρνουν περισσότερη εξουσία. Και εδώ πρέπει να σκεφτούμε την ένταση που μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στη δημοκρατία από το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να είναι αποτελεσματικό για να έχει κύρος στο διαθεσμικό ε, παιχνίδι, αλλά και τη δημοκρατία εντό του ίδιου του δημοκρατίου. Δεν πρέπει να γίνουν όλα αυτά βάρο τη δημοκρατική λειτουργία του ίδιου του Κοινοβουλίου και τη εικόνα του. Και έτσι πάω στο δεύτερο θέμα μου. Η εικόνα, η δημόσια του σώματος είναι κάπως συγκεχημένη. Από τη μια πλευρά έχουμε ένα κοινοβούλιο που διαφοροποιείται όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητά του. Έχουμε διάφορους ευρωσκεπτικιστέ και πολιτικές ομάδες οι οποίες είναι λιγότερο συμπαγείς από πολιτικής άποψη. Αυτό μπορεί κανείς να το θεωρήσει καλό γιατί έχουμε έτσι ένα σώμα το οποίο αντικατοπτρίζει την κοινωνία. Δεν είναι γραφειοκρατικό όργανο το κοινοβούλιο αλλά μεταφράζει όλα τα χάσματα, τις αποκλήσεις που μπορεί να υπάρχουν στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε ένα σώμα το οποίο φαίνεται να διευθύνεται από μια συμμαχία που ισχύει ανάμεσα στο ΕΛ και τους σοσιαλιστές και την ΑΛΔΕ και υποστηρίζει την, την Κομισιόν. Και υπάρχει ο φόβος μήπως απλώς ε, το Κοινοβούλιο γίνει ένα, μετατραπεί σε ένα απλά διεκπαιρεωτικό όργανο οι κοινοβουλευτικές ε, επιτροπές κατανοούν πολύ καλά πώς μπορούν να λυθούν αυτά τα θέματα. Δηλαδή αναζητείται ναι μεν η συνένεση, αλλά θα πρέπει αυτό να γίνει μέσω διαπραγμάτευσης, επιχειρηματολογίας και ούτω καθεξής. Και πιστεύω πως οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και το Κοινοβούλιο δείχνουν μια κολακευτική εικόνα της Ευρωπαϊκής ε, Δημοκρατίας, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει πάντα στην Ολομέλεια, ε, λόγω των περιορισμών της των περιορισμών ε, της, του εξορθολογισμού. Τώρα, οι μελέτες αντικτύπου έχουν γίνει το Ευαγγέλιο και κατά κάποιο τρόπο όλα τα θεσμικά όργανα καλούνται να τις συγκρίνουν γιατί δήθεν όλα αυτά τα συντάσσουν οι επιστήμονες. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει αναπτύξει μια στρατηγική για να το καταπολεμήσει λίγο αυτό. Υπήρξε μια έκθεση το 2011 και μια ειδική επιτροπή που δημιουργήθηκε, μια μονάδα μάλλον που δημιουργήθηκε για να εκτιμά, να αξιολογεί τις ε, μελέτες αξιολο... Ε, αντικτύπου. Αλλά είναι μια μικρή μονάδα που ε, δεν έχει πολλές δυνατότητες. Πρέπει να επιβάλλουμε μια μελέτη αντικτύπου στους βουλευτές για τις τροπολογίες, να περιμένουν δηλαδή 6 εβδομάδες δεν μπορούν να καταθέσουν τροπολογίε που έχουν όμω πολιτικό νόημα χωρί να γίνει αυτή η μελέτη. Νομίζω πως έτσι γίνεται, μπαίνει τροχοπέδι στην εργασία των βουλευτών. Θα μπορούσαν να γίνουν μελέτες εξ εκ των υστέρων για να αξιολογείται η πολιτική αυτή και αυτό το κάνει η Οικονομική και η Κοινωνική Επιτροπή και είναι πάρα πολύ ε, ε, καλό αυτό, πολύ θετικό. Τώρα, στρατηγική καμπή στι διαθεσμικές σχέσεις βλέπουμε εδώ. Πρέπει να επανακαθοριστούν, να, να προσδιοριστούν. Εδώ πρόκειται για πολιτικές επιλογές ε, το θέμα της προσέγγισης ε, όσον αφορά την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ξανασυζητηθεί και τέλος πιστεύω πως υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο προόδου για το Κοινοβούλιο όσον αφορά τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες. Έχουμε νέες προσδοκίες όσον αφορά την νομιμοποίηση και τον εκδημοκρατισμό και ε, η μόνη, επιλυση... η λύση είναι περισσότερος κοινοβουλευτισμός και άρα πρέπει το Ευρωκοινοβούλιο να δράξει αυτή την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έχουμε 40 λεπτά στη διάθεσή μας για τη συζήτηση. Θα αρχίσω να ζητώ από τους συναδέλφους όσο γίνεται πιο σύντομη να είναι και να... Ε, αν θέσουν ερωτήσεις να είναι συγκεκριμένοι. Και αρχίζουμε με τον George Σέπλεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, θα είναι πολύ συγκεκριμένες οι ερωτήσεις και θα είμαι και πάρα πολύ σύντομος. Καταρχάς να σας καλωσορίσω όλους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δέσατε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις. Η πρώτη μου ερώτηση είναι για τον κύριο Μπετοντσίνη. Ευθύς εξ αρχής αναφερθήκατε στην ομοιοποίηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αλλά με εξέπληξε το γεγονό ότι δεν αναφερθήκατε στου πολίτε, δεν αναφερθήκατε και στου ενδιαφερομένου. Και έχω την εντύπωση ότι η νομιμοποίηση όλες της ευρωπαϊκής ε, διαδικασίας ε, δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτούς. Και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η αποψή σας επ' αυτού. Δεύτερη παρατήρηση, από περιέργεια και μόνο, είπατε ότι είναι πρόβλημα για κάποιες χώρες που δεν έχουν πια δύο επιτρόπους. Ε, μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω. Ε, ποιον έχετε κατά νου. Τρίτη παρατήρηση, η οποία προκύπτει ακριβώς από αυτό που μας είπατε. Αναφερθήκατε στη νέα αυτή δυνατότητα του speech and candidate και πραγματικά εγώ θεωρώ ότι αυτό αποτελεί σοβαρή αλλαγή στον θεσμικό, ε, στη θεσμική τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλό δε μάλλον όταν αναφερθήκατε στην τροποποίηση του άρθρου 17 17-7 για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες εξουσίες για τον ορισμό και την απόλυση επιτρόπων. Και θεωρώ ότι αυτό ουσιαστικά περικόπτει τις εξουσίες των κρατών μελών. Και θα ήθελα να ξέρω αν εσείς ε, το βλέπετε από το ίδιο πρίσμα. Και τώρα να σας πω δύο λόγια στον κύριο Πέτερ. Αναφερθήκατε Ε, νέες αλλαγές ε, στη διαδικασία ολοκλήρωσης ε, και είπατε ότι άλλαξε το κέντρο βάρους, αλλά εγώ θα ήθελα να ξέρω αν έχουμε την πολιτική βούληση που ξεκινά τη διαδικασία, η έλλειψη πολιτικής βούλησης που οδήγησε για παράδειγμα στην αποτυχία της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άμυνας. Θα ήθελα να ξέρω δηλαδή αν υπάρχει κάτι ποιοτικά διαφορετικό για τη δημιουργία συνένεσης σε σχέση με το που βρισκόμαστε σήμερα. Επίσης, θεωρείτε ότι οι θεσμοί του Συμβουλίου, τους οποίους αναλύσατε με πολύ ενδιαφέρον, μπορούν να έχουν κάποια ανεξαρτησία όσον αφορά την ε, ε, μέθοδο εργασίας και από τον τρόπο με τον οποίο ε, δρούν παραδοσιακά, αν θέλετε. Έχω την εντύπωση εγώ βέβαια είμαι εξωτερικός παρατηρητής, ότι όλοι σε κάποιο βαθμό είναι αποκομμένοι από τα κράτη-μέλη και θεωρώ ότι υπ' αυτή την έννοια ε, η θεσμική θεωρία θα λειτουργήσει λίγο διαφορετικά, σαν να είναι σε ένας διαφορετικός δικός τους κόσμος. Και το θέμα είναι ποια είναι η νομοποίηση αυτής της διαφορετικής λειτουργίας, πώς ελέγχεται, πού υπάρχει διαφάνεια και ούτω καθεξής. Και τέλος, προς τον κύριο Κώστα, το θέμα της αμφισημίας που αναφέρατε προς το τέλος της πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας, ε, δεν διαφωνώ μαζί σας σε καμία περίπτωση, αλλά εγώ από τα 10 και κάτι παραπάνω χρόνια που βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρώ ότι η διαχωριστική γραμμή δεν είναι μεταξύ αριστεράς και δεξιάς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει διαχωρισμό μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, αλλά η βασική διαχωριστική γραμμή είναι οι ευρωπαϊστές και οι μη ευρωπαϊστές. Ευχαριστώ, Υπερβάνη Περές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ στους τρεις εμπειρογνώμονες που μας διευκρίνησαν κάποια πολύ σημαντικά πράγματα και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό που γίνεται αυτή η ακρόαση στην αρχή της θητείας. Έχω τρεις ερωτήσεις για τον κύριο Μπερτονσίνη. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει την εποπτεία και να αφήνει την αυτονομία στα κράτη-μέλη. Λίγο τηλεγραφικά, αλλά λίγο πολύ αυτό μα είπατε. Δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα, διότι δίνει μια εικόνα πάρα πολύ αρνητική για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ε, θεωρούμε έτσι ότι απλώς υποπτεύεται ο ρόλος μας και αυτό νομίζω ότι δεν οδηγεί πουθενά. Νομίζω ότι προσπαθήσατε να πείτε ότι το πολιτικό κόστος της μη Ευρώπης είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως και το κόστος της υπερβολικής Ευρώπης, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένας χώρος για τους Ευρωπαίους πολίτες που κάποιος πρέπει να καταλάβει. Κύριε Πέτερ, εσείς είπατε ότι η διαφορά μεταξύ του νομοθετικού και του μη νομοθετικού είναι πάρα πολύ σημαντική. Και το βλέπουμε και σε τομείς όπως η οικονομική πολιτική, η πολιτική ανταγωνισμού, όπου βρισκόμαστε στο επίκεντρο των δυσκολιών, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε καθορίσει ένα νομοθετικό πλαίσιο και υλοποιούνται οι πολιτικές και εκεί μπαίνουμε στην ουσία του προβλήματος και εκεί είναι ε, το ερώτημα πώς μπορεί να παρέμβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ, για παράδειγμα, στην προ... Ε, η ηγούμενη θητεία είχα προτείνει το Κοινοβούλιο να είναι συνομοθέτης. Δεν έγινε βέβαια και τόσο πολύ καλά δεκτό. Ε, δεν θεωρώ ότι είναι αποδεκτά τα επιχειρήματα γιατί υπάρχουν πολιτικά κύματα και το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να παρέμβει αν θέλει. Συμφωνείτε εσείς προς αυτή την κατάσταση. Αναφερθήκατε επίσης στη σχέση μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και κρατών μελών και το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θεωρείτε ότι η λύση που εξευρέθη στο σύμφωνο σταθερότητας, ε, ε, στο δημοσιονομικό σύμφωνο, συγγνώμη, ε, λειτουργεί ή πρέπει να προσφέρουμε και άλλα. Προς τον κύριο Κώστα. Εσείς ήσασταν πάρα πολύ αυστηρός με τους τρισμερείς διαλόγους μεν, αλλά εδώ θα ήθελα να σας πω δύο πράγματα. Καταρχάς, το θέμα του χρόνου της θητείας, αυτό δεν είναι ε, θέμα κοινοβουλίου, πρέπει να το λέμε συνεχώς. Εάν μας πιέζουν να εγκρίνουμε πράγματα σε πρώτη ανάγνωση, είναι γιατί καθυστερεί το Συμβούλιο. Επομένω, ε, να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Δεύτερον, ναι, μεν, εντάξει, όλα αυτά δεκτά για τους ε, τριμερείς διαλόγους, αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος για τη διαφάνεια, ε, πρέπει και αυτό να το πούμε, τη διαφάνεια του Συμβουλίου. Πρέπει, είμαστε συνομοθέτες και από την άλλη υπάρχει διαφάνεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους τριμερείς διαλόγους και στο Συμβούλιο διαφάνεια μηδέν. Και απλώς ε, πρέπει να δεχτώμαστε αυτά τα μικρά θέματα που έχουν συζητήσει μεταξύ τους και έχουν συμφωνήσει κάτι φίλοι μεταξύ τους. Υπάρχει λοιπόν κάτι πάρα πολύ ε, κακό, το οποίο επινέωσε ε, ο ε, κύριος Μπαρόζο στο τέλος της θητείας του, το λεγόμενο ρίφιτ. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα μαύρο κουτί που δεν ξέρουμε τι θα το κάνουμε και είναι μια, ένας τρόπος να αποδομήσουμε τελείως τη συναπόφαση. Και να πω επίσης και κάτι που δεν ανέφερε κανένας από τους τρεις ομιλητές και που κατά την άποψή μου είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι κάνουμε τώρα ε, με τις ε, νομοθετικές εξουσίες ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η Λισαβόνα τα επιδίνωσε αυτά και έχουμε αρχίσει να κάνουμε λισαβονοποίηση των εξουσιών το είδαμε και στην προηγούμενη θητεία με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είτε όσον αφορά τα ποσά αυτά κάθε αυτά και όσον αφορά την νομοθεσία που απορρέει από αυτά. Και στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για θέματα κλίματος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λέει ότι θα μείνει εκεί που είναι. Τι θα πει αυτό. Ε, όσον αφορά τη διαδικασία της συναπόφασης λοιπόν, το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ συναντικό και κατά την άποψή σας τι θα έπρεπε να κάνουμε, τι πρέπει να αλλάγουμε για να μην είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συναπόφαση και να είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, όχι αυτό το οποίο κάνει συστάσεις, αλλά αυτό το οποίο τελικά καθορίζει απόλυτα τις πολιτικές. Ευχαριστώ, Ραμάν Χαουρέγγι. Καλημέρα σας. Να ρωτήσω τους εισηγητές δύο πράγματα, τα οποία έχουν σχέση με τη λεγόμενη απουσία νομοθετικής πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάποιοι από εσά ε, εξέτασαν ποια είναι η στατιστική συμπεριφορά τα τελευταία 20 χρόνια για τις ε, ε, εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου και πώς τις αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, το Κοινοβούλιο προσπαθεί να αναλάβει πρωτοβουλίες με εκθέσεις για θέματα τα οποία θεωρεί απαραίτητα, αλλά δεν έχουμε εμεί δυνατότητα νομοθετική πρωτοβουλία. Κάνουμε εκθέσεις και η ερώτησή μου είναι τι τις κάνει αυτές οι Ευρωπαϊκές Επιτροπές και αν ε, θα πρέπει ίσως να νομιμοποιήσουμε την ε, νομοθετική μας πρωτοβουλία με μεγαλύτερη ισχύ ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, όσον αφορά την υπόσχεση που έδωσε ο κύριος Γιούνκερ για την ιδέα του να υπάρχει συνένεση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν ε, αναλάβει τις πρωτοβουλίες τους. Αν μπορούσε αυτό να επισημοποιηθεί με κάποιο τρόπο, διότι εμείς δεν είμαστε ένα κοινοβούλιο ε, σύνηθες, δεν έχουμε μια πολιτική πλειοψηφία που να στηρίζει την κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισήμως δεν υπάρχει αυτό. Σε ε, πλαίσιο πολιτικής πρακτικής, ναι. Λίγο πολύ υπάρχουν κάποιες πολιτικές ομάδες που υποστηρίζουν και την ευρωπαϊστική δύναμη, θα έλεγα εγώ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι τόσο την οδεολογική και πολιτική στάση της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σαφέστατα εδώ υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ρεύμα το οποίο ενώνεται ε, και είναι υπέρ της προόδου της Ένωσης και της, ε, του θεσμικού ρόλου της Ένωσης. Και ε, διερωτώ με, ποιο τρόπο θα μπορούσε να επισημοποιηθεί η συνένωση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κυρίου Γιούνκερ ίσως και τους εκπροσώπους των μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων, ώστε οι κύριοι πολιτικοί στόχοι της νομοθεσίας να μπορούν να υλοποιηθούν. Ευχαριστώ. Ο Γιολάινεν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, δυστυχώς δεν μπόρεσα να ακούσω τον πρώτο μου. Ήρθα πολύ καθυστερημένα από το Βερολίνο. Μία ερώτηση προς τον κύριο Πίτερ. Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πράγματι ε, είναι μυστικοπαθές. Και θυμάμαι ε, αυτά που είπε η κυρία Περάνσο, όπου τα δύο τρίτα της ε, διακυβερνητικής ήταν αντίθετη στο να γίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, θεσμός και ε, επέρασε αυτή η άποψη και είχαμε υποψιαστεί ότι θα δημιουργήσει προβλήματα, ότι θα υπάρξει μετατόπιση από τους θεσμικούς οργανισμούς προς αυτούς τους διακυβερνητικούς και μέχρι και το Συμβουλίο. Και να, έγινε υπάρχουν και αποδείξει. Η κυρία σου το ανέφερε. Στη συνδιάσκεψη κορυφής του Οκτωβρίου, εκεί ήταν απαράδεκτο. Ακόμα και σε ποσοστά το Συμβούλιο διεκδίκησε το δικαίωμα να παρεμβαίνει τη στιγμή που ο νομοθέτης έχει λάβει διαφορετική απόφαση. Ενδέχεται λοιπόν να φτάσει αυτή η χρονική στιγμή όπου ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να βρεθεί υπόλογο απέναντι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να το εγκαλέσουν για παραβίαση καθηκών. Αναφέρθηκε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει περισσότερες αρμοδιότητες και μεγαλύτερη εξουσία. Και εγώ ρωτώ, πού οφείλεται αυτό, μήπως οφείλεται στην αδυναμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διαπιστώσαμε ότι όταν εμένεται η κρίση δεν ε, εκπλήρωσε τα καθήκοντά της. Το άρθρο 126 προσφέρει πολλέ δυνατότητες, όμω η Επιτροπή Μπαρόζο ήταν πάρα πολύ παθητική και περίμενε απλά να λάβουν αποφάσει οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Τώρα λοιπόν ρωτώ, μήπω είμαστε καταδικασμένοι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να έχει όλο και περισσότερε αρμοδιότητες, ενώ θα έπρεπε ίσω να ενισχύσουμε τι διαδικασίε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίω με δραστηριοποίηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Κώστα είπε αρκετά ενδιαφέροντα για το Κοινοβούλιο. Δεν κατάλαβα όμω καλά γιατί το άρθρο 225 που προβλέπει το έμεσο δικαίωμα ανάληψη πρωτοβουλειών, γιατί λέτε εσείς ότι εμείς δεν κάνουμε χρήση αυτού του δικαιώματος. Ε, κοιτάξτε, εδώ πράγματι ίσως πρέπει να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο, κυρίως όταν πρόκειται για θέματα πολιτών που τα καταλαβαίνει η κοινή γνώμη, που πρέπει να αναλάβουμε την πρωτοβουλία και όχι να περιμένουμε μέχρι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ολοκληρώσει τον γύρο των διαπραγματεύσεων και επιτέλους να έρχεται σε εμά με μία πρόταση. Απ' την άλλη, κάνατε μία παρατήρηση που πράγματι ευσταθεί. Δηλαδή, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ορισμένοι εργάζονται, πάρα πολύ, πρέπει να εργάζονται αλλά δεν το πράττουν και εργάζονται όλο και λιγότεροι. Τι εννοώ, έχουμε ας πούμε το θεσμό του εισηγητή και ο εισηγητής είναι ένα πρόσωπο με εξουσία. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε το κατά πόσον αυτό θα διαιωνίζεται ή όχι. Διότι στην περίπτωση αυτή του εισηγητή ή της εισηγήτριας μιλάμε για πολιτική εξουσία αυτό δεν ισχύει βέβαια στα Εθνικά Κοινοβούλια. Εκεί η εξουσία κατανέμεται περισσότερο στις ομάδες εργασίες ε, των κομμάτων, στα ίδια τα κόμματα. Πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε λοιπόν λιγάκι το θέμα του συγητή. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει να προτείνει κάτι συγκεκριμένο. Η κυρία Σπινέλη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, μάλλον τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσε εισηγήσει. Θα μιλήσω στα γαλλικά, γιατί μιλώ γαλλικά, βασικά στον κύριο, απευθύνομαι στον κύριο Μπερτοντσίνη. Όσον αφορά το κεντρικό χαρακτήρα των κρατών μελών, και για το γεγονός ότι δεν μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις εκτός αυτών. Διερωτώ με μήπως εδώ κάτι το εικονικό υπάρχει εδώ, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που βλέπω από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό και από το Συμβούλιο, είναι ακριβώς ο κεντρικός χαρακτήρας ορισμένων κρατών και η περιφερειοποίηση άλλων κρατών. Οπότε η επιστροφή στην διακυβερνητισμό στην ουσία είναι επιστροφή στην ε, εξουσία των ε, ισχυροτέρων εντός της Ένωσης. Αυτό είναι ο κίνδυνος και δεν είναι τυχαίο που δεν μιλάμε για διακυβέρνηση της κρίσης, αλλά για governance, που δεν είναι κυβέρνηση, είναι διακυβέρνηση. Τώρα, όσον αφορά το επικεφαλής των εκλογικών ε, καταλόγων και του συνασπισμούς, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ε, ο κύριος ε, Μπερτοντσίνη για το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοαλιτσιόν Φερχάντουλεγκ στην ίδια την πολιτική Τη Ένωση. Και αυτό που θα ήθελα να ακούσω από τους ομιλητές είναι πώς ε, βλέπετε εσείς αυτή την διαπραγμάτευση ανάμεσα στα θεσμικά όργανα, εάν είναι ανάμεσα στις κυβερνήσεις ή αν είναι ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. Ε, Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τη γνώμη σας από αυτού και όσον αφορά την σύγχυση που επικρατεί ανάμεσα στο καθόλου Ευρώπη και στο υπερβολικά πολύ Ευρώπη. Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε με θεσμικές συμφωνίες, διοργανικές συμφωνίες, αλλά ποιος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για αυτό σε μεγάλο βαθμό θα έπρεπε αυτή η πρωτοβουλία να ληφθεί από το Κοινοβούλιο το ίδιο. Αλλά θα έπρεπε να υπάρχει και μια συμφωνία, μιλάμε για τριμερή διάλογο, αλλά αυτό είναι κάπως παράξενο. Ε, ο διάλογος γίνεται και ανάμεσα στους τρεις. Ο ε, ε, Η λέξη διάλογος ετοιμολογικά δεν προέρχεται από τη συνομιλία μεταξύ δύο, όταν ε, δεν μπορούμε να λέμε τρίλογος, πρέπει να είναι ε, πολυμερής ή πολύπλευρος διάλογος. Ή τριμερής ή τετραμερής. Μπορούμε να καλέσουμε και τους πολίτες στο διάλογο. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Κώστα, για την πολιτική συμφωνία που βασιλεύει εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι κάτι πολύ ισχυρό στην Ολομέλεια και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε, ότι μέσα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές υπάρχει όντως ε, πλουραλισμός, ακούγονται πολλές φωνές, ενώ στην Ολομέλεια υπάρχει ένα ε, συμπαγές ε, πλειοψηφικό μπλοκ και διερωτώ με τελικά κατά πόσο όντως υπάρχει πλουραλισμός μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και πώς εκφράζονται οι Ευρωπαίοι πολίτες και πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση που πολλές φορές είναι, μας φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Ευχαριστώ. Μπάρμπαρα, η κυρία Μπρέσο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να επανέλθω στο θέμα των δύο ομιλητών που μίλησαν ε, για τον πιο πολιτικό ρόλο της Κομισιόν και για τη σχέση πιο, της πιο πολιτικής αυτής Κομισιόν και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αλλά κυρίως του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την άλλη, γιατί βρισκόμαστε στην αρχή μιας περίπλοκης εξέλιξης που μάλλον θα οδηγήσει σε νέο καθορισμό ρόλων, σε αναπροσδιορισμό ρόλων και σχέσεων. Να δούμε όντως πώς αυτές οι πολιτικές συμφωνίες σε κάποιο βαθμό οδηγούν στην αξιολόγηση των, ε, των υποψηφίων που έπρεπε να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση για πολιτική στήριξη της Κομισιόν. Αντίθετα, κατά τη γνώμη μου ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον το ε, αποτέλεσμα γιατί ο πρόεδρος της Επιτροπής μέσω των επιστολών για, σχετικά με τις αποστολές που ανέθεσε στους επιτρόπους θύμισε ε, ποια είναι, ποιος είναι η πηγή της δημοκρατικής ε, αλλαγής. Και θα πρέπει να το ξαναδούμε σε λίγο καιρό για να δούμε πώς αυτός ο πολιτικός ρόλος της Κομισιόν που έχει πολιτική στήριξη ε, θα, θα εξελιχθεί. Αν δούμε όμως τα ομοσπονδιακά συστήματα στην Ευρώπη, βλέπουμε για παράδειγμα ε, ε, είναι, συστήματα συνενετικά, νοσιακά. Γίνονται δηλαδή ευρείες, συμμαχίε συμμαχίες και συνασπισμοί. Πρόκειται όμως ε, είναι για πολιτικές που μέχρι στιγμές, ε, ε, στιγμής έχουν βρει την στήριξη της Κομισιόν γιατί και η νομοθετική εργασία μπορεί να αλλάξει. Κάποιοι από εσά ότι, κάποιος από εσάς είπε ότι θα μπορούσαμε να φανταστούμε μια προεπαλήθευση από πλευρά της Κομισιόν με τους εκπροσώπους κάποιας πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο. Αυτό έχει ήδη γίνει με το Συμβούλιο και επίσης με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είναι το πιο σημαντικό ε, είναι λιγότερο αληθινό για το Κοινοβούλιο, θα μπορούσε όμως να είναι αληθινό και να αλλάξει ε, ίσως τις ε, σχέσεις ισχύω. Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιστεύω ότι στις μελλοντικές, στους μελλοντικούς και σε αναλύσεις που θα κάνουμε θα πρέπει να διευκρινίσουμε καλύτερα το ρόλο του. Αν πρόκειται δηλαδή για συλλογική προεδρία, όπως συχνά το λέμε, θα πρέπει να περιορίζεται ο ρόλος αυτός στη χάραξη των βασικών πολιτικών γραμμών. Εάν όμως θέλει να αναλάβει και νομοθετικό ρόλο, τότε αυτό σημαίνει αλλαγή των συνθηκών. Και ε, περιορισμό των ψήφων, γιατί από χτες ε, οι διαδικασίες ψηφοφορίας έχουν αλλάξει στο Συμβούλιο με πιο ισχυρό ρόλο για την πλειοψηφία. Από τη Λισαβόνα και μετά είχαν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι ομοφωνία, είναι διαφορετική η συνθήκη. Επ' αυτού θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας λοιπόν. Πιστεύω πως ε, ο Σπίτσεν Καντιντά έχει αλλάξει τις σχέσεις μεταξύ Κομισιόν και Κοινοβουλίου με θετικές πτυχές αλλά και κάποια από εσάς το τόνισαν και με αρνητικές πτυχές. Είναι προφανές αυτό ισχύει για όλους όσους στηρίζουν μια κυβέρνηση. Υπάρχει μια απώλεια αυτονομίας από πλευράς των κοινοβουλίων όταν εκπροσωπώνται ομάδες που στηρίζουν το κοινοβούλιο. Και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει, να δούμε αν τελικά είναι αυτό πλεονέκτημα για το κοινοβούλιο. Πιστεύω πως για την πολιτικοποίηση της Ευρώπης και άρα για να είναι πιο προφανής ε, η ε, πολιτική συζήτηση δεν είμαι βεβαία ο αν τελικά δεν έχει συνέπεια τον περιορισμό της ελευθερίας του Κοινοβουλίου να φτάσει σε προτάσεις και να μπορεί να τις συζητήσει όλες. Ε, ε, μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα και θα ήθελα να δω τι εσείς μας προτείνετε αν θεωρείτε πως είναι αυτό περιοριστικό τελικά. Χωρίς όμως αυτό, πώς μπορούμε να φανταστούμε να μην υπάρχει γραφειοκρατική Ευρώπη και να υπάρχει ε, πολιτική Ευρώπη. Σημαίνει αυτό μεγαλύτερε ευθύνε για το Κοινοβούλιο και για τι πολιτικέ δυνάμει που θα πρέπει να φροντίσουν να βρουν συμφωνίε μεταξύ του. Και σε αυτή την περίπτωση θα περιοριστεί και η εξουσία του Συμβουλίου, γιατί τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις αντιπροσωπεύουμε στις χώρες μας και μπορούν αυτές οι πολιτικές δυνάμεις να εργαστούν και στο Συμβούλιο. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Υπάρχει και μια εργασία πριν το Συμβούλιο. Ο Πάουλο Ράντζο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ε, κοιτάξτε, τις ε, παρεμβάσεις σας ε, τις βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και υπήρξαν και κάποια καινούργια στοιχεία για να τα σκεφτούμε και εμείς στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Όμως, θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας σε δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα, Πιστεύω ότι οι τρεις παρεμβάσεις ε, είναι πολύ χρήσιμες ε, με την εξής έννοια ότι έχουν μία διοικητική προσέγγιση και όχι τόσο ευρωκρατική. Δηλαδή η δική σας η ερμηνεία των ε, κοινοτικών θεσμών θα έλεγα ότι είναι η κλασική και είναι τόσο διοικητικής φύσεως όσο και πολιτικής. Παραδείγματος χάρη, συμφωνώ με τον κύριο Κώστα που ανέφερε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο στο Κοινοβούλιο να υπάρχουν διαδικασίες ολοκλήρωσης. Γιατί αυτό ακριβώς είναι η κινητήρια δύναμη της, ε, του ομοσπονδιακού κινήματος ε, σε όλες του τις εκφάνσεις και η σημαντικότερη ε, διαφορά ήταν η διαφορά όπου είχαμε αφενός τις δυνάμεις υπέρ και αφετέρου αυτές που αντίστανται. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια διοικητική προσέγγιση αρκετά πολιτική που νομίζω ότι είναι και πολύ χρήσιμη. Όμως εκείνο που λείπει κατά την άποψή μου, είναι μια συνταγματική προσέγγιση. Αυτή λείπει και στις τρεις ε, παρεμβάσεις. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε το τι είδους ε, πολιτικό σύστημα έχουμε τώρα. Έχουμε προεδρικό κοινοβουλευτικό ή ημιπροεδρικό. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μάλλον ημιπροεδρικό με την εξής έννοια, ότι έχουμε νομοθετικό φορέα με δύο ε, επίπεδα, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και κατόπιν υπάρχει ο εκτελεστικός φορέας, το εκτελεστικό όργανο, που είναι πολύ συγκεκριμένο, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά όμως έχουμε και ένα συλλογικό όργανο που είναι ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που δεν έχει νομοθετικές αρμοδιότητες, αλλά έχει αυτές τις αρμοδιότητες ε, που οι Ιταλοί θα χαρακτήριζαν ως ε, αρμοδιότητες προς πολιτική κατεύθυνση ή με πολιτικό πρόσταγμα. Έχουμε λοιπόν ένα σύσταγμα, ένα σύνταγμα με την εξής έννοια. Όπως και στη Γαλλία Είχαμε το βέλτιστο παράδειγμα του Γκολ και του Μιτεράν που ε, μας έδωσε ένα παράδειγμα που μπορούμε να μιμηθούμε. Αυτό λοιπόν που θα μπορούσε να μας βοηθήσει για να ερμηνεύσουμε τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζουμε και για να ξέρουμε ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναλάβουμε, είναι ότι πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση, συνταγματικής φύσεως. Γιατί πάρα πολύ συχνά ακούει κανείς τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι αναφέρονται σε αυτές τις ιδιαίτερα περίπλοκες θέσεις ανάμεσα στους θεσμούς. Όμως δεν μας δίνει ένα μοντέλο, ένα μοντέλο με μια σφαιρική πρόπτικη. Αυτό είναι εκείνο που λείπει για μένα. Δηλαδή τελικά τι είδους μοντέλο υπάρχει. Παραδείγματος χάρη θα μπορούσε το όλο θέμα να ξαστεί κάτω από διαφορετική προοπτική, διαφορετική από αυτήν που υπάρχει εδώ. Όμως υπάρχουν και πολλές ομοιότητες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Βρετανική πολιτική ιστορία. Έχουμε θεσμούς που παίζουν συνταγματικό ρόλο χωρίς όμως να υπάρχει κράτος. Αυτό ισχύει τώρα, αλλά αν πάει κανείς να ανατρέξει στη Βρετανία του 18ου και 19ου αιώνα, υπήρχε κοινοβούλιο, υπήρχαν δικαστήρια, αλλά δεν υπήρχε το κράτος όπως υπήρχε στη Γαλλία, στην Προσία ή στα κράτη της Ευρωπαϊκής Επίρου που τότε βέβαια ακόμα δεν ήταν δημοκρατίες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με θεσμούς που βρίσκονται σε ένταση, συγκρούονται μεταξύ τους, χωρίς όμως να υπάρχει πίσω από αυτούς ένα κράτος. Υπάρχει πρόφαση, η πρόφαση των ε, θεσμών. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση είναι πραγματικά συνταγματική, που όμως ε, δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει. Αυτή είναι μία παρατήρηση δική μου πρέπει να φύγω σε καμιά ώρα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ακούσω τις απαντήσεις, έτσι απλά ήθελα μόνο να σας προβοκάρω. Ευχαριστούμε πολύ Παόλο και εγώ έχω μια ερώτηση πολύ σύντομη την εξή. Δηλαδή όλοι μας εδώ κατανοούμε τις υποχρώσεις μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, πώς πρέπει να την τροφοδοτήσουμε, να την ενισχύσουμε, αλλά μία ερώτηση προς τον κύριο Κάστα. Ε, είμαστε αποτελεσματικοί ή αναποτελεσματικοί. Ο σκύτερη είναι προς το Συμβούλιο. Ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ε, δημιουργήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρακτική Δεν ξέρω αν εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να επανέλθει το πρώτο Γενικό Συμβούλιο που είχε συσταθεί να είναι πραγματικά διαφανές και έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί πολύ πιο εύκολα να συνεργαστεί με αυτό. Αυτά όσον αφορά στις ερωτήσεις μας. Βλέπετε ότι εμείς ε, είμαστε επιθαρχημένοι. Ε, μπορούμε να μιλήσουμε ε, και μέσα σε ένα λεπτό. Δεν έχετε πολύ χρόνο για να απαντήσετε, αλλά ε, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε μπορείτε να τοποθετηθείτε. Δεν ξέρω ποιο θέλει να ξεκινήσει. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω εγώ. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι δύσκολο να απαντήσουμε σε τόσο λίγο χρόνο, αλλά για να είμαι σαφής και συγκεκριμένος θα ξεκινήσω από ε, μία παρασύρηση του Τομάζο Παρασκιώπα, το οποίο, η οποία προέκυψε από τα όσα μας είπε η κυρία Σπινέλη, ο οποίος έλεγε ότι αν εξετάσουμε τα θεσμικά και συνταγματικά πολιτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θελήσουμε να εφαρμόσουμε και το πλεονέκτημα της δημοκρατίας, θα πρέπει σίγουρα να τα βλέπουμε από την άποψη του Δήμου, των πολιτών, αλλά και από την άποψη του κράτους, της δημοκρατίας. Η δημοκρατία, και το η δημοκρατία είναι Δήμος και κράτος. Και όπως βλέπουμε ότι στο πρώτο θέμα, στο Δήμο, όσον αφορά τους πολίτες, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πιο σαφή, πιο διάφανα, πιο κατανοητά, αλλά εξακολουθούν να είναι περίπλοκα. Ε, ο Δήμος ε, είναι κάτι μακρινό, κάτι ε, απομακρυσμένο και για παράδειγμα τα πάντα γίνονται για έναν, ένα κόμμα, ένα θεσμό σε σχέση με τη Γαλλία ας πούμε, αλλά δεν μπορεί να κυβερνήσει μόνος του γίνονται ακριβώ γι' αυτό. Και αυτό φυσικά εκφύσεω θα είναι περίπλοκο. Σε χώρε όπω στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση σε εξουσίες. Υπάρχει ένα άνθρωπο, ένα θεσμό και αυτό συγκεντρώνει τι περισσότερε εξουσίε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να είναι πιο σαφή τα πράγματα. Υπάρχει η διαδικασία του candidate, η οποία αναφέρθηκε. Και ουσιαστικά δίνουμε πρόσωπο ε, σε αυτές τις ε, διαχωριστικές γραμμές. Οι διαχωριστικές γραμμές υπάρχουν και πρέπει ε, απλώς να τις φέρουμε στην επιφάνεια. Υπάρχει, για παράδειγμα, το ΕΛΚ, το οποίο κατέβηκε στις εκλογές και υπέβαλε τον τάδε υποψήφιο. Τις επόμενες ευρωεκλογές θα είναι πιο σαφή τα πράγματα. Αυτή τη φορά δεν είχαν καταλάβει όλα, την επόμενη θα διευκρινιστούν περισσότερο. Και αν πούμε ότι ο τάδε ε, έχει την εξουσία να ε, καθορίσει και την ομάδα του. Αυτός λοιπόν που είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει μόνο δικαίωμα να απολύσει έναν επίτροπο, αλλά μπορεί και να τον ορίσει ποιος θα είναι. Αναφέρομαι λοιπόν στο άρθρο 17.7. Ο κύριο Σόπφλη μα είπε ότι από πλευρά κρατών μελών ίσω δεν είναι ικανοποιητικό να υπάρχει αυτή η εξουσία στα χέρια κάποιου άλλου, αλλά υπάρχει μια εγγύηση. Του προσφέρουμε έναν επίτροπο. Τώρα βρίσκεται αυτό σε συνθήκε. Αν ο κύριο Γιούνκερ ήταν σε θέση να επιλέξει αυτό μόνο του, σίγουρα θα το είχε κάνει σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί να βγάλει από το καπέλο του τον κύριο Τάβε, ε, που δεν θα ήθελε η Μέρκελ για τη Γερμανία ή που δεν θα ήθελε ο Λάντ ε, για τη χώρα του, α πούμε. Αλλά σίγουρα θα γίνει με μεγαλύτερη αυτονομία και θα είναι σαφές ότι θα είναι αυτός και επομένως οι πολίτες με την ψήφο του που περνούν στη διαδικασία έγκρισης ε, κάποιου. Και αυτό να το πω και παρεπιπτόντως στον κύριο Σόπφλιν, ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να διευκρινίσουμε σε ποια χώρα το γεγονός ότι υπάρχει ένας επίτροπος ανακράτος μέλος πλέον είναι πρόβλημα, να σας πω για τη χώρα μου, τη Γαλλία. Ε, πραγματικά θεωρήθηκε ότι ε, ε, είναι ε, έλλειψη ισορροπίας το να υπάρχει ένας Γάλλος επίτροπος και τρεις από τις χώρες της Βαλτικής, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι τμήμα αυτής της αδυναμίας, το οποίο όμως εξισορροπείται αν υπάρχει πάντα ένας επίτροπος ανά ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά χώρα και ε, ε, μπορεί ίσως να επιλέξει λίγο καλύτερα, ίσως θα έχουμε καλύτερους καρπούς από ό,τι τώρα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της υποκότητας. Υπάρχουν συγκεκριμένε ε, πολιτικές δυνάμεις, υπάρχουν διτές αναφορές έστω ότι υπάρχει μια ψηφοφορία, ποιος θα πρέπει να αποφασίσει από εκεί και πέρα το πρόγραμμα δράσης. Ε, τα κράτη-μέλη, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, παραδείγματο χάρη αυτό που κάνει πολιτικές δυνάμεις μετά τις εκλογές ε, στη Γερμανία, κάνουν ένα πολύ σημαντικό έργο για να ετοιμάσουν τις προγραμματικές τους δηλώσεις. Και εδώ θα πρέπει να γίνει σε θεσμικό επίπεδο. Υπάρχει χρόνος μεταξύ των ευρωεκλογών και της ανάληψης των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτός ο χρόνος επιτρέπει να γίνονται αυτοί οι διάλογοι, αλλά πάντα με το βλέμμα στις διαχωριστικές γραμμές. Παραδείγματο χάρη να ξέρουν οι πολίτες ότι υπάρχουν οι τάδε πολιτικές ευαισθησίε, υπάρχουν αυτές οι θεσμικές ε, ευαισθησίε και αυτές οι πολιτικές ευαισθησίε. Και με αυτό ολοκληρώνω. Ε, ο Λιβιέ Κωστά δικαίω είπε ότι θα πρέπει να τονίσουμε και τι γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Επιτροπές. Γιατί εκεί σε μια λογική αντιπαράθεσης διαπραγμάτευσης ε, υπάρχει και αυτή η κομματική πτυχή η οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί από εκεί και πέρα για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό και να εγκρίνουμε αποφάσεις. Ε, δεύτερον, πολύ σύντομα να απαντήσω για το κράτος, για την εξουσία. Αυτό είναι εξίσου σημαντικά και πολύ συχνά το ξεχνούμε. Σας είπα προηγουμένως ότι οι Βρυξέλλες ε, είναι σαν τη Washington για τους πολίτες. Είναι πολύ μακριά. Ε, οι πολίτες θα ήθελαν ε, οι Βρυξέλλες να δρουν προς όφελος τη ζωή τους. Δεν ξέρω αν οι Αμερικανοί θα ήθελαν η Washington να δρά προς όφελος της δικής τους της ζωής. Αλλά υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε εξουσίες ε, για το κράτος και πρέπει να δούμε πολύ καλά πώς γίνεται. Και εδώ να απαντήσω στην κυρία Περές για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο διακύβευμα. Ε, φεύγουμε από μια θητεία την οποία έχει στιγματίσει η Τρόικα. Η ε, Τρόικα είναι ένα ε, ουσιαστικά Διεθνές Νομισματικό Ταμείο της Ευρώπης. Η Τρόικα είναι ένα θεσμός που δημιουργείται με τις χώρες που ζητούν βοήθεια. Ναι, υπήρξαν οικονομικά προβλήματα, κάποια στιγμή έχουν ανάγκη βοήθειας και επομένως η λογική Τρόικας κρατών μελών είναι μια ε, λογική ερεσιμότητας. Ε, ε, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανακάνει. προέκυψε ως ανάγκη, αλλά αυτό δημιούργησε ένα τελείως διαφορετικό πνεύμα. Η Τρόικα είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο της Ευρώπης. Και υπάρχει και το θέμα της ε, μεταρρύθμισης της διακυβέρνηση τη Οικονομικής και νομισματική Ένωση. Εγώ σας είπα ότι η Τρόικα είναι η, Ευρώπη, ε, ε, η Ευρωπαϊκή ε, το Ευρωπαϊκό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και επίσης υπάρχει και το Σύμφωνο Σταθερότητας. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να υπερβούν κάποια όρια. Αυτή είναι η έννοια της ε, Νομισματικής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη έχουν κυριαρχία, αλλά αν περάσει στην άλλη πλευρά είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και αυτό είναι το Σύμφωνο Σταθερότητας. Θέτει όρια. Αυτό είναι και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Και αυτό θέτει όρια. Ε, υπάρχει το όριο του 3% του ελλείμματος. Και πέραν των ορίων, ε, εντός μάλλον των ορίων, τα κράτη-μέλη είναι κυρίαρχα, αλλά εκτός ορίων εκεί αρχίζουν οι αλλαγέ. και θα πρέπει να διευκρινιστεί αυτό, διότι δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την ονομοποίηση. Και επίσης η Ευρώπη ε, είναι η Ευρώπη οσά. Υπάρχουν... Ε, ε, ε, οι διαφορές ορισμένες φορές θεωρούν ότι είναι τα ίδια πράγματα, αλλά δεν είναι αλλά πρόκειται για συστάσεις. Συστάσεις δεν σημαίνει διαταγές και αυτό θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές και από πλευράς πραγματικών εξουσιών του κράτους και υπάρχει και μια Ευρώπη φυσικά την οποία θα πρέπει να υπερασπιστούμε είναι η Ευρώπη Παγκόσμια Τράπεζα. Επειδή πληρώνει μπορεί να έχει ένα ρόλο ε, για να δώσει χρηματοοικονομικά τουλάχιστον κίνητρα. Ε, Αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά για να υπάρχουν και ε, διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις και ενισχύσεις. Και σας λέω ότι υπάρχουν δύο ε, χώρες οι οποίες έφυγαν από το Ιμάν, μνημόνιο, κάποιες άλλες προσπαθούν να φύγουν. Αλλά το θέμα είναι να αντιληφθούμε και ποιο είναι το πνεύμα των πολιτών. Και επίσης θα πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ σαφής για τη φύση των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υποκορικές ε, εξουσίες οι οποίες ε, είναι πολύ σημαντικές, το λένε και οι συνθήκες σε κάποιους τομείς, για παράδειγμα οι Αλίες και οι Γεωργοί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η ζωή τους ρυθμίζεται από τις Βρυξέλλες, από το Στρασβούργο. Αλλά κάποιοι άλλοι Ευρωπαίοι θεωρούν και έχουν δίκιο ότι δεν γίνονται τα πάντα εδώ, αλλά σε εθνικό επίπεδο πρώτα, στη χώρα τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το υπενθυμίσουμε, ιδίω σε περίοδου που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Διότι αν θεωρούμε ναι, ότι όλα απορρέουν από τι Βρυξέλλε και τα πράγματα δεν πάνε καλά, τότε φταίνουν οι Βρυξέλλε. Θα πρέπει όμω εμεί να τα δούμε λίγο πιο διεξοδικά και ναι μεν έχουν οι Βρυξέλλες εξουσίες αλλά δεν έχουν όλε τι εξουσίε. Ε, υπάρχουν για παράδειγμα το, το περίφημο παράγωγο των κλοβών των πουλιών. Η ε, κλοβή ε, είναι θέμα κανονισμού, είναι επιτροπολογία. Θα πρέπει λοιπόν να το δεχτούμε ότι αυτό προέκυψε από επιτροπολογία και επαναλαμβάνω ότι οι κανόνες ε, δε μήνυμης δεν είναι κάτι ε, το οποίο θα έπρεπε να απασχολούν τους, Ευρωπαίους, ε, τους Ευρωβουλευτές. Αν ήταν εθνικοί βουλευτές θα ασχολούνταν ίσως με αυτό. Υπάρχουν κάποιες γενικές γραμμές, κάποιες κατευθύνσεις και από εκεί και πέρα υπάρχουν εθνικοί κανονισμοί οι οποίοι ακόμα και αν υπάρχουν πολιτικές προκλήσεις θα αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτά λοιπόν από πλευρά μου. Ευχαριστώ. Um, okay, um, I, I started on the, I think, uh... Θα τοποθετηθώ σε πολλές από τις ε, ερωτήσεις. Ε, θέλω να διευκρινίσω λιγάκι την έννοια της συνένεσης. Ε, την έτσι λιγάκι και ο κύριος Σόφλιν. Πράγματι υπάρχει πρόκληση και αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της εξ αρχής. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση γίνεται μια ε, πρόκληση σε καθημερινή βάση και αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει με το νομοθετικό τομέα, όπου βλέπουμε να υπάρχει διεκδίκηση της ε, συνένεσης σε συγκεκριμένες ε, χρονικές στιγμές και συνταγματικής φύσεως. Αν δούμε όμως λιγάκι το θέμα της οικονομικής ε, διακυβέρνησης, εκεί η συνένεση είναι μία μόνιμη πρόκληση. Και θα ήθελα να προσθέσω και το εξή. Υπάρχει το θέμα της αυτονομίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου ως θεσμοί. Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση αυτή. Υπάρχουν μελέτες για τη γραμματεία του Συμβουλίου. Εγώ όμως θεωρώ ότι όσον αφορά το θέμα της ανεξαρτησίας και κυρίως ανεξαρτησίας των κρατών μελών, δεν βλέπω να υπάρχει καμία σημαντική ένδειξη, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει ε, ένας ολόκληρος διοικητικός μηχανισμός και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές σημαντικές επιτροπές ε, όπως ε, η Eurogroup, η Ανώτατη Επιτροπή της ΚΠΑ που αποτελούνται από εκπροσώπους των κρατών μελών. Επεκτείνεται λοιπόν η γραφειοκρατική δομή αλλά με κάποιο πολύ περίεργο τρόπο. Πολλές άλλες ερωτήσεις αφορούσαν τη σύγκρουση αυτών των δύο μοντέλων, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο κύριος Γιου Λάινεν αναφέρθηκε ε, στις ε, τροποποιήσεις ε, που έχουν λάβει χώρα μετά από παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και αναφέρθηκε επίσης και το θέμα του κοινοβουλευτισμού. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό και έχει οργανωθεί γύρω από τον αυταρχικό τρόπο λήψη αποφάσεων που όμως δεν αφορά στο Συμβούλιο. Εγώ θα ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός ε, στο να κάνουμε κάποιες προβλέψεις για το μέλλον. Βεβαίως ε, και περιμένω το Κοινοβούλιο να διεκδικήσει τις εξουσίες του, να επιμείνει στο ότι θέλει και εκείνο να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όπως ε, συμβαίνει ήδη στο νομοθετικό τομέα και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό να το διεκδικήσει το Κοινοβούλιο. Νομίζω όμως ότι το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή ευνοεί περισσότερο το ότι οι κυβερνήσεις ε, θα είναι αποκεντρωμένος και ε, το πραγματικό κέντρο βάρους ε, τα θέματα εξωτερικών υποθέσεων και στα δημοσιονομικά, εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιορισμένες αρμοδιότητες. Πολύ σωστά αναφέρθηκε το θέμα της συνταγματικής διάστασης. Αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι υπάρχει κάποια ρευστότητα. Η συνθήκη της Λισαβόνας προσπάθησε να διορθώσει λιγάκι το όλο θέμα, αλλά είναι και πολύ δύσκολο να του δοθεί μια τελική μορφή, γιατί υπάρχει και μια λογική ένταση έμφυτη στο σύστημα. Οι εθνικές κυβερνήσεις ε, προφανώς ε, και θέλουν στο θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης να υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία. Το ίδιο ισχύει και για την εξωτερική πολιτική. Αν δούμε την Επιτροπή Μπαρόζο και τη νέα Επιτροπή, παρότι αυτή τη στιγμή προβαίνω προφανώς σε παραδοχές, αυτό που βλέπουμε μετά τη Λισαβόνα, βλέπουμε να υπάρχει αποδυνάμωση της Επιτροπής. Η Επιτροπή παίζει και έπαιξε βέβαια κατά διάρκεια της κρίσης σημαντικό ρόλο, αλλά όχι πολιτικό. Εγώ λοιπόν πρέπει να πω θα με ξέπλητε πάρα πολύ αν ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής που νομίζω ότι είναι ο μακροβιότερος ε, στο Συμβούλιο και ήταν και πρόεδρος της Eurogroup. Ίσως αλλάξει την κατάσταση δραματικά, ριζικά, κυρίως σε επίπεδο κρατών μελών. Πάντως ε, βλέπω περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίζει σημαντικό ρόλο. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις ανάμεσα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Αυτό θα μας αποσχολήσει εμάς τους ε, ερευνητέ. Το θέμα της προσωποποίησης των συμφωνιών δεν νομίζω ότι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα αναλάβει το ρόλο που πρέπει. Ίσως το αναγκάσει κανείς, άτυπα όμως. Γιατί είναι απαραίτητο οι κυβερνήσεις ε, των κρατών μελών να βρουν ένα χώρο όπου θα έχουν την ανταλλαγή απόψεων. Υπάρχουν και άλλα ομόσπονδα συστήματα όπως το καναδικό. Εκεί υπάρχουν οι προνομίες, οι τυπικές του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου. Υπάρχουν όμως και κάποιες φαίες Δεν ξέρω αν μπορεί να λυθεί το συνταγματικό θέμα. Πάντως είναι και κάτι το οποίο λύνεται περισσότερο μέσα από την πρακτική εφαρμογή και όχι τόσο μέσα από επίσημες ε, συμφωνίες και αλλαγές συνθήκων. Σας ευχαριστώ πολλά ενδιαφέροντα ερωτήματα και θα προσπαθήσω εν συντομία να ε, επανέλθω όσον αφορά τις διαφορές στο Κοινοβούλιο έχουμε τις υπέρ και τους κατά της Ευρώπης όσον αφορά το θέσμο ε, την ε, ομοσπονδιοποίηση και μετά έχουμε κοινωνικές αποκλήσεις αλλά και αποκλήσει για τον προπολογισμό, το κοινό θα πρέπει να αρχίσει να το καταλαβάνει. Δεν είναι ένα στοιχείο το οποίο διαταράζει την εικόνα του Ευρωκοινοβουλίου τόσο. Τώρα, όσον αφορά τους τριμερείς ε, διαλόγους, κυρία Μπερέζη, δεν θέλησα να ε, κατηγορήσω το Κοινοβούλιο. Είναι θεμητό να ανησυχούμε για τη σωστή λειτουργία και να μην μπλοκάρονται τα πάντα συνέχεια και να ανησυχούμε και περισσότερο για την έλλειψη διαφάνεια από από το Συμβούλιο και όχι από το Κοινοβούλιο Κοινοβούλιο τόσο. Δεν είναι τόσο ικανοποιητικό αυτό το στοιχείο από δημοκρατική άποψη και άρα το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει στρατηγικέ διακρίσει και διαχωρισμού στα κείμενα που πρέπει να περάσουν πρώτη ανάγνωση και εκείνα που πρέπει πραγματικά να αναλυθούν ε, μέσω συζητήσεων στην Ολομέλεια από το Κοινοβούλιο. Ε, τώρα, η έκπληξη των θεσμικών εξελίξεων των τελευταίων ετών είναι κάτι που κανένας δεν το περίμενε. Το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να αντιμετωπίσει μια τελείως νέα ε, ε, αρχιτεκτονική, θεσμική και ίσως το Ευρωκοινοβούλιο κατά κάποιο τρόπο έχει μείνει και έχει ξεχάσει ότι το 80 ε, κατέκτησε νομοθετικές εξουσίες απορρίπτοντας τον προϋπολογισμό στην αρχή της συναπόφασης επίσης απέρριψε κείμενα για να καταδείξει ότι δεν συμφωνούσε με τη στάση του Κοινοβουλίου. Ένα σωρό τρόπους έχει το Κοινοβούλιο να θέσει βέτο και έχει και δυνατότητα να πάρει το λόγο κάθε φορά και κάποιες στιγμές θα πρέπει ίσως να, να, να τα στυλώσει και να αποφασίσει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Τώρα, θα πρέπει και πάλι ε, και για, για όλα τα θέματα να δημιουργηθούν σχέσεις ε, ε, εξουσίας και δυνάμεων. Εφόσον υπάρχουν κείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στι ανησυχίε τη κοινωνία των πολιτών, ο πρόεδρο του Κοινοβουλίου έχει να παίξει σημαντικό ρόλο εδώ. Να χρησιμοποιήσει τι ομιλίε που κάνει στο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τι διμερεί επαφέ με τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση, ώστε να εστιάσει την προσοχή σε κάποιε πρωτοβουλίε οι οποίε θεωρούνται πολύ σημαντικέ. Και πιστεύω κυρίω ότι το Ευρωκοινοβούλιο δεν πρέπει να αφαιθεί να ξεπεραστεί από τι πρωτοβουλίε των πολιτών, γιατί αυτό θα ήταν ε, και εις βάρος της αντιπροσωπευτικότητάς του κατά κάποιο τρόπο. Για το θέμα των συμμαχιών υπάρχει κάτι που είναι ενδιαφέρον. Το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές έχουν αυτή την ε, συμφνήθεια να συνεργάζονται εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά δεν έχουμε μπει σε μια νέα διαδικασία στις σχέσεις με την Κομισιόν. Και ένα σημείο το οποίο δεν αναφέρθηκε και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχει συμφωνία ΕΛΚ ε, σοσιαλιστών στο διαθεσμικό επίπεδο απλά και μόνο για το γεγονός ότι ο πρόεδρος Σούλτς επανεκλέγει πρόεδρος. Είναι πρώτη φορά που μιλάμε για ε, υπερθεσμικά, δηλαδή εσείς θα πάρετε το Κομισιόν και εμείς το Κοινοβούλιο. Και η παράδοση ήταν να μην επανεκλέγεται ποτέ κανένα ένας πρόεδρος στην ίδια ε, θέση. Υπάρχει λοιπόν εδώ πολιτική συμφωνία σε επίπεδο ε, θεσμών τώρα πρέπει να μείνουμε σε αυτό το πνεύμα και αν δεν λειτουργήσει το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει πάλι να θυμώσει και να κάνει την Κομισιόν να καταλάβει ότι δεν πάει έτσι, ε, δηλαδή η σύγκρουση ε, φέρνει αποτελέσματα. Έχει επιτρέψει το Κοινοβούλιο να έχει περισσότερε εξουσίε, να αυξήσει τον έλεγχο στην Επιτροπή και στο Ευρωκοινοβούλιο. Επίση να δείξει ότι η πολιτική μπορεί να λειτουργήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Κοινοβούλιο ε, το, το 95 ας πούμε για τι πυρηνικέ δοκιμέ, για την οδηγία Μπόλκενστάιν, για την απόρριψη διαφόρων άλλων κειμένων. Αυτό τονίζει την διαφορετικότητα, τη διαφορά του Ευρωκοινοβουλίου και, και χαλάει την εικόνα του γραφειοκριτικού ε, θεσμού. Τώρα, Όλα όσα έχουν γίνει από το 2009 λόγω κρίσης θα πρέπει να γραφτούν ε, ε, και τα όσα έγιναν με τον πρόεδρο Γιούνκερ γιατί διαφορετικά θα ξεχαστούν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ε, δεν θα πρέπει να μείνουν μόνο σε θεσμικό επίπεδο. Εάν η ενιαία πράξη λειτουργήσει είναι επειδή υπήρχε σύνδεση ανάμεσα στο θεσμικό και στο ε, πολιτικό σκέλος. Και εδώ θα πρέπει να, εάν υπάρξει νέα μεταρρύθμιση θεσμική, θα πρέπει να ξεκίσουμε ότι αυτά όλα δεν είναι μόνο για να χαρούν οι ευρωβουλευτές, αλλά για να είναι, νομιμοποιηθούν θεσμοθετηθούν οι νέες αρμοδιότητες. Τώρα, τι είναι ένα αποτελεσματικό Ευρωκοινοβούλιο, δεν ξέρω, είναι ένα... Ε, ε, ένα θέμα που δεν πρέπει να το κρίνουμε σε σχέση με τη ρουτίνα ε, ε, και ε, δεν είναι η Κορεπέρ ούτε οι νομικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιες για να λένε στο Ευρωκοινοβούλιο ποιο είναι η αποτελεσματική λειτουργία. Ε, να βρίσκω πως το Ευρωκοινοβούλιο έχει κάνει πολύ τον καλό απέναντι στη Κομισιόν και το Συμβούλιο προς το συμφέρον της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσει και άλλα μέσα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολλά. Ε, πολύ θα ταράξετε τους ε, όσους μας ακούνε στο διαδικτύο. Πολλά, πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα τα όσα μας είπατε. Φυσικά μπορείτε να μείνετε μαζί μας όσο μπορείτε και περνάμε αμέσως στο επόμενο πάνελ differentiation of the European... Που αφορά την ε, διαθεσμική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νίπετ, Βέρσελς, αυτός ο Γερμανός, κολονία ή όχι. I am ah, sorry. Ε, Madam Chairperson, life, world is difficult and complicated. Ο κύριος Βέρσελ από το Πανεπιστήμιο. Κυρία Πρόεδρε, η ζωή είναι δύσκολη. Και θα ήθελα να σας πάω δύο βήματα μπροστά και να σας αναφέρω το έργο ενός λαμπρού ε, φοιτητή διδακτορικού μου που του πήρε ένα χρόνο να τα ετοιμάσει όλα αυτά. Βλέπετε εδώ στη διαφάνεια και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα κατανοήσουμε αυτό. Εγώ έχω μία προσέγγιση 3α. Μια ανάλυση για να δούμε λίγο πώς έχει κατάσταση, πώς είναι οι τάσεις ε, στην ε, ε, εποχή αυτή. Θα κάνω μια αξιολόγηση και από εκεί και πέρα θα σας δώσω κάποιες συμβουλές. Και πρέπει να σας πω ότι αντιθέτως ε, με τα όσα πιστεύουμε, όπου εμείς οι ακαδημαϊκοί συνήθως δίνουμε καλές συμβουλές, θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα μετριοπαθείς ως πανεπιστημιακοί, γιατί έχουμε όρια στα στιγμή αυτά. Σε κάποια άλλα όχι, αλλά εδώ νομίζω ότι εκκρεμούν πάρα πολλά ερωτήματα, στα οποία πραγματικά δεν μπορούμε να σας δώσουμε εμείς την καλύτερη συμβουλή, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια στο σημείο αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε με την ανάλυση. Έχουμε συνεχώς ε, πολυπλοκότητα λόγω μεγάλης διαφοροποίησης πολλών ε, θεμάτων και πολλών ε, χωρών. Εδώ βλέπετε ποια χώρα βρίσκεται σε ποια σύνθεση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφοροποίηση. Έχουμε κάποιες χώρες που είναι εντός, κάποιες άλλες που είναι εκτός και αν προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε την όλη διαδικασία, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο περίπλοκα. Διότι ε, κάθε μία από αυτές τις δομές έχει διαφορετικές διαδικασίες, διαφορετικές νομικές βάσεις, διαφορετικούς συμμετέχοντες, ε, διαφορετικές εξουσίες για τα εθνικά κοινοβούλια και επομένω είναι πολύ περίπλοκη κατάσταση. Αν δούμε την εξέλιξη, εδώ έχουμε το έργο κάποιων άλλων συναδέλφων που σαν τις διαδικασίες και τις ε, δράσεις και βλέπουμε ότι ορισμένα πράγματα έχουν αυξηθεί και έχουμε διαφοροποιημένη ολοκλήρωση. Το ερώτημά μου είναι γιατί γίνεται αυτό. Η μία παρατήρηση είναι ότι ε, κάποια κράτη-μέλη δεν βρήκαν αρκετές δυνατότητες να χρησιμοποιήσουν τις υφιστάμενες θεσμικές δομές και συνταγματικές δομές και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε ως σημείο κίνησης υπάρχουν κάποια νομικά και συνταγματικά όρια, αλλά μπορεί να υπάρχουν και ε, πολιτικοί φραγμοί. Ε, Παραδείγματο χάρη, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο μπλοκάρει μια υπόθεση, για παράδειγμα. Υπάρχουν και διάφορα τέτοια στοιχεία στο παρελθόν και σε κάποιο βαθμό μπορούμε να εξηγήσουμε αυτή τη διαφοροποίηση. Επίσης, να πω ότι αυτό το οποίο αναφέρεται στη συνθήκη του Άμστερνταμ για την ενισχυμένη συνεργασία είναι κατά την άποψή μου μια ανελαστική μορφή για ευελιξία. Διότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι πελωτικοί περιορισμοί και υπάρχουν πολύ λίγα περιορισμένες δυνατότητες. Επομένως ε, έχει χρησιμοποιηθεί δύο φορές μόνο και η τρίτη ακόμα συζητάται και εκεί θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί. Επομένως η ενισχυμένη συνεργασία μέχρι τούδε δεν έχει αποτελέσει την πεπατημένη που θα προσέφερε επαρκείς ευκαιρίες να τη χρησιμοποιήσουμε και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με κάποιες μονοχώρες και όχι με όλες. Και τώρα να περάσω στην αξιολόγηση. One point is, uh, Το ένα θέμα είναι ότι σχετίζεται με την ανάλυση. Είχε κρύο σήμερα το πρωί στο σταθμό στην Κολονία, που είχε και απεργίες και έκατσα πολλή ώρα στο σταθμό, κρύωσα. Να, εδώ με βοηθάνε λίγο οι φίλοι μου, μου φέρανε λίγο νεράκι. Σας ευχαριστώ. Analysis and assessment. In the analysis... Ανάλυση και πάμε στην αξιολόγηση. Στην αξιολόγηση νομίζω ότι υπάρχει κάτι βασικό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι ότι θα λειτουργούσαν αυτά μόνο αν ήταν μόνο γαλλογερμανική συνεργασία μέχρι τώρα. Το θέμα είναι κατά πόσο θα ξαναπροκύψει το θέμα αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Μέχρι ποιου σημείου μπορούν να συνεργαστούν οι δύο αυτές χώρες και να βρουν και επαρκή υποστήριξη από άλλες χώρες. Γιατί όπως είπα εδώ είναι ικανή αλλά όχι επαρκή συνθήκη αυτό και τα επόμενα χρόνια θα πάει τελείως διαφορετικά, διότι δεν φαίνεται κατά πάσα πιθανότητα ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες πρωτοβουλίες από τις δύο αυτές χώρες μαζί. Τώρα, αξιολόγηση έγινε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο, μια δήλωση και μου, αν μου επιτρέπετε, ε, ε, διατυπώσατε και ένα δόγμα για τη διαφοροποίηση. Υπάρχουν κάποιες σαφείς δηλώσεις, δεν είναι αρνητικό αυτό, όπου λέτε ότι η συμμετοχή ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσδίδει αυξημένη νομιμοποίηση σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και δεν υπάρχει καμία ε, αμφισβήτηση της ε, δυνατότητας διαφοροποίησης από, για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και νομίζω ότι υπάρχουν δύο στοιχεία εδώ σε αυτό το δέγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά υπάρχει και η διάσημη ρίση ε, της Αμερικανικής Επανάστασης που είπαν ε, ότι δεν υπάρχει ε, δυνατότητα κειμένου χωρίς εκπροσώπηση, ε, χωρίς φόρος μάλλον χωρίς εκπροσώπηση. Νομίζω ότι εμείς έχουμε πολλές περιπτώσεις στις οποίες είναι τελείως αντίθετη κατάσταση. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγεστε διότι είστε αιρετοί ε, στις, εθνικούς, στις εθνικές λίστες. Τα μέλη λοιπόν που δεν τους αφορά αυτό το μέτρο ε, θα πρέπει να έχουν ευρωβουλευτές που έχουν άποψη επί του ζητήματος.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 ε, κάτι και θα αλλάξει αν επιβάλλεται ψηφοφορία για θέματα τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, στη Φιλανδία και στη Γερμανία τα μέλη της Πολωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου κλπ. θα πρέπει να ψηφίζουν κάτι το οποίο δεν επηρεάζει τους πελεονούς ε, και δεν αφορά τους δικού μας ψηφοφόρους. Θα μπορούσε να γίνει πολύ μακρά συζήτηση από αυτό. Το θέμα όμως δεν είναι ποιο έχει δίκιο και ποιο έχει άδικο, αλλά το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει κοινή γνώμη από αυτού. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ πολύ σημαντικό εδώ και εδώ τίθεται και το θέμα ε, και είμαστε και πάλι στην αξιολόγηση των σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια διότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να μπορέσουμε να περιορίσουμε λίγο τα προβλήματα της νομιμοποίησης αν μπορούσε να υπάρχει συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια από αυτού. Κάτι το οποίο αναφέρετε και εσείς στο δόγμα σας ε, ε, είναι ότι μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση ε, σε κάποιες εσωτερικές διαδικασίες. Παραδείγματο χάρη κάποιες ειδικέ επιτροπές, κάποιες υποεπιτροπές όπου μόνο τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις ενδιαφερόμενες χώρες θα μπορούσαν να συμμετέχουν. Νομίζω ότι πρέπει να σας πω ότι έξωθεν αυτό το ανταλαμβάνονται ως κάτι καλοπιστικού χαρακτήρα. Το θέμα είναι ποιος λαμβάνει αποφάσεις εν τέλει. Μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα η δομή και η διαφορετική σύνθεση, αλλά δεν ενδιαφέρει το, τη δημόσια συζήτηση το θέμα αυτό. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να βρούμε είναι διαφοροποιημένες στρατηγικές κατά την άποψή μου. Και νομίζω ότι είναι αδύνατο να προβλέψουμε για τα επόμενα πέντε χρόνια ποιε θα είναι οι προκλήσεις της διαφοροποίησης. Νομίζω ότι μία θα είναι ε, μεγαλύτερη διαφοροποίηση στον τομέα της νομισματικής Ένωση. Τη της του προπολογισμού της Ευρωζώνης. Έχουμε ήδη δει κάτι στην Τραπεζική Ένωση, όπου το Κοινοβούλιο ήθελε περισσότερες εξουσίες ε, για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και επομένως θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις εκεί. Επίσης κάτι άλλο σημαντικό μπορεί να είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και τη ιδέα ενός ε, από τους πρώην ευρωβουλευτές ε, του Άντριου Νταφ να έχουμε ε, σχέση σύνδεσης ουσιαστικά και νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσπαθήσει να παρακολουθήσει τη συζήτηση και να προετοιμαστεί για τις πιθανές εξελίξεις. Ακόμα και συνταγματικές αλλαγές. νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα θα συζητήσετε αν μπορεί να γίνουν αλλαγές στη συνθήκη. Αν οι αλλαγές στη συνθήκη είναι και αυτές το θεματολόγιο μας, το θέμα είναι πώς θα μπορέσει να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ίσως και σε κάποιο βαθμό να προωθήσει και να συναποφασίσει με, για μορφές διαφοροποίησης με συνδεδεμένα μέλη. Και νομίζω ότι η Επιτροπή σας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη να κάνει κάποια πράγματα, ακόμα και αν δεν προκύψει το θέμα στη συζήτηση για τα επόμενα ένα-δύο χρόνια. Το να είστε προετοιμασμένοι θα είναι εξίσου σημαντικό. Επίσης, κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να δείτε και μορφές εσωτερικής διαφοροποίηση. Εδώ νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάποια προετοιμασία και δεν νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για τον έξω κόσμο και τις συνέπειες της δημόσιας συζήτησης. Τώρα, συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια, εδώ πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να το επανεξετάσετε το θέμα αυτό. Ε, υπήρχε, για παράδειγμα, η όλη συζήτηση για το άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου και κατά πόσον αυτή είναι η σωστή άκουσα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το δείτε κι εσείς. Εγώ ε, μπορώ να το δω μόνο ως εθνική αντίδραση. Κανείς δεν ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει αυτό το άρθρο 13. δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ετοιμάσουν και κανονισμό. Αν δείτε το πρωτόκολλο ε, ε, της ε, Λισαβόνας για την Πρόζακ, ε, ε, Εκεί λέγεται ότι εκπρόσωποι των κοινοβουλίων δεν μπορούν να λάβουν ε, καμία δεσμευτική απόφαση. Αυτές οι μικτές επιτροπές λοιπόν σαφέστατα έχουν πολύ περιορισμένη επιρροή στη διαδικασία απόφασης. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να το ε, εξετάσετε περαιτέρω. Δεν θα πρέπει να το λησμονήσετε για κάποιες συγκεκριμένες μορφές διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να περιμένετε και το αναπάντεχο μπορεί, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, για παράδειγμα στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο, πριν από πέντε χρόνια Κανείς δεν θα έλεγε να έλεγε τι θα γίνει ε, ε, να εξετάσουμε το δημοσιονομικό σύμφωνο. Αν δούμε τι περιμέναμε. Ήταν κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο τότε και τελικώς ήταν αναπόφευκτο να γίνει. Είναι πολύ βέβαια ασαφής ε, σύσταση, δεν είναι σαφής και πολύ συγκεκριμένη, αλλά θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο τομέα της διαφοροποίησης θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για, τα, για τον απάντεχο. Ευχαριστώ. Και εμείς ε, ευχαριστούμε. Νομίζω ότι προσθέσατε και εσείς ερωτήσεις σε ήδη ένα μακροσκελέστατο ε, κατάλογο ερωτήσεων που υπάρχουν ήδη. Η επόμενη ομιλήτρια από το Πανεπιστήμιο του Μάστρες. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Η κυρία Μόνικα Κλάες. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, μου ζήτησαν ή μου ζητήσατε να παρουσιάσω κι εγώ ε, κάποια άλλα στοιχεία στην εικόνα που περιπλέκουν περαιτέρω το θέμα της, ε, του συντάγματος, του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Πρόκειται για τα εθνικά συντάγματα, συνταγματικές τάξεις, αν θέλετε, με μεγαλύτερη ακρίβεια. Θα προσπαθήσω λοιπόν καταρχήν να ορίσω τις τάσεις που υπάρχουν σε αυτό τον τομέα, μετά θα δω λιγάκι τις ε, προκλήσεις και κατόπιν θα προσπαθήσω να καταθέσω και εγώ προτάσεις για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Όσον αφορά λοιπόν τα εθνικά συντάγματα και τις εθνικές ε, συνταγματικές τάξεις, αυτές είναι ένα καθοριστικό τμήμα της ευρύτερης ε, συνταγματικής υποδομής. Αν βέβαια μπορούμε να μιλήσουμε για ένα ευρωπαϊκό συνταγμα. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε. Αυτό είναι ένα, ένα σύνθετο συνταγματικό πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή στοιχεία. Άρα δηλαδή, επειδή έχουμε αυτά τα ε, εθνικά και τα ευρωπαϊκά στοιχεία που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, η συνταγματική αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διαδραματίζεται την ίδια στιγμή σε διάφορα επίπεδα σε διαφορετικούς χώρους που είναι αλληλεξάρτητοι μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν ε, τα εθνικά συντάγματα μπορούν να αντιμετωπιστούν ως κρίκοι στον ε, ενωσιακό μηχανισμό και δεν πρέπει να γνωρούνται. Η σημασία των εθνικών συνταγμάτων για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθοριστική σημασίας, αλλά παράλληλα τα εθνικά συντάγματα δεν ε, είναι απόλυτα ανεξάρτητα με την έννοια ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι πλέον απόλυτα ελεύθερα στο να υιοθετήσουν όποιο σύνταγμα τους αρέσει, ακόμα και αν τα εθνικά συντάγματα αποτελούν την κύρια ε, έκφραση κυριαρχικών εξελίξεων σε μια χώρα. Υπάρχουν προϋποθέσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όσον αφορά τη συνταγματική τάξη που πρέπει να τηρείται στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν οι θεμελιώδεις αξίες του συνταγματισμού. Εγώ θα αναφερθώ στη σχέση ανάμεσα στα εθνικά συντάγματα και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εδώ υπάρχουν υπέρ και κατά. Τα το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι τα εθνικά συντάγματα επιβάλλουν κάποιες προϋποθέσεις στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Και υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίσματος. Το θέμα ότι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια η Ένωση επιβάλλει προϋποθέσεις στα εθνικά συντάγματα. Και στους δύο τομείς διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν αρκετές προκλήσεις. Το πρώτο λοιπόν, ε, βλέποντας τη μία πλευρά του νομίσματος, τα εθνικά συντάγματα, τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ας δούμε το ρόλο των εθνικών συνταγμάτων και συνταγματικής τάξης στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πρώτον, διευκολύνουν την ολοκλήρωση, την καθιστούν δυνατή, να μπορεί ένα κράτος μέλος να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Από την άλλη όμως περιορίζουν και τη δυνατότητα συμμετοχής στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Σε ορισμένε ε, χώρες μάλιστα αυτά αποτελούνται, αντιμετωπίζονται ως προπύργια στην όλη εξέλιξη ε, αντίδρασης προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αν θέλετε, θεματοφύλακες των ε, εθνικών συνταγμάτων και ως εκ τούτου και του κράτους. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι προϋποθέσεις που επιβάλλουν αυτά τα εθνικά συντάγματα. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι αυτά τα συντάγματα και οι περιορισμοί δεν αναφέρονται απαραίτητα στα συντάγματα, πρέπει κανεί να δει τις ερμηνείες των δικαστηρίων και μπορεί να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στις ε, καθημερινές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε καθημερινή βάση, ανάμεσα σε αυτό και αφετέρου στο πώς προχωράει η ολοκλήρωση υπάρχουν ε, μεγαλύτερες συνταγματικές ε, αλλαγές με την έννοια της ε, τροποποίησης της συνθήκης. Και εδώ τα εθνικά συντάγματα παίζουν ρόλο και στα δύο επίπεδα. Αν δούμε τώρα τις πρώτες αλλαγές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καθημερινή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εθνικά συντάγματα επιβάλλουν τρεις, τριών ειδών προϋποθέσεις τρεις ομάδες προϋποθέσεων που είναι και επίμαχες. Πρώτον, πρόκειται για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πολλοί θα θυμάστε ότι σήμερα αναφερόμαστε σε αυτές ε, κατά κανόνα με την αναφορά απόφαση Ζολάγκε, όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε περιορισμούς ε, στο Ευρωπαϊκό, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δηλαδή είπανε ότι δεν ισχύει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο εφόσον δεν σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σήμερα λοιπόν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι έχουμε φτάσει σε ένα είδος διευθέτησης του θέματος. Όμως εύθραυστη η διευθέτηση με την έννοια τα συνταγματικά δικαστήρια δεν ήραν ποτέ τις προϋποθέσεις και επιπρόσθετα, κατά περίεργο τρόπο, υπάρχει τώρα μια αλλαγή σε αυτή την ένταση που υπήρχε ανάμεσα στα εθνικά συστήματα προστασίας και το ευρωπαϊκό. Οι εθνικοί φορείς δεν ενδιαφέρονται πλέον για το ότι δεν υπάρχει αρκετή προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια διαφορετική μορφή προστασία σε εθνικό επίπεδο. Αν θέλετε λοιπόν υπάρχει διαφορά στι ισορροπίες. Υπάρχει βέβαια κάποιο περιθώριο για να εμφανιστούν συγκρούσεις και αντιθέσεις κυρίως διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναφέρεται σε τομείς που είναι καθοριστική σημασία για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρόκειται λοιπόν για τη νομιμοποίηση που μας ενδιαφέρει και που πάρα πολύ εύκολα μπορεί να αντικατοπτρίζεται και μέσα από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θεμελιώδη δικαιώματα, όπως επίσης και μέσα από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ένας άλλος τομέας επίμαχος είναι τα εθνικά δικαστήρια που ισχυρίστηκαν ότι μόνο μερός μπορούν να ελέγχουν κατά πόσον μία νομοθετική πράξη Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει στον τομέα αρμοδιοτήτων αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, ε, το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμένει μια ιστοριά τη, σωστό αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι τα δικαστήρια αποφασίζουν μονομερός για μία χώρα. Αυτό βέβαια είναι μόνο η επίσημη πλευρά της υπόθεσης και βεβαίως αυτή η υπόθεση έχει επηρεάσει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει μόνο μία περίπτωση ενός δικαστηρίου που έχει ε, αποφασίσει ότι δεν ισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό συνέβη στην περίπτωση των συντάξεων στην ε, Τσεχία. Μικρό βέβαια. Αυτό που ενδιαφέρει ε, είναι άλλες πιο σημαντικές υποθέσεις που εκκρεμούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τα εθνικά συνταγματικά δικαστήρια διεκδικούν την αρμοδιότητα να προστατεύουν τη συνταγματική ταυτότητα του κράτους μέλους. Τι είναι αυτό? Αυτό ποικίλει ανάλογα με το κράτος μέλος. Και όλη αυτή η έννοια του τι μπορεί να σημαίνει η συνταγματική ταυτότητα, η ερμηνεία που δίδεται είναι διαφορετική σε κάθε κράτος μέλος. Πάνω σε αυτό που ισχύει είναι ότι ένα συνταγματικό δικαστήριο θα μπορεί να αποφασίζει για ενωσιακά μέτρα τα οποία επηρεάζουν στη, την ε, συνταγματική ταυτότητα ενός κράτους και για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να εφαρμόζονται. Αυτά όσον αφορά την καθημερινή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δούμε τώρα την ε, τροποποίηση της συνθήκης, ε, τα εθνικά συντάγματα επιβάλλουν ακόμα πιο αυστηρούς περιορισμούς. Σε αυτόν τον τομέα του, της τροποποίησης της συνθήκης, αν δει την ομολογία των δικαστηρίων και συζητήσεις που γίνονται σε συνταγματικό επίπεδο, θα διαπιστώσει ότι μερικές φορές φτάνει κανείς τα όρια του, του τι είναι συνταγματικά εφικτό. Σε ορισμένες χώρες η κατανομή της εξουσίας αυτή καθε αυτή είναι προβληματική και μάλιστα τίνει να απειλεί και την κυριαρχία της εθνικής δημοκρατίας. Σε άλλες χώρες γίνεται αναφορά σε σημαντικές αξίες του συντάγματος, δηλαδή η ολοκλήρωση στην για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι κατοχυρωμένα στο σύντογμα. Εδώ ε, η αντίδραση είναι προβληματική γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στο άρθρο 2 αναγνωρίζει αυτές τις αξίες, όμως ε, η τα κράτη-μέλη δεν αναφέρονται τόσο σε αυτό όσο στην εθνική εκδοχή αυτών των δικαιωμάτων. Και βεβαίως κατόπιν υπάρχουν και ε, διάφορες άλλες προϋποθέσεις για την ε, τροποποίηση και επικύρωση συνθηκών, τα δύο τρίτα, ε, τα δημοψηφίσματα. Αυτά θα το πει ο επόμενος ομιλητής. Οι προκλήσεις λοιπόν είναι αυτές που σας παρουσίασα. Αν δούμε τώρα λιγάκι. Την άλλη πλευρά αυτής της υπόθεσης θα δούμε ότι ε, ε, ποιοι είναι οι όροι που επιβάλλουν στα εθνικά θεσμικά όργανα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, θα δούμε ότι τα συντάγματα όσον αφορά την σεβασμό στις συνταγματικές αξίες που απορρέει από την ιδιότητα του μέλους ευρύτατα ορίζονται στις συνθήκες. Θα βρίσκουμε αυτά στο άρθρο 2 των συνθήκων. Υπάρχει ε, μάλλον τη φάση της ε, ειστοχής είναι πιο αυστηρή η Ένωση υπό τα κριτήρια της Κοπενχάγης, όμως όταν μπουν τα μέλη πια ε, οι συνθήκες, οι όροι είναι ασαφείς. Άρα λοιπόν έχουμε Ε, το θέμα της υπερακολούθησης και του σεβασμού για αυτές τις βασικές αξίες. Το πρώτο πρόβλημα λοιπόν που βλέπουμε ε, είναι ότι δεν υπάρχει σαφήνεια όσον αφορά τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις των κρατών μελών. Δεν είναι σαφές το τι απαιτεί η Ένωση όσον αφορά το σεβασμό του κράτους δικαίου, για παράδειγμα. Παραμένουν όλα αυτά σαφή. Όσον αφορά την παρακολούθηση και την εποπτεία. Το σύστημα αυτό δεν είναι πάρα πολύ όριμο γιατί τα κράτη-μέλη μέχρι στιγμής δεν έχουν θελήσει ένα όριμο σύστημα παρακολούθησης και εποπτείας. εφόσον υπάρχει και περιορισμένη εντολή στον οργανισμό για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν είδαμε ότι ο πίτροπος Τίμερμανς είπε ότι θα εστιάσει ε, στην πρόληψη της απόκλησης των κρατών μελών. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο άμα δεν υπάρχουν προδιαγραφές και σύστημα εποπτείας. Και έπειτα, για το μηχανισμό επιβολής, για τη μορφή των διαδικασιών επιβολής, σύμφωνα με το TFU, τις συνθήκες, δηλαδή άρθρο 6, το οποίο σπανιότατα χρησιμοποιείται. Και πάλι είναι πολύ δύσκολο να τα χρησιμοποιήσει κανείς όλα αυτά, εάν δεν έχει, για παράδειγμα, τις προδιαγραφές με βάση τις οποίες να αποφασίσει αν υπάρχει συστημική απειλή στο κράτος δικαίου. Αν εξετάσουμε το θέμα των εθνικών ε, θεσμών που επιβάλλουν ε, ε, τα όρια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ε, το θέμα δεν είναι τόσο τι μπορεί να κάνει η Ένωση και τα θεσμικά της όργανα, γιατί δεν μπορεί να επιβάλλει στα κρατημέλη να περιορίσουν ε, οι, τους όρους και τις προϋποθέσεις που επιβάλλουν τα ίδια τους τα συντάγματα. Άρα λοιπόν αυτό που μπορεί να κάνει και πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τουλάχιστον να γνωρίζει, να συνειδητοποιήσει ότι αυτές οι συνταγματικές ε, ανησυχίες υπάρχουν σε καθένα από αυτούς τους τομείς που ανέφερα και να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των κρατών μελών των ίδιων. Για παράδειγμα, όσον αφορά την αναθεώρηση, ε, σημαίνει ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να δείξουν ότι γνωρίζουν ε, τους περιορισμούς ε, των αρμοδιοτήτων κτλ. κτλ. ανταπόκριση λοιπόν στην, στους κανόνες και από την άλλη πλευρά τι μπορεί να κάνει η Ένωση τα προβλήματα του συστήματος όσον αφορά την παρακολούθηση ε, εποπτεία και επιβολή των βασικών ε, θεμελιωδών αξιών και εκεί πρέπει πολλά ακόμα να γίνουν. Καταρχήν, όσον αφορά την αποσαφήνιση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στα κρατη άρθρο 2, τι σημαίνει ακριβώς, τι σημαίνει να είναι κανείς μέλος της Ένωσης και τι απαιτεί αυτό για τα ίδια τα κρατημέλη, να, να διευκρινιστούν αυτές οι αξίες Και ε, δεύτερον, ε, μηχανισμός παρακολούθησης ε, για να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε τον εκτροχιασμό των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Και θα ήθελα να ζητήσω από τον καθηγητή Steve Pierce τώρα να πάρει το λόγο. Προέρχεται από το Πανεπιστήμιο του Essex και ειδικεύεται στον Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Is my presentation set up, the PowerPoint version? Do I just press? Okay, excellent. Thank you very much for inviting me to this. Καλημέρα σας. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε σε αυτό το πολύ σημαντικό σεμινάριο. Για όσους μπορεί να μπουν στο πειρασμό να σκεφτούν ότι πρόκειται για κάποια σκοτεινή επιτυχία του Ευρωπαϊκού νόμου. Αν είναι, αν είναι κανείς ε, Βρετανός Ευρωβουλευτής, ίσως να είδε το πρωτοσέλιδο μιας από τις εφημερίδες μας σήμερα, της Daily Telegraph, όπου, όπου ε, παρουσιάζεται μια επιστολή 40 ακαδημαϊκών, δικαστών κτλ. να κάνει πίσω στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Είναι τμήμα μια τεράστια συζήτηση που γίνεται τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα μόνο παράδειγμα βέβαια των διαφορετικών ειδών διαφοροποίησης που έχουν αναπτυχθεί στη διάρκεια των ετών. Και ένα από τα βασικά στοιχεία χαρακτηριστικά είναι ότι δεν υπάρχει ένα είδος διαφοροποίησης, αλλά διάφορα είδη διαφοροποίησης και αλλαγή χρονικά, καθώς και ε, η χρήση των αλλαγών διαχρονικά. Ο τρόπος με τον οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί όλα αυτά και η συχνότητα το, της χρήσης τους. Έχουμε εδώ ένα γράφημα όπου δείχνει την αλλαγή διαχρονικά σε διάφορες ε, διατάξεις που αναφέρονταν σε διαφοροποιημένη ολοκλήρωση. Δεν έχω προετοιμάσει το γράφημα αυτό, αλλά πιστεύω πως θα ήταν ενδιαφέρον να το συγκρίνουμε αυτό με ένα διαφορετικό ε, γράφημα που θα υπολόγιζε την χρήση της διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης, τη χρησιμότητα μάλλον, γιατί αυτό το γράφημα όταν άρχισε να ισχύει η συνθήκη του Μάστριχτ, ε, είχε προβλεφθεί. Αλλά οι διατάξει του Μάστριχτ είναι η διαφοροποιημένη ολοκλήρωση. Ενώ τα όσα υπόθηκαν αργότερα, η Νομισματική Ένωση ναι, δεν ε, ξεκίνησε παρά μόνο το 1999, το κοινωνικό πρωτόκολλο δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ στη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Αν σε φτιάξει κανείς ένα γράφημα της χρησιμότητας της διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης, λοιπόν, θα δει πως υπάρχει μια μικρή ε, αύξηση τη δεκαετία των 90, μεγάλωμα το 99 όταν άρχισε η Νομισματική Ένωση, μετά ομαλή αύξηση στη διάρκεια των επόμενων ετών και μια μεγάλη αύξηση πάλι από το 2011. 10 ε, με συγχωρείτε. Αυτό είναι το κλειδί, μάλλον μια από τις τάσεις κλειδί στην διαφοροποιημένη ολοκλήρωση. Αυξάνεται διαχρονικά, αλλά το ποσοστό χρήσης του χρήσιμου αυξάνεται, επιταχύνεται και επιταχύνεται κυρίως στα έτη ανάμεσα στο 2010 μέχρι 2014. Και ποιος ξέρει αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός. Σίγουρα αυτή είναι η κατάσταση μέχρι σήμερα. Αν δούμε λοιπόν τις λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας, έχουμε τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, παρουσίασε δύο βασικά είδη διαφοροποιημένη ολοκλήρωσης, κοινωνικό πρωτόκολλο και νομισματική ένωση. Και αν δείτε την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία των τελών της δεκαετία του 90 όταν υπογράφηκε η συνθήκη του Άμστερνταμ, φαινόταν ότι θα ήταν μια μικρή και σύντομη απόκληση προς την διαφοροποιημένη ολοκλήρωση. Ε, μέχρι το 1999, όπου στη συνθήκη του Άμστερνταμ το κοινωνικό πρωτόκολλο περίφθη, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλεία ε, το Ηνωμένο Βασιλείο έμεινε εκτός ε, από τα έξι μέτρα ε, στα διάρκεια των έξι ετών που ίσχυε. Μετά τελικά τώρα ε, ε, ε, υπήρχε μία ψευδής ρήτρα sunset που ποιος ξέρει τώρα μέχρι πότε θα εξελιχθεί γιατί έκτοτε μόνο εξελίσσεται. Τώρα με την Νομισματική Ένωση δεν είχαμε μόνο δύο δυνητικά μόνιμα opt-out, η Νοβένο Βασίλειο και η Δανία, αλλά και μια ενσωματωμένη δυνατότητα στα ορισμένα κρατημέλη να προχωρήσουν χωρίς τα υπόλοιπα. Αν και όλα τα κρατημέλη απεφάσισαν ότι αυτοί οι δυο ε, βασικά ήταν ε, υποχρεωμένοι να συμμετέχουν. Άρα λοιπόν έχουμε το συνδυασμό δύο διαφορετικών βασικών μοντέλων διαφοροποίησης. Το μοντέλο όπου κανείς τρέχει να προλάβει, δηλαδή κάποιοι έχουν προχωρήσει και οι υπόλοιποι τρέχουν να προλάβουν αργότερα, όπως έκανε η Ελλάδα και άλλοι ε, για την νομισματική ένωση, αλλά έχουμε και το δυνητικά μόνιμο opt-out, δηλαδή την μη συμμετοχή, όπως για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Δανία. Και αυτές οι δύο κατηγορίες κάπως έχουν ε, ε, συγχωνευτεί γιατί και η Σουηδία φαίνεται να μην ε, θέλει να συμμετέχει και δεν το υποχρεώνεται κιόλα. Λοιπόν, τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν ενταχθεί το 2004. Εκ τότε δεν έχουν ενταχθεί τρία. Από τα δέκα που εντάχθηκαν το 4, οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες ε, δεν έχουν ε, ενταχθεί με την οικονομική έννοια. Τρεις λοιπόν ε, στους δέκα είναι πάντα περισσότερο από το 30% των οικονομιών των δέκα κρατών μελών που προσεχώρησαν. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε να υποτυπούμε την πρακτική σημασία της μη συμμετοχής στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Όσον αφορά τώρα το τη διαφοροποίηση, το κατά πόσο χρησιμοποιεί κανείς το νέο νόμισμα ως μόνο του μοναδικό νόμισμα ή όχι, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση περιλαμβάνει και διαφορετικούς κανόνες σε σχέση με το τι ισχύει για την οικονομική διακυβέρνηση. Τα κράτη της Ευρωζώνης και αυτά που είναι εκτός βρίσκονται σε σχετικά διαφορετική θέση. Το χάσμα έχει ενταθεί με την πάροδο του χρόνου, όμως αρχικά ήταν μικρή η διαφορά. Ας πούμε, δεν προβλέπονται κυρώσεις στα μικρά τιμέλη της Ευρωζώνης εάν υπερβούν τον κανόνα περί υπερβολικού ελλείμματος. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, όχι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν ε, σαφώς ε, την υποχρέωση βέβαια να μην ε, προβαίνουν σε υπερβολικό έλλειμμα. Δυστυχώς βέβαια το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή έχει τεράστιο έλλειμμα. Ακόμα και παρότι αυτός ο διαχωρισμός κάπως ε, ε, θόλωσε στην πράξη, υπήρξαν ε, κυρώσεις σε περίπτωση υπερβολικού ελλείμματος όμως ήταν πολιτικά δύνατο να εφαρμοστούν αυτές οι κυρώσεις. Και υπήρξαν πάρα πολλές ανησυχίες μετά από αυτό. Το αποτέλεσμα, το, το χάσμα λοιπόν ανάμεσα στα κράτη και τα μη κράτη της Ευρωζώνης δεν ήταν τόσο μεγάλο όσον αφορά την ε, ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, όπως θα μπορούσε να είναι με βάση αυτά που είχα προβλεφθεί στη συνθήκη. Μετά ακολούθησε η συνθήκη του Άμστερνταμ το 1999 μόλις είχε αρχίσει να εφαρμόζεται η ΟΝΕ. Και έτσι εντάχθηκαν δύο νέα στοιχεία διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το ένα αφορά την ε, δικαιοσύνη και τις ιστορικές υποθέσεις και το άλλο αφορά την ενισχυμένη συνεργασία που το τελευταίο κατά την περίοδο της συνθήκης ε, του Άμστερνταμ ε, δεν ήταν τόσο μεγάλης και καθοριστικής σημασίας γιατί τα κράτη-μέλη επέμειναν σε τόσες πολλές ε, ασφαλιστικές δικλείδες ουσιαστικές και πιο λιγότερο ουσιαστικές που ήταν αδύνατο να εφαρμοστούν όλα αυτά. Και έτσι λοιπόν ορισμένα κράτη-μέλη έκαναν κάποιες συζητήσεις ε, για ας πούμε ένα είδος ευρωπαϊκής εταιρείας. Τότε βέβαια αυτό κρίθηκε ανέφικτο και ε, η Ισπανία κατέθεσε βέτο ή το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αν θέλετε. Αυτό ε, εγκρίθηκε και υπογράφηκε από ορισμένα κράτη-μέλη. Στην πράξη τώρα, το πιο σημαντικό τουλάχιστον για 10 ολόκληρο χρόνια ήταν το opting out ε, σε θέματα δικαιοσύνης και ιστορικών υποθέσεων. Παρότι υπήρχαν δύο μορφές opting out αυτοεξαίρεσης σε αυτά τα θέματα. Η διαφοροποίηση έλαβε διαφορετικές μορφές ανάλογα και με το θέμα. Η πρώτη μορφή στην πούμε είναι το Schengen. Ήδη υπήρχε διαφοροποίηση εκτός της ε, νομικής τάξης ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σέγγεν υπογράφηκε, υπογράφηκε το 90, εφαρμόστηκε το 95 και εκεί τότε η συνθήκη του Άμστερνταμ είχε ενταχθεί στη νομική τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε γίνει μια μορφή διαφοροποίησης μέσα στο ίδιο το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχαν λοιπόν διάφορα στοιχεία του Σέγγεν, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία και πάλι έχουν μόνιμο opt-out η Δανία εφαρμόζει τους κανόνες σε μεγάλο βαθμό, αλλά έχει μια διαφορετική μορφή opting out και για τα νέα κρατημέλη έχουμε μια διαδικασία του να προλάβουν να ε, καλύψουν το κενό. Τα νέα κρατημέλη καλούνται καταρχήν να εφαρμόζουν τη συνθήκη Schengen αλλά και αυτό εφόσον υπάρχει ομοφωνία από πλευράς μελών του Schengen. Ε, ορισμένα κράτη μπήκανε λοιπόν στη συνθήκη του Σέγκεν, αλλά πάλι όχι. Υπήρξαν κάποια πολιτική φύσεως προβλήματα με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία που δεν τις ενέκριναν για να μπουν ε, στη ζώνη του Σέγκεν. Αυτό είναι το πρώτο opting out. Υπάρχει και το δεύτερο opting out σε θέματα δικαιοσύνης και ιστορικών υποθέσεων που απορρέει από τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Αυτό είναι opting out για Ηνωμένο Βασίλειο και την Δανία όσον αφορά τα μέτρα μη Σέγγεν, μετανάστευση, άσυλο και αστικό δίκαιο. Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχουν άλλη δυνατότητα να κάνουν opting in, να συμμετέχουν δηλαδή στα μέτρα που επιθυμούν. Αλλά η Δανία δεν μπορεί, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, το opting in. Στην πρακτική, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία μέχρι το 2009 άσκησαν αυτό το δικαίωμά τους ε, του opting in σε θέματα αστικού δικαίου ε, και ε, ασύλου, αλλά όχι τόσο για θέματα μετανάστευσης. Η συνθήκη της Νίκαιας άλλαξε λίγο τα πράγματα. Εκεί δόθηκε ιδιαίτερη σημασία σε, ενισχυμένους, σε κανόνες ενισχυμένης συνεργασίας. Και υπήρξε εξή παραδοχή, ότι πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή λόγω τη εντωμεταξύ εκκρεμούσα διεύρυνση. Ε, τότε, αυτό ήταν το, γενικότερα το θέμα που απασχολούσε τη συνθήκη της Νίκαια, που είχε ως στόχο τη διεύρυνση. Ε, έτσι λοιπόν ήρθε το θέμα της ε, έκτακτης ανάγκης. Αυτό ήταν και το πιο σημαντικό που παρεμπόδιζε την ενισχυμένη συνεργασία. Αυτά δεν εφαρμόστηκαν μέχρι τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η Μπαρόσο 1, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη δεν διαφέρθηκαν τόσο πολύ, ακόμα και μετά τη διεύνηση στο να εφαρμόσουν αυτή τη συνθήκη, μέχρι που ήρθε η συνθήκη της Λισαβόνας. Έτσι λοιπόν η συνθήκη της Λισαβόνας είναι το Big Bang, αυτή η μεγάλη έκρηξη που διευκόλυνε τη σημαντική αύξηση χρήσης της διαφοροποίησης μέσα στην ευρωπαϊκή νομική τάξη. Άλλαξε και τις τρεις βασικές μορφές. Ε, πρώτον, ε, κανόνες διαφοροποίησης στην πράξη όπως και σε ιστορικές υποθέσεις, η Νομισματική Ένωση προάγει τη συνεργασία. Τα τελευταία πέντε χρόνια βλέπουμε μεγαλύτερη διαφοροποίηση εκτός του ενωσιακού νομικού πλαισίου, αλλά σε σχέση με αυτό. Κατά το παρελθόν το ΣΕΝΚΕΝ ε, δεν ήταν συνδεδεμένο. Είχαμε το λόμπινγκ, τους ε, ελέγχους ε, στα σύνορα, την ανταλλαγή αστυνομικών πληροφοριών. Έτσι λοιπόν Όλα αυτά συνέδικαν με το νοσιακό δίκαιο, αλλά δεν υπήρξαν ουσιαστικοί ε, θεσμικοί δεσμοί. Δεν είχαμε δηλαδή αυτές τις διεθνείς συνθήκες ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η συμφωνία του Σέγκεν είχε άμεση σχέση με το ενωσιακό δίκαιο και αυτό λοιπόν βιώνουμε από τη συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία η ίδια συνθήκη δεν τοποθετείτε σε αυτά, αλλά ζούμε τι συνέβη τα τελευταία πέντε χρόνια. Και θα σας τα εξηγήσω περισσότερα αργότερα. Περισσότερο αργότερα. Ας δούμε το νέο άρθρο 136 της ιδρυτικής Συνθήκης που επιτρέπει μέτρα οικονομικής διακυβέρνησης μόνο για την Ευρωζώνη. Το 6-pack και το 2-pack ισχύουν μόνο στην Ευρωζώνη. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε περισσότερο τη χρήση της διαφοροποίησης σε σχέση με την οικονομική διακυβέρνηση. Όπως σας είπα υπάρχουν και συνθήκες εκτός της ένομης τάξης ε, ή της νομοθετικής μάλλον τάξης. Έχουμε σύμφωνα σταθερότητας. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Έχουμε ένα, μια συνθήκη για το Ταμείο διάσωσης που αυτό όμως δεν έχει ακόμα θεσπιστεί αλλά πρόκειται για οικονομική ε, υποστήριξη, ε, για διάσωση οικονομική τραπεζών και άλλων. Αυτό έχει άμεση σχέση με την νομική τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα σημαντικό στοιχείο αυτών των συνθήκων είναι ότι ε, καταργείται πλέον η ομοφωνία και επιπλέον με τι έννοια. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ομοφωνία στα 28 κράτη-μέλη για τα περισσότερα, για όλα. Δεν χρειάζεται ομοφωνία στα κράτη της Ευρωζώνης. Δεν είναι απαραίτητη πλέον η ομοφωνία. Έχουμε απλουστευμένους ε, κανόνες, βεβαίως άλλους κανόνες για την ενισχυμένη συνεργασία, όμως έχουμε τις ίδιες βασικές αρχές. Και μόνο τα κράτη βέβαια που επικυρώνουν τη συνθήκη δεσμεύονται και από αυτήν. Άρα εδώ αυτό μοιάζει με τη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο ποιος θέλει μπορεί να συμμετέχει στην ενισχυμένη συνεργασία. Επίσης, κάτι που είναι δύσκολο να το περιγράψει κανείς, αλλά είδαμε πέρυσι την ανάπτυξη ε, ενωσιακών μέτρων που αφορούν σε όλα τα κράτη-μέλη. Ενωσιακή νομοθεσία που ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη, όμως κατ' ουσίαν μέτρα αφορούν μόνο την Ευρωζώνη. Ας πούμε τα μέτρα για τη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση. Αν δούμε τη νομοθεσία για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τραπεζική Εποπτεία, προβλέπονται διατάξεις που δεν κάνουν διαφοροποίηση ανάμεσα σε κράτη Ευρωζώνης και μη. Αν δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση, η Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να εποπτεύει τα κράτη εκτός Ευρωζώνης. Πάντως η διατύπωση της συνθήκης και η συγκεκριμένη νομική βάση λένε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτοεξαίρεσης, opting out, η ευρωπαϊκή νομοθεσία σημαίνει όμως ότι οι αποφάσεις δεν ισχύουν για όλα τα κρατημέλη. Τώρα, στο Ταμείο Διάσωσης, βεβαίως ε, οι διατάξεις ισχύουν για όλα τα κράτη, αλλά στην πρακτική αποφασίστηκε ότι μόνο τα κράτη που συμμετέχουν στην Ευρωζώνη και άλλα που το επιθυμούν δίνονται να συμμετέχουν και να εφαρμόζουν την νομοθεσία περί ε, Ταμείου Διάσωσης. Αυτό θα μπορούσε να διεδοθεί περαιτέρω. Παρότι υπάρχουν και κάποιες επιφυλάξεις αν επεκταθεί πέρα από τον τομέα της νομισματικής ένωσης, ε, αν θα υπάρχει σαφή διαφοροποίηση ανάμεσα ε, σε Ευρωζώνη και εκτός Ευρωζώνης κράτη για θέματα ε, τραπεζικά. Πάμε τώρα στις ιστορικές υποθέσεις, στη δικαιοσύνη. Ε, το δικαίωμα του Ηνωμένου Βασιλείου, το opting out, επεκτάθηκε και το χρησιμοποίησε μάλιστα το Ηνωμένο Βασίλειο περισσότερο από ό,τι συνήθιζε. Στην πρώτη φάση, κατά κύριο λόγο, εξαιρέθηκαν ε, από τη δεύτερη φάση από την ε, νοσιακή νομοθεσία. Ας δούμε λιγάκι την, ε, το ποινικό, την ποινική νομοθεσία. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εξαιρεθεί ε, σε πάρα πολλά μέτρα, ποινικά μέτρα. Βέβαια επανήλθε σε 35 εξ αυτών και υπάρχουν άλλες τρεις λεπτομέρειες για να εξετάσει κανείς τις λεπτομέρειες. Ας πούμε, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Αυτό είναι κάτι το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο και νομίζω το έχω ήδη αναφέρει σε αντίθεση με τη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την νομολογία και το ποινικό δίκαιο. Υπάρχει ένα παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά ε, είναι αντίθετα με το ρεύμα που είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Στην ενισχυμένη ε, συνεργασία και πάλι άλλαξαν οι κανόνες, η πολιτική βούληση εφαρμόζεται στην πράξη ο φόρος ε, συναλλαγματικών συναλλαγών δεν εφαρμόζεται και κάποιες ε, περιπτώσεις ε, τις νομολογίες που έχει προκύψει, ούτε και αυτές ισχύουν. Παρότι υπάρχουν πολλές συζητήσεις σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία, οι περισσότερες συζητήσεις βασίζονται στην παραδοχή ότι πρέπει να υπάρξει διεύνηση, διότι τα νέα κράτη-μέλη δεν μπορούν να εφαρμόσουν τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην πρακτική δεν υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στο ρόλο των παλαιών και των νέων κρατών. Βλέπετε λοιπόν ότι ένα παλαιό ή τα παλαιά κράτη που είχαν θυμώσει για τα μέτρα ενισχυμένη συνεργασία... η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ άλλων είχαν μάλιστα απευθυνθεί μέχρι και ε, το δικαστήριο ε, στα θέματα διαζυγίων ας πούμε εκεί συμμετείχαν και παλιά και νέα κρατημέλη ε, στον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και εκεί βλέπουμε ότι είχε προταθεί να συμμετέχουν και παλιά και νέα κρατημέλη όμως η διαφοροποίηση αποδείχθηκε μία δυνατότητα για να λυθούν άλλες διαφορές. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει προβεί σε ευρύτατη προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή της ενισχυμένης συνεργασίας. Λέει ότι ο νομοθέτης, ο Ευρωπαίος, μπορεί να προχωρήσει εφόσον το επιθυμεί. Και υπάρχει και άλλη μία συνθήκη ανάμεσα στα κράτη-μέλη που έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Νομοθετική Τάξη σχετικά ε, η συνθήκη σχετικά με το ευρωπαϊκό δικαίωμα ευρεσιτεχνίας. Σχετική νομοθεσία και η σχετικά με το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας δεν μπορεί να ληφθεί καμία συγκεκριμένη απόφαση αν δεν εφαρμόζεται αυτή η συνθήκη. Και πάλι λοιπόν υπάρχει αρκετή ευελιξία, ε, χάνεται η ομοφωνία, ούτε τα 28 είναι απαραίτητα, ούτε και χρειάζεται και να επικυρώσει κανείς αυτή η συνθήκη για να αρχίσει να ισχύει και για να ε, θεσπιστεί νομοθεσία για το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ας δούμε τώρα τις μελλοντικές ε, προοπτικές. Μίλησαν πολύ για αυτό το θέμα, όμως υπάρχουν πολλές τροποποιήσεις στη συνθήκη. Η δυνατότητα λοιπόν να υπάρχουν νέοι κανόνες της συνθήκης ε, για τις νέες πτυχές της διαφοροποίησης θα προκύψει από μία επαναδιαπραγμάτευση των συνθήκων που σχετίζεται με την επαναδιαπραγμάτευση του Ηνωμένου Βασιλείου για τη συμμετοχή του. Θα είναι πολύ δύσκολο αλλιώ να το αντιμετωπίσουν κατά την άποψή μου, αλλά θα είναι δύσκολο να υπάρχει κάτι για τη διαπραγμάτευση του Ηνωμένου Βασιλείου και από τις δύο πλευρές. Εάν αυτό όμως μας δώσει τη δυνατότητα, και νομίζω ότι αυτό θα το δούμε και σε ένα-δύο χρόνια, να δούμε κατά πόσον η συνθήκη εν γέννη Αντιμετωπίζονται ίσω κάποια θέματα που είναι πρωτίστως του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και κάποια πιο γενικά θέματα, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερη διαφοροποίηση εντός της συνθήκης. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δει αν θα πρέπει να ε, αναθεωρήσει τη θέση του και θα πρέπει να δούμε και αυτές ε, τις συνθήκες και εκτός ε, της ένομης τάξης. Παραδείγματος χάρη, τι θα γινόταν αν προσπαθούσαμε να τα φέρουμε στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εναλλακτική λύση θα ήταν βέβαια να προσπαθήσουμε να έχουμε συστηματικά μη ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και να έχουμε ένα σύστημα το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ε, κάποιες εξουσίες ε, ε, στα εθνικά κοινοβούλια το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει και συμμετοχή έτονη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης κάτι άλλο θα μπορούσε να είναι να ενισχύσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις συνθήκες αυτές εκτός του Ευρωπαϊκού Νομικού Πλαισίου, αλλά σε σχέση με αυτό. Παραδείγματο χάρη, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο που έχει λίγο μεγαλύτερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε σχέση με τα υπόλοιπα. Είναι θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί ήδη για το πώς θα ήθελε κάποιος να αναδιαρθρώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή όπως σας είπα να δημιουργήσει ένα κοινοβούλιο της Ευρωζώνης ή να υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Would του ευρωπαϊκού πλαισίου, λοιπόν, θεωρώ ότι όλα τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένοι ούτως ή άλλως να συμμετάσχουν. Όπως έγινε και με την Νομισματική Ένωση και με το Σέγγεν. Ελάχιστα κράτη-μέλη έχουν από νομική σκοπιά μόνιμη δυνατότητα opt-out. Και επίσης, ε, Υπάρχει και το εξή. Χρησιμοποιείτε και δύο το ευρωπαϊκό σύστημα για να εγκρίνετε του κανόνε σα και από εκεί και πέρα κάθε κράτο μέλο μπορεί να συμμετέχει ανα πάσα στιγμή. Και στα δύο αυτά τα διαφορετικά πλαίσια αυτό είναι το επιχείρημα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετέχουν. Και επίση να τονίσω ότι δεν έχει τεθεί και το κατά πόσον ε, ε, ευρωβουλευτές από κράτη-μέλη που δεν συμμετέχουν είναι υποχρεωμένοι να ψηφίσουν ή όχι. Ε, είναι πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ευρωβουλευτών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν όμως ε, ε, ευρωβουλευτές μιας χώρας μέλους που υπερψηφίζει κάτι, τότε δημιουργείται έτσι μια πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δημιουργήσει κάτι τέτοιο πολιτικό πρόβλημα μόνο αν οι ευρωβουλευτές από τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν είναι διαιρεμένοι και επομένως οι ψήφοι αυτών που δεν συμμετέχουν ε, θα είναι καθοριστικές για να κρίνουν το αποτέλεσμα και ουσιαστικά θα επιβάλλουν κάτι το οποίο δεν είχε την υποστήριξη της πλειοψηφίας ε, στα κράτη-μέλη που συμμετείχαν. Βεβαίως αυτό από τεχνική σκοπιάς είναι δυνατόν, αλλά επειδή ακόμα δεν έχει συμβεί και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συμβαίνει συχνά, δεδομένου ότι υπάρχει ένα σύστημα κομμάτων εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μήπως ε, στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα όπως ε, θα μπορούσαν να το θεωρούν κάποιον. Ε, εδώ έχετε και τα σημεία επαφής μου στην τελευταία διαφάνεια αλλά νομίζω ότι αυτά ήθελα να θίξω σε γενικές γραμμές. Ε, έχουμε μία μακροπρόθεσμη τάση, η οποία επιταχύνεται πάρα πολύ γρήγορα τα τελευταία χρόνια και Έχουμε τελείω διαφορετικέ μορφέ ολοκλήρωση, αλλάζει στου διάφορου τομεί, ε, καθώ επίση και πιο γενικά στον τομέα τη ενισχυμένη συνεργασία και λαμβάνει και νέε μορφέ. Η συνθήκη εκτό του νομικού πλαισίου και φυσικά και η νομοθεσία εντός του συνηθισμένου νομοθετικού πλαισίου που δεν είναι μεν διαφοροποιημένη αλλά στην πράξη είναι διαφοροποιημένη. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν τα οποία θα πρέπει ε, να τα λάβουμε υπόψη με κάποιο τρόπο. Επίσης κάτι τελευταίο. Ο επίσημος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δώσει το έναυσμα για την ενισχυμένη συνεργασία ποιος θα είναι. Από νομική σκοπιά, η ενισχυμένη συνεργασία μπορεί να ξεκινήσει μόνο αν τη ζητήσουν κάποια κράτη-μέλη, υπάρξει πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γίνει δεκτή και μόνο τότε μπορεί να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω τη συνένεσή του. Αλλά το κοινοβούλιο το να εγκρίνει ψηφίσματα και να λέει ε, δημοσίως ότι πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία ενισχυμένη συνεργασία και μάλιστα αν γίνεται αυτό συστηματικά ε, Δηλαδή, η Επιτροπή σας μαζί με τις αρμόδιες κάθε φορά επιτροπές ε, θα μπορούσαν μέσω νέων κανόνων και νέων κανονισμών να εξετάζουν κατά πόσον θέλουν να πιέσουν σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα υπέρ της ενισχυμένης συνεργασίας. Ε, επειδή δεν υπάρχει κάποια συστηματική διαδικασία ε, στα κράτη-μέλη, κάποιος από τους άλλους ομιλικέ είπε ότι δεν υπάρχει γαλλογερμανική πίεση, για παράδειγμα, για ένα θέμα. Ε, όταν δεν υπάρχει λοιπόν κάτι τέτοιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να προσπαθήσει να διαδραματίσει πολιτικό ρόλο, ώστε να παρακινήσει τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τομεί που έχουν σταματήσει για πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, ε, το καθεστώ των ιδιωτικών επιχειρήσεων, ε, η ε, αρχή τη μη διάκριση βάση σεξουαλικού προσανατολισμού κλπ. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία κολλησιεργούν συνεχώ η Επίτροπος Ράιχουτ, για παράδειγμα, στα τελευταία, στις τελευταίες 36 ώρες ε, που ήταν ε, αρμόδια, ε, είπε ότι ε, πρέπει να έχουμε ενισχυμένη συνεργασία. Βέβαια, αν κάποιο έχει μια μισή μέρα θητεία ακόμα, δεν μπορεί να πιέσει και πολύ τα πράγματα. Θα μπορούσατε όμω να πιέσετε τη νέα επιτροπή, την κυρία Γιούροβα ή τον κύριο Τίμερμαν, να πιέσουν αυτοί αυτά τα θέματα για να υπάρχει αυτή η συστημητική αναθεώρηση και να εξετάζεται κατά πόσον θα μπορούσε να είναι χρήσιμη η ενισχυμένη συνεργασία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαν από εκεί και πέρα να αντιγράψουν και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προσπαθήσουν όλα τα θεσμικά όργανα ευρύτερα να κάνουμε μια τακτική αναθεώρηση, κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει και στην ε, πιο συχνή χρήση της ενισχυμένης συνεργασίας. Η εναλλακτική λύση για την ενισχυμένη συνεργασία θα μπορούσε να είναι ολοκλήρωση εκτός του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλασίου, χωρίς να έχει τόσο σημαντικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι ουσιαστικά η θεσμική περίπτωση. Αυτές είναι πολιτικές τις οποίες βεβαίως θα μπορούσαν να κάνουν 10-15 κράτη-μέλη που αλλιώς δεν θα γίνονταν. Ή αλλιώς δεν θα γίνονται ε, εντό ε, του ευρωπαϊκού θεσμικού ε, Πλασίου. Ευχαριστώ πολύ. Uh, ευχαριστώ καθηγητή Πύρη, σας ευχαριστώ πολύ. Να σας καλημερίσω όλους. Έχουμε καθυστερήσει τώρα λίγο. Και θα θέλαμε να κάνουμε μια συζήτηση τώρα. Έχετε θίξει πολύ σημαντικά ζητήματα. Λοιπόν, να περάσουμε στην τελευταία παρέμβαση εκ μέρους των ομιλητών του Πάλελ να δούμε λίγο το μέλλον της σταγματικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τον καθηγητή Κάρλος Κλώσσα Μοντέρο εδώ για να μας παρουσιάσει για ε, τα διάφορα θέματα ε, όπως τα βλέπει αυτός. Καταρχάς να σας πω ότι είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. οι περισσότεροι από αυτούς που κάθονται εδώ στο πάνελ ανέφεραν το έργο μου και πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η Επιτροπή ε, άπτεται κάποιων θεμάτων που συνήθως είναι το έργο μου. Ασχολήθηκα ε, και με την ολοκλήρωση και με τη διαδικασία κύρωσης της συνθήκης και πολλά από τα μέλη της Επιτροπής ασχολήθηκαν με τα θέματα αυτά. Ο Ρίτσαρ Κόρμπεν, ο Γιολάιλεν ε, και φυσικά θα πρέπει να αναφέρω και τον Αλτιέρο Σπινέλη, που είναι ένας από τους ε, ε, πιο εγνωσμένου κύρους ε, εκπροσώπους της Επιτροπής σας. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τους μελλοντικούς δρόμους ε, της συνταγματικής εξέλιξης. Μπαίνουμε σε άγνωστα μονοπάτια ε, δεν μπορεί κανεί βέβαια να κοιτάξει στη μαγική μπάλα, στην κρυστάλλινη μπάλα για να δει τι θα γίνει. Αυτό λοιπόν που θα προσπαθήσω να κάνω είναι να σα παρουσιάσω πολύ γρήγορα ένα δίλημα για το μέλλον. Και το δίλημα θα μπορούσε να διατυπωθεί ω εξή. Η πρώτη μεταρρύθμιση της συνθήκης ε, εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη δεκαετία του 50 είχαμε ε, περίπου 8 διαφορετικές διαπραγματικές μεταδιαπραγματεύσεις διαπραγματεύσεις της συνθήκης ε, ξεκινήσαμε από τις πρώτες, μετά περάσαμε στο Μάστριχτ, στο Άμστερνταμ, στη Νίκαια, στη Λισαβόνα και φυσικά έχουμε και το ε, Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον. Ε, θέλουμε να περάσουμε σε πρωτογενές δίκαιο, πράγματα τα οποία είτε βρίσκονται σε δευτερογενές ε, δίκαιο, είτε σε άλλες θεσμικές ρυθμίσεις αλλά φαίνεται ότι δεν υπήρχε γενικότερα διάθεση μετά το 2005 και τα δημοψηφίσματα για νέες αναθεωρήσεις συνθήκης. Ε, τελικά όμως είχαμε δύο αναθεωρήσεις συνθήκης και κάποιες άλλες διακυβερνητικές ε, συμφωνίες. Ε, και φαίνεται ότι παρά τη διάθεση του 2005 που έλεγε ότι δεν θα γίνουν άλλες αναθεωρήσεις συνθήκη, φαίνεται ότι αυτή είναι συνειφασμένη με την ίδια τη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πρώτο τμήμα του διλήμματος. Το δεύτερο θέμα του διλήμματος είναι ότι τα αιτήματα για αναθεώρηση της συνθήκης ε, αντιβαίνουν τις απαιτήσει του άρθρου 48 που απαιτούν ομοφωνία συν ε, εσωτερική έγκριση σε εθνικό επίπεδο. Μέχρι λοιπόν αυτό ο συνδυασμό των ε, αιτήσεων και των απαιτήσεων ε, δεν υπάρξει, τότε κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνει αναθεώρηση του συντάγματος, της συνθήκης είναι όλο ένα λοιπόν και πιο δύσκολο να γίνεται αναθεώρηση της συνθήκης. Και φυσικά οι πιο σημαντικές εναλλακτικέ λύσεις κατά την άποψή μου είναι ακόμα πιο προβληματικές για λόγους τους οποίους θα σας εξηγήσω εντός ολίγου. Καταρχάς να σας πω πολύ σύντομα ποια είναι τα τρέχοντα αιτήματα τα οποία οδηγούν στο αίτημα για αναθεώρηση της ε, συνθήκης στο εγγύς παρελθόν. Η γερμανική κυβέρνηση, ε, ε, αν και φαίνεται ότι αυτό αναθεωρήθηκε τώρα, ε, κάποια στιγμή αναφερόταν πολύ συγκεκριμένα στην ανάγκη αναθεώρησης για να διαχωρίσουμε τον εποπτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τους υπόλοιπους ρόλους της και ενισχυμένος έλεγχος στις πολιτικές προπολογισμού. Ε, σε εθνικό επίπεδο και αυτό θα έπρεπε να γίνεται με αναθεώρηση συνθήκης καθώς επίσης και τις συμβατικές ε, ε, συμφωνίες που αποφασίζονται στη ΟΤΟΥΠΑΚ σε αυτή τη δέσμη των δύο μέτρων. Το Συντηρητικό Κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το συνδυάσω ίσως και με τον Βρετανό Πρωθυπουργό αλλά ας μιλήσω στο κόμμα, για το κόμμα καλύτερα αναφέρθηκε σε δύο διαφορετικές δυνατότητες ε, αναθεώρησης. Το ένα είναι η κατανομή των εξουσιών, κυρίως στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της μετανάστευσης όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία και επίσης ε, ε, η συμβολικού χαρακτήρα και επισημοποιημένη ανάγκη για όλο ένα και περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπάρχουν και χώρες οι οποίες έχουν λάβει αρνητική στάση. Ε, ε υπήρχαν για παράδειγμα 100 χώρες που ε, θεώρησαν ότι δεν χρειάζεται αλλαγή τη συνθήκης και ε, μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές βάσει αυτών. Και επίσης και η γαλλική κυβέρνηση και ο πρόεδρος Ολάντ και ο πρωθυπουργός του είπαν ότι δεν χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση της συνθήκης. Ε, τα πράγματα βέβαια είναι λίγο ασαφή. Πριν από τι ευρωεκλογέ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφερόταν σε κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορεί να χρειάζονταν κάποιε μεταρρυθμίσει στι παρούσε συνθήκε. Ε, το ένα είναι ε, τα ευρωομόλογα και το Ταμείο ε, του Χρέους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τώρα δεν έχει αναφερθεί σε μεταλλοντική μεταρρύθμιση της συνθήκης και δεν έχει συζητηθεί κατά πόσον αυτό είναι χρήσιμο και ουσιαστικό και ε, δυνατό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, εδώ έχουμε μια σειρά από πράγματα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι οριστικά. Ποια είναι οι περιορισμοί της διαδικασίας ε, που σας ανέφερα προηγουμένως. Καταρχάς είναι συνδυασμό δύο πραγμάτων. Καταρχάς υπάρχει ο κανόνας της ομοφωνίας, που δημιουργεί μια πολύ περίπλοκη κατάσταση. Ο κανόνας της ομοφωνίας θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ αυστηρός ε, και επιτρέπει συγκεκριμένους κανόνες, γιατί πρέπει όλοι να δίνουν τη συγκατάθεσή τους για συγκεκριμένους κανόνες. Αλλά επίσης ο κανόνας της ομοφωνίας μας έχει βοηθήσει να εντοπίσουμε και ποιες είναι οι πρακτικές δυσκολίες της ομοφωνίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ομοφωνία, μπορεί ο καθένας να μπλοκάρει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για να υπάρξει ε, συνένεση. Ε, είναι δημοκρατικό μεν στη θεωρία, αλλά στην πράξη είναι ένας πάρα πολύ δύσκολο κανόνας και δεν εφαρμόζεται εύκολα. Επιπλέον, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το άρθρο 48 δημιουργεί μια περίπτωση ΚΑΤΣ όπου ε, η ομοφωνία μπορεί να αλλάξει μόνο ομόφωνα. Έχουμε λοιπόν ένα φαύλο κύκλο. Δεν μπορεί να αλλάξει η ομοφωνία εύκολα γιατί χρειάζεται ε, ε ομοφωνία για την αλλαγή του ίδιου κανόνα. Επομένως θα είναι πολύ δύσκολο. Το πρόβλημα με την ομοφωνία είναι ότι υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερος αριθμός ε, ε, παραγόντων που ε, σε εσωτερικό επίπεδο παρεμβαίνουν. Έχουμε διάφορα κοινοβούλια. Αυτή τη στιγμή έχουμε 52 κοινοβούλια τα οποία θα παρέμβουν σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση, ανάλογα φυσικά με τις εξουσίες που έχουν. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο έχουμε μέχρι και 7 ε, κοινοβούλια ε, αλλά, και ο καθένα έχει διαφορετική συμμετοχή, αλλά φυσικά είναι πολύ μεγάλο ο αριθμό. Επίση, ε, τα ανώτατα συνταγματικά δικαστήρια παρεμβαίνουν σε πολλέ περιπτώσει και έχουν αποφάσει που ζητούν θέματα αναθεώρησης και υπάρχει και συνταγματική μεταρρύθμιση που έχει ε, ενσωματωμένη την αλλαγή της συνθήκης και αυτό σημαίνει ότι είναι και από πρακτική σκοπιάς πολύ δύσκολα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών μέσω δημοψηφισμάτων. Και εδώ ε, είναι πολύ ε, σημαντικό το θέμα αυτό γιατί στο παρελθόν ήταν ελληματική η χρήση του και επανήλθε από το Ηνωμένο Βασίλειο στη δεκαετία του 70, δεν θα έλεγα ε, παρεπιπτόντως, αλλά σίγουρα δεν το ε, υπολόγισαν σωστά τα πράγματα όταν το επανέφεραν. Και υπάρχει κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό στη, συζήτηση αυτή, είναι ότι αλλάζουν ε, συνεχώς οι κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες μεταξύ των ε, σταδίων της διαπραγμάτευσης της συνθήκης και της κύρωσης της συνθήκης. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Μπορείτε να δείτε και τι γίνεται με την ίδια τη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά και στο παρελθόν. Αυτό που έχουμε είναι ότι έχουμε ε, αυξημένο αριθμό διαφόρων παικτών, διαφόρων παραγμόντων που συμμετέχουν στη συζήτηση. Εδώ έχετε ένα διάγραμμα το οποίο σας δείχνει λίγο πώς έχει κατάσταση και η πιο σημαντική γραμμή, αν θέλετε να δείτε εδώ, είναι η μπλε γραμμή με τα κόκκινα τετράγωνα που δείχνει τη διάρκεια σε μήνες οποιασδήποτε διαδικασίας κύρωσης. Και αυτό που βλέπετε είναι ότι υπάρχει μια τάση αύξησης τη διάρκεια ε, διαδικασίας κύρωσης με δύο σημεία καμπή που είναι η Ευρωπαϊκή ε, Κοινότητα Άμυνα και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα πιο πρόσφατα. Εκεί σταμάτησε η διαδικασία και γι' αυτό κόβεται και η γραμμή. Επίσης, στην κόκκινη γραμμή έχουμε τον αριθμό των χωρών που κυρώνουν και νομίζω ότι αυτό ε, δεν είναι απόλυτα συσχετισμένο. Υπάρχει μια σχέση μεταξύ των κρατών που κυρώνουν και τη διάρκεια της διαδικασίας κύρωσης. Και εδώ ας σας κάνω μια προσωμείωση. Ε, η διάρκεια είναι αντίστοιχη με τις δυσκολίες. Όσο πιο μακρά είναι η διαδικασία, τόσο μεγαλύτερες είναι οι δυσκολίες και έχουμε και ορισμένες ε, αποτυχίες οι οποίες πρέπει να κυρωθούν σε κάποιες περιπτώσεις, όπως βλέπουμε σε αυτά τα δύο κενά. Τώρα, το διάγραμμα αυτό Δεν θα σας το αναλύσω, θα περάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο που, σημαίνει την που μιλά για την αλλαγή των κανόνων επικύρωσης σε καιρούς κρίσης. Όπως γνωρίζετε, στη διάρκεια της κρίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη της έχουν επεξεργαστεί νέες συνθήκες για την οικονομική διακυβέρνηση και αυτές οι συνθήκες προχώρησαν στην επικύρωση χωρίς ομοφωνία. Η πρώτη από αυτές τις συνθήκες παραδόξως ούτε καν επικυρώθηκε. Ήταν ε, η διευκόλυνση ε, για την δημοσιονομική διευκόλυνση και μάλιστα σε κάποια κράτη, σε κάποιες περιπτώσεις ούτε καν επικυρώθηκε. Συζητήθηκε από τα κοινοβούλια, εγκρίθηκε στα κοινοβούλια, ενώ η οικονομική συνεισφορά που έπρεπε να ε, βάλει κάθε κράτος δηλαδή και αυτή πέρασε έτσι, συζητήθηκε μόνο από τα κοινοβούλια. Τώρα, Έχουμε την αναθεώρηση του άρθρου 136 και τη, για το EFSF και τη διαφορετικούς μηχανισμούς για την επικύρωση. Το 136 απαιτεί τη φυσιολογική διαδικασία, δηλαδή ομοφωνία και η παραπομπή στην χώρια διαδικασία επικύρωσης. Ενώ μετά έχουμε τα 12 από τα 17 κρατημέλη και πλήρη ανανέωση, καινοτομία όσον αφορά την επικύρωση των συνθήκων. Τέλος, η συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας οδήγησε, σχετίζει μάλλον την επικύρωση με το μέγεθος συμβολής στο Ταμείο. Ένα ενδιαφέρον ε, στοιχείο σε αυτή τη συνθήκη όσον αφορά την επικύρωση είναι ότι το, ο μήνυμο αριθμός ε, κρατών ήταν 8. Πολύ μικρός αριθμός δηλαδή. Και ακόμα πιο σημαντικό και ενδιαφέρον είναι ότι τέσσερα κράτη-μέλη απαιτούνταν να επικυρώσουν για να αρχίσει να ισχύει η συνθήκη λόγω του μεγέθους της συμβολής τους. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Αυτές ήταν οι χώρες που πάντοτε χρειάζονται για να αρχίσει να ισχύει μια συνθήκη. Και αυτό δημιούργησε μια συμμετρία ανάμεσα στις αξίες επικύρωσης για κάποιες χώρες, διότι η συνθήκη ισχύει το ίδιο για όλα τα συνυπογράφοντα κράτη, ωστόσο η ποιότητα των διαφόρων διαδικασιών ήταν ε, διαφορετική ανάλογα με τη συμβολή του στο Ταμείο. Ποιε είναι οι επιπτώσει αυτών των νέων τα κανόνων που εισήχθησαν μέσω αυτών των τριών συνθηκών. Έχω φτιάξει αυτό το άλλο γράφημα που πολύ συχνά δείχνει τι αλλαγέ. Και εδώ οι ενδιαφέρουσε γραμμέ είναι αυτή η μαύρη που έχουμε τον αριθμό των ε, κρατών που επικυρώνουν την πράσινη γραμμή που αντικατοπτρίζει τη διάρκεια της διαδικασίας και βλέπετε πως υπάρχει απόλυτο συσχετισμός ανάμεσα στην απέτηση ελάχιστου αριθμού κρατών και τις, δια... και τις σχέσεις με τη διαδικασία. Βέβαια, επίσης είναι ενδιαφέρον, ενδιαφέρουσα η κόκκινη γραμμή που λέει το βάρος για τα κράτη. Για το 136 έχουμε απόλυτη σύμπτωση ανάμεσα στις τρεις γραμμές, αλλά βλέπετε ότι στο τέλος περισσότερα κράτη από αυτό που ήταν απαραίτητα τελικά επικύρωσαν, την, τη συνθήκη. Ενώ στο Fiscal Compact όλα τα κράτη εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο επικύρωσαν ε, παρά το γεγονός ότι δεν χρειαζόταν η ομοφωνία. Δηλαδή, η αφαίρεση της ομοφωνίας δεν αποκλείει ότι σχεδόν ομόφωνα γίνεται η επικύρωση των συνθηκών αυτών. Έχοντας αυτό υπόψη, θα σας παρουσιάσω και το εξή, δηλαδή το... θα ε, κοιτάξω <laughs> κρυστάλλινη σφαίρα μου, ε, προβλέψεις για το μέλλον εάν θέλει να προχωρήσει η Ένωση στην αναθεώρηση των συνθηκών. Και εδώ βλέπουμε τέσσερα διαφορετικά σενάρια. Το πρώτο ακριβώς ε, δεν προβλέπει τίποτα όσον αφορά την επίσημη συνταγματική μεταρρύθμιση και την εφαρμογή του άρθρου, 148. Ε, Εδώ ε, το έχω ήδη αναφέρει στο πρώτο τμήμα, αφορά διαθεσμικές διοργανικές συμφωνίε, για παράδειγμα ή άλλου είδους άτυπους μηχανισμούς και έπειτα έχουμε και τις συνθήκες προσχώρησης που δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να τυποποιήσουν αυτές τις ε, αλλαγέ. Αλλά εγώ θεωρώ πως δεν είναι και πολύ νομιμόφρον ε, λύση γιατί ε, μέσω της συνέλευσης το Εθνικό Κοινοβούλιο μπορεί κάθε φορά μέσω του άρθρου 48 να έχει την αρμοδιότητα. Οι περισσότερες κυβερνήσεις εκτός από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο επειδή έχει μπει στην ημερήσια ε, διάταξη μόνο μπορεί να αυτό να συζητηθεί εντός του Κοινοβουλίου. Όπως σας είπα, <clears throat> αυτές οι, οι περισσότερες κυβερνήσεις προτιμούν την ε, άτυπη προσέγγιση. θα κάνουμε. Επίσης, ε, το δεύτερο σενάριο αφορά την τρέχουσα διαδικασία και ε, αυτή προβλέπει την ομοφωνία συν την επικύρωση. Εγώ πρέπει να σα πω ότι έχω ήδη υπογραμμίσει ορισμένα από αυτά τα στοιχεία. Αυτός ο μηχανισμός λοιπόν μπορεί να εφαρμοστεί πολύ συγκεκριμένα για τη συμπερίληψη του φορολογικού στοιχείου στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που προβλέπει η συνθήκη. Αυτό όμως που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι το εξή παράδοξο. Από τη μια λέμε ότι το δημοσιονομικό σύμφωνο δεν είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι που αφορά μόνο ως ε, συμμετέχουν ε, και αφορά στα κράτη-μέλη. Από την άλλη όμως λέμε ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται ευρύτερα. Αυτό είναι ένα παράδοξο. Τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχουν μέσα από τη συνθήκη. Βεβαίως αν υπάρξει τελικά μια ουσιαστική τροποποίηση της ε, συνθήκης. Τώρα, α δούμε τα μειονεκτήματα. Ενδέχεται πάρα πολλά κρατημέλη να μην θελήσουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Αναφέρθηκα στη Γαλλία, ο Πρωθυπουργό και ο Πρόεδρος είπαν ότι δεν θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο και υπάρχει και άλλη μία άλλη σημαντική προϋπόθεση. Ε, αν αρχίσει, αυτό το θεματολόγιο μπορεί και να διευρυνθεί, περαιτέρω. Ε, ο Γκόμεσος να μην μπορέσει να ελέγξει το όλο θέμα εκ των προτέρων και Κατ' ουσίαν βεβαίως ε, ένα σημαντικό παράγων είναι το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φτάνουμε λοιπόν στην επιλογή παριθμών 3 είναι η επιλογή που ανέφερα και πριν από λίγο αφορά το χρονικό διάστημα πριν από 10 χρόνια αφορά το μοντέλο της Πινελόπης όπως αποκαλείται και αυτός είναι ένας ε, μηχανισμός ε, για την εφαρμογή των συνθήκων άρθρο 48 όμως ε, παράλληλα να υπάρχει και μια δήλωση με βάση την οποία τα κράτη-μέλη τα οποία δεν προτίθενται να συμμετέχουν στη νέα συνθήκη παρόλα αυτά θα πρέπει να επικυρώσουν τη συνθήκη αυτή για να μπορούν να εφαρμόσουν άλλα κράτη-μέλη. Εδώ προκύπτουν κάποια θέματα. Είναι το θέμα ε, της, ε, του σκότους που δημιουργεί αυτή η συνθήκη. Το δεύτερο πιο σημαντικό ερώτημα είναι ότι και πάλι εμφανίζεται μια κατάσταση του στυλ catch 22. Αν τα κράτη δεν θέλουν και δεν συμφωνούν, γιατί τότε να πρέπει να επικυρώσουν μια συνθήκη. Πάλι η ίδια κατάσταση catch 22 και αυτό το σκηνικό εμένα δεν μου φτάνει πολύ ε, πρακτικό Πάμε στο τέταρτο σενάριο, αναθεώρηση εκτός των συνθήκων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ υπάρχουν ε, υποστηρικτές ε, και κύριος υποστηρικτής είναι το Συντηρητικό Κόμμα, το οποίο θα ήθελε να αποδώσει κάποιες ιδιαίτερες εξουσίες σε μια μελλοντική κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως θα θυμάστε, η Βρετανική κυβέρνηση δεν ήθελε να ακολουθήσει τη μεταρρύθμιση το άρθρο 48 και αυτό ανάγκασε ε, πολλούς να επικυρώσουν τη συνθήκη εκτός του ίδιου του νομοθετικού πλαισίου. Ε, υπάρχει βέβαια ένα προηγούμενο και αυτό το προηγούμενο σημαίνει ότι αυτά θα πρέπει να είναι εφικτά και αποτελεσματικά ε, τουλάχιστον ε, για το πώς πρέπει να προχωρήσουν τα κράτη-μέλη. Και εδώ φτάνουμε και σε άλλο ένα σενάριο. Είναι η δημιουργία ενός ε, πυρήνα δηλαδή αυξημένη διαφοροποίηση όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και από την καθηγήτρια Western. Για να ολοκληρώσω θέλω να σας πω το εξής. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον μεγαλύτερο αριθμό εκείνων που καταθέτουν βέτο και σε πόσο πιο δύσκολο είναι να περνάει πλέον μια συνθήκη με την αρχή της ομοφωνίας. Προκύπτουν νέες διαδικασίες αναθεώρησης ε, που ε, συνδυάζουν το ε, διεθνές δίκαιο με εσωτερικές διαδικασίες. Αυτό που είναι πολύ πιο πιθανόν είναι οι νέες συνθήκες να ακολουθήσουν τη νέα διαδικασία παρακάπτοντας ε, πρώην προϋποθέσεις που υπήρχαν σε προηγούμενες συνθήκες. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία, κύριε καθηγητά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε και τώρα περνάμε στις ε, ερωταπαντήσεις. Και έχω κάποιες ερωτήσεις. Ξεκινάμε με την ε, κυρία Σπινέλη. Έχει το λόγο. Thanks very Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που είπατε. Έχω δύο ερωτήσεις να υποβάλω. Η μία αφορά την καθηγήτρια κυρία Μόνικα Κλάις και η άλλη ε, τον καθηγητή κύριο Κλόζα, αλλά και μία ε, ερώτηση προς τον καθηγητή Πίερς. Steve Η πρώτη ερώτηση αφορά στα συνταγματικά δικαστήρια. Πολλοί αρέσκονται στην ιδέα ότι τα εθνικά συνταγματικά δικαστήρια ε, μπορούν να λειτουργήσουν κατά της ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης, αν αυτή θεωρηθεί ότι είναι κάτι το αρνητικό. Βλέπουμε να υπάρχει ένα είδος αντίδρασης των εθνικών δικαστηρίων και προς την ολοκλήρωση είναι μια αντίδραση απέναντι στην απειλή να γνωηθεί η απόφαση των δικαστηρίων. Και έχουμε και απειλή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που και αυτό υφίσταται αυτή την απειλή να γνωηθεί νοηθεί να χάσει την εξουσία του από κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά κυρίως ε, σε σχέση με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, ε, το οποίο κάπως είναι και εκτός των αρμοδιοτήτων των ε, κυβερνήσεων. Άρα λέει τι προκύπτει. Προκύπτει η συγκέντρωση της εξουσίας στην εκτελεστική εξουσία, αυτό που ο μας αποκαλεί την ομοσπονδιοποίηση των εκτελεστικών ουξιασιών. Και θα ήθελα να μας πείτε ε, τι πιστεύετε για αυτές τις εξελίξεις, που κατ' ουσίαν ε, εδώ πρόκειται για μια μεταρρύθμιση των συνθήκων. Η μεταρρύθμιση προχωράει ακόμα και αν δεν την έχουμε θεσπίσει. Ίσως λοιπόν η εναλλακτική λύση υπαριθμών 4 που περιγράφηκε από τον καθηγητή κύριο Κλόζα, αυτή να ισχύει, δηλαδή να πρόκειται για συνθήκες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ελέγχονται ούτε από τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά ούτε και από το Ευρωπαϊκό. Κατόπιν υπάρχει η ερώτηση της αυτοεξαίρεσης που την ε, παρουσίασε ο καθηγητή κύριος Στίβ και θέλω να ρωτήσω κατά πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει ένα μόνιμο opting out. Μόνιμη αυτοεξαίρεση, διότι εσείς θέσατε και το θέμα της μόνιμης διαφοροποίησης ε, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και ρωτώ, πώς θα εφαρμοστούν οι πολιτικές μετανάστευσης, ε, χορήγησης ασύλου, που είναι ευρωπαϊκές πολιτικές και περιλαμβάνουν αυτή τη μόνιμη δυνατότητα αυτοεξαίρεσης. Τώρα, το opting out στο ευρώ. Κύριε καθηγητά Πίερς, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει αυτό, opting out από το ευρώ. Ε, και ζητώ συγγνώμη που κρυγόρησε, πρόεδρος. Μόνο πέντε λεπτά έχουμε. Κύριε Γιουλάινεν, έχετε το λόγο. Αφού έχουμε μόνο πέντε λεπτά, δεν θα κάνω ερωτήσεις. Απλώς θα αναφερθώ στα συμπεράσματά μου. Αυτά που ακούσαμε λοιπόν είναι το εξής, ότι με τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση προκύπτει και λιγότερη διαφάνεια. Και όσον αφορά εμάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει όλο και πιο περιορισμένη δυνατότητα δημοκρατικού ελέγχου. Αυτό όμως πρέπει να μας απασχολήσει. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν με όλα αυτά τα πρότυπα και τις συνθήκες πώς είναι δυνατόν να επανέλθει ο δημοκρατικός έλεγχος. Άκουσα αυτά που προτείνατε και θέλω να σας πω το εξής. Η δική μας άποψη είναι ότι οι συνθήκες αυτές θα πρέπει να επανέλθουν στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη ακριβώς όπως το εκβιάσαμε με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Δηλαδή, η πρώτη εναλλακτική λύση για μας είναι αυτές οι ειδικέ συνθήκες να γίνουν πάλι κανονικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε εμείς να διαδραματίσουμε ρόλο εκτός των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, ναι εντάξει θα άκουγαν την άποψή μας, αλλά δεν θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε για τίποτα και αυτό δεν μπορεί να είναι εναλλακτική λύση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εν ολίγης, τι θα γίνει στο μέλλον, για να δούμε και τι θα κάνουν τα δικαστήρια, γιατί ξέρετε, βαδίζουμε επί ξηρού ακμής. Αυτή τη στιγμή το μπαλάκι πάει από την Καλσρούη στο Λουξεμβούργο, Κατ' ουσίαν όμως οι συνθήκες ε, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Χρειαζόμαστε ένα καλύτερο πρωτογενές δίκαιο, λειτουργούμε contra legem και Απλά αυτό γίνεται ανεκτό διότι κανείς δεν θέλει την καταστροφή. Όμως χρειαζόμαστε μια νέα νομοθετική βάση για την ΟΝΕ. Το Κοινοβούλιο κατά την προηγούμενη θητεία προέβησε τρία ψηφίσματα σχετικά με τη συντακτική συνέλευση γιατί έχουμε αυτό το δικαίωμα πρωτοβουλίας και ελπίζω ε, σε αυτή τη θητεία να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυνατότητά μας γιατί ξέρετε η συντακτική συνέλευση θα είχε την ευκαιρία όλα αυτά να τα τακτοποιήσει και να εξάγει πολιτικά συμπεράσματα. Για μένα λοιπόν η συντακτική συνέλευση για μένα είναι η μόνη δυνατότητα να επιφέρουμε διαφάνεια και ε, ουσιαστική νομιμοποίηση. Έχετε ένα λεπτό παρακαλώ. Δύο ερωτήσεις ήθελα να κάνω. Κύριε γλώσσα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχει δυνατότητα να προτείνουμε μία μεταρρύθμιση, σημαντική μεταρρύθμιση των συνθήκων μας, σε μορφή πολιτικής ερώτησης προς τους πολίτες και αν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει δημοψήφισμα τώρα που είναι και στη μόδα, ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι ώστε να μπορούν να απαντήσουν σε μία εντολή η οποία θα είναι αποαιρέγγυτη από πολιτική σκοπιά για μία σειρά από μεταρρυθμίσει, α τι αποκαλέσουμε ομοσπονδιακέ ε, ευρωπαϊκέ. Έστω ότι κάποιο προτείνει μία μεταρρύθμιση. Μπορούν να συγκαλέσουν ε, δημοψήφισμα για όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν θα ήταν ε, άρση ουσιαστικά όλων των συζητήσεων περί εθνικής νομιμοποίησης. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω ε, την κυρία Κλάες αν είναι δυνατόν μέσω της κύρωσης που γίνονται στην Ευρώπη, αν μπορούμε να ξεπεράσουμε και την ανάγκη εθνικής επικύρωσης. Διότι αυτή τη στιγμή πρέπει να επικυρωθεί οτιδήποτε από τις 28 χώρες μέλη. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Κάνουμε συμφωνίες με πολλές πλευρές του κόσμου. Μήπως θα μπορούσαμε να αποφύγουμε αυτή την περιττή λοιπόν επικύρωση από όλα τα εθνικά κοινοβούλια για αυτές τις διεθνείς ε, ε, συμφωνίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο πολύ σύντομα. Um, guest speakers. Στους ομιλητές μας. Παρακαλώ. να πω αυτή την ιδέα για την πρωτοβουλία στο άρθρο 48. Ε, να σας πω ότι αυτό είναι κάτι καινούριο στη συνθήκη της Λισαβόνας. Το Εθνικό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία. Και εγώ πραγματικά θα ήθελα να σας παρακινήσω να το κάνετε. Θα βρούμε και εμεί δουλειά, η πανεπιστημιακή, γιατί θα πρέπει να γράψουμε και μελέτε, να αναπτύξουμε ιδέε και να συμμετέχουμε και στη συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν και χρήσιμο. Βεβαίω χρειαζόμαστε και την πλειοψηφία των κρατών μελών. Απλή πλειοψηφία κρατών μελών. Αν ξεκινήσει λοιπόν αυτή η διαδικασία, ποιε θα ήταν οι βασικές πτυχέ που θα επιτρέψει ε, να έχετε και τη συμμετοχή των ε, περισσότερων κρατών μελών για να ξεκινήσει η διαδικασία. Και εδώ νομίζω ότι θα ξεκινήσουν και διαφορετικές εναλλακτικέ λύσεις ε, που όπως για παράδειγμα για την Ευρωπαϊκή ε, αυτή τη ε, διάσκεψη που γινόταν για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, το οποίο ήταν τελείω διαφορετικό τη δεύτερη φορά από την πρώτη. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, εγώ το υποστηρίζω και μάλιστα αυτή είναι η πιο περιορισμένη συμβουλή που θα μπορούσα να σας δώσω, να είστε προετοιμασμένοι για διαφορετικές λύσεις και διαφορετικές εξελίξεις και ειδικά η Επιτροπή σας θα πρέπει να ε, το προτείνει αυτό, να εξετάζει τα διάφορα ενδεχόμενα, διότι ορισμένες φορές κάπως πρέπει να πλαισιώνονται όλες αυτές οι ιδέες, οι οποίες δεν είναι πάντα στο καθημερινό θεματολόγιο, αλλά μπορεί να έχουν ε, σημαντικές συνέπειες. Ε, πολλές ε, μελέτες, και νομίζω ότι θα το ακολουθήσουν και οι συνάδελφοι, καταλήγουν στο αποτέλεσμα ότι το σχέδιο κειμένου του Σπινέλη το 1964 δεν ήταν το το κείμενο το οποίο τελικά ψηφίστηκε, και αλλά θα δούμε ότι πολλά από αυτά που είχε προτείνει τότε βρίσκονται τώρα στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστώ κυρία Κλάης. Θα απαντήσω την ερώτηση της κυρίας Πινέλη και μετά θα το περάσω στο, στον και Κάρλος Κλώσσα γιατί νομίζω απευθυνόταν και στους δυο μας. Γιατί λέει ε, λέτε ε, και πώς θα αντιδράσουμε σε αυτο ε, το κίνδυνο κένωσης νοήματος του Κοινοβουλίου υπάρχει ή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, ε πιστεύω πως θα πρέπει να υπάρξει διάκριση γιατί στα εθνικά συνταγματικά δικαστήρια σε περιπτώσεις τροποποίησης των συνθήκων ή υπό τις συνθήκες όπως ισχύουν. Τα συνταγματικά δικαστήρια σε περίπτωση μεταρρυθμίσεων ε, συνθήκων μπορούν να μπλοκάρουν τα συνταγματικά δικαστήρια για την επικύρωση γιατί δεν υπάρχει υποχρέωση. Παραδόξως δεν το έχουν κάνει ποτέ αυτό. Δηλαδή καμία τροποποίηση της συνθήκης δεν έχει ποτέ σταματήσει.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 Υπάρχει, όντω αισθάνονται ότι πρέπει να αντισταθμίσουν την απώλεια εθνική δημοκρατία και του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων. Δύο όμω ολόκληρη την εικόνα κανεί, Έχω ένα πρόβλημα με τα εθνικά συνταγματικά δικαστήρια, τα οποία κατά κάποιο τρόπο πιστεύουν ότι μπορούν να αντικαταστήσουν την εθνική δημοκρατία και τα εθνικά κοινοβούλια και να αποφασίσουν για το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. σε μονομερή τρόπο. Το μονομερέ του θέματο με ενοχλεί εμένα. Ίσως ο Κάρλο Κλώσσα βέβαια να πει κάτι άλλο. Ε, ευχαριστώ κύριε Κλώσσα Ματέρο. Εδώ σας ε, ρωτούν και σας ξαναρωτούν. Παρακαλώ σύντομα να απαντήσετε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα προσπαθήσω. Ευχαριστώ την κυρία Σινόλ, Σπανέλη, Σπινέλη για την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, αλλά θα πω αγγλικά τα υπόλοιπα. Ε, το θέμα δεν είναι αν τα συνταγματικά δικαστήρια είναι οι θεματοφύλακες των συνταγματικών αξιών ή όχι. Ε, πρέπει πιο μακροπρόθεσμα να το δούμε αυτό. Είναι μια διαδικασία που σημαίνει συνταγματική ε, αλλαγή ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα όσον αφορά τα δημοσιονομικά και μακροοικονομικά μακροοικονομική διακυβέρνηση υπήρξαν αλλαξές. Καταρχήν έχουμε αλλαγή για το ε, διπλό και το εξαπλό πακέτο και έπειτα έχουμε εθνικές συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις όπως στη χώρα μου η δημοκρατική ποιότητα αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι <laughs> αφισβητήσιμη. Έχουμε δηλαδή μια διαδικασία βαθιάς μετατροπής της ουσίας των κανόνων χωρίς όμως ουσιαστική ε, ε, ε, συμβολή των δημοκρατικών διαδικασιών. Έτσι πρέπει να το δούμε και η αντίδραση των συνταγματικών δικαστηρίων θα πρέπει να αναμένεται. Και με, που δεν είναι και εντυπωσιάζει που δεν είναι και πιο έντονη η αντίδραση των συνταγματικών δικαστηρίων. Συνδεόμενη με αυτή είναι ίσως η ερώτηση του κύριου Χαωρή όσον αφορά την επικύρωση των διεθνών συνθηκών, διότι σε μεγάλο τμήμα αυτών των εθικών είναι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και δεν έχω καμία ειδική θέση που να Πρέπει να έχουμε ένα σύνολο στην ουσία που δημιουργείται ένα είδος πολύ συμπαγούς συνόλου κανόνων για το ποιο είναι, είναι το σωστό οικονομικό σύνταγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν το κάνουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε ισχυρή δημοκρατική ε, συμβολή, ε, συμμετοχή. Για, πραγματικά διστάζω να σας το αιτιολογήσω αυτό γιατί δεν νομίζω πως μπορείτε να, να το κάνουμε αυτό γιατί τελικά ένας επιπλέον μηχανισμός ελέγχου είναι και στην περίπτωση της TTIP είναι ε, αυτό το θέμα που πρέπει να κρατήσουμε υπόψη μας ε, γιατί μπορεί να προκύψουν εκεί ε, αντιφάσεις και συγκρούσεις. Τώρα, για σε σχέση με ένα ευρωπαϊκό δημοψήφισμα, δεν νομίζω πως κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Και ούτε και είναι και θεμητή αυτή η πρόταση. Δεν είναι θεμητό και δεν είναι εφικτό γιατί σε ορισμένε χώρες έχουν, διαφορετικ... έχουν περίεργο καθεστώς τα δημοψηφίσματα στη Γερμανία κυρίως αλλά και αλλού και στην Ολλανδία το δημοψήφισμα του 2005 ήταν ε, παράξενο. Για άλλες χώρες όπως το Βέλγιο ίσως ήταν δύσκολο να εισαχθεί κάτι τέτοιο. Ένα κάτι άλλο όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ακόμα και αν έχουμε μια πλειοψηφία πολιτών που υπερψηφίζουν μια συγκεκριμένη πρόταση, πώς μπορεί αυτή την πλειοψηφία να την επιβάλλει σε δομικές μειονότητες μειοψηφίε μάλλον. Ας πούμε ότι οι Έλληνε θα είναι πάντοτε διαρθωτικά ε, μειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού είναι πιο λίγοι. Δεν είναι, δεν είναι τόσο καλή ιδέα το πανευρωπαϊκό δημοψήφισμα όπως πιστεύουν κάτι. Δεν νομίζω θα λύσει τίποτα. Πρέπει να επανεξεταστεί η ομοφωνία κατά τη γνώμη μου. Γιατί έτσι οποιαδήποτε χώρα μπορεί να λάβει την απόφαση που θέλει και δεν ε, επιβάλλει την απόφαση σε άλλες χώρες. Λυπούμε που είμαι τόσο ομός, ε, αλλά έπρεπε να είμαι σύντομος. Ε, σας ευχαριστώ, αλλά έχουμε ωράρια που πρέπει να τα σεβαστούμε. Τρία δευτερόλεπτα για ένα τελικό μήνυμα, κυρία Steve Pierce. Κοιτάξτε, υπάρχουν ε, μόνιμα opting out για την νομισματική ένωση, ακριβώς όπως ε, και στις εσωτερικές υποθέσεις και την ισχυμένη συνεργασία. Υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία που έχουν μόνιμο opting out και κανείς δεν τις αμφισβητεί. Ε, τώρα, κατά πόσον θα είναι δυνατόν να εξαιρεθεί κανείς από το ευρώ, ε, νομίζω νομικά είναι αδύνατον. Αν τελικά συμβεί στην πρακτική, ε, θα πρέπει να υπάρξει μια αναδρομική τροποποίηση της συνθήκης, γιατί αλλιώς θα υπάρξει νομικό και οικονομικό χάος. Εν πάση αν δώσουμε την δυνατότητα θα πρέπει νομικά κάτι τέτοιο να συμβεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους εμπειρογνώμονες, λέει ο Πρόεδρος, για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα θα συνεχίσουμε μετά την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Τίντεμανς. Στις 3 θα ξεκινήσουμε. Τα λέμε αργότερα. Γεια.